Good afternoon, everybody. Thank you. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε που ήρθατε στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Καλησπέρα σε όλους. Στα γαλλικά λέει ο κύριος Σταγιάννη, ο πρόεδρος και καλησπέρα και στους ε, Ισπανόφωνους. Και τώρα θα σας τα πω στα Ιταλικά αγαπητέ κύριε πρόεδρε Ζων Κλοντ, κύριε αγαπητέ επίτροπε Τίμπορ. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί από Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία και Λετωνία. αγαπητοί Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων. Αγαπητέ Διευθυντή Ορχήστρας Μισελ Ζαρ, αγαπητέ Διευθυντή Ορχήστρας Μπάρεμπον, κυρίες και κύριοι, με τιμή μου κυρίσω την έναρξη αυτής της διάσκεψης για την πολιτιστική ευρωπαϊκή κληρονομιά που οργανώνεται στα πλαίσια της χρονιάς της πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη του 2018. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την οποία το Κοινοβούλιο και η ε, Επιτροπή Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων ε, έχει στρατευτεί και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ήρθατε σήμερα εδώ και πρώτα-πρώτα τους μουσικούς της ε, ορχήστρας των νέων της Ευρώπης οι οποίοι ε, με τόση μαεστρία μας ε, έπαιξαν ε, κομμάτια του Χάουαρτ, του Βέρντι και του Μπετόβεν. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες της ορχήστρας Europa Encanto και ιδίω αυτά τα 40 παιδιά 6 με 12 ετών οι οποίοι τραγούδησαν κάποιες άριες από την ΑΕΝΤΑ. Καλώς ορίσατε παιδιά. περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η ώρα να σας ακούσουμε. Εδώ στο Κοινοβούλιο, στον οίκο των πολιτών, είμαστε πεπισμένοι ότι η δημιουργικότητα είναι η ψυχή της ευρωπαϊκής μας ουσίας και σήμερα έχουμε προσκαλέσει ε, όλους αυτούς τους σπουδαίους ε, Ευρωπαίους και είμαστε υπερήφανοι καλώς ορίζουμε τον Ζων Μισελ Ζάρτ, συνθέτη, μουσικό και παραγωγό, τον διευθύντη οργή τον Ντενιέλ Μπάρενμποιν, που είναι πιανίστα. αλλά και διευθυντής σα, τον Έτσιο Μπόσο, ε, επίσης συνθέτης τον Τιερή Μάρξ, ο οποίος είναι σεφ Μάγειρα και επίσης ε, την ε, Ματίν Τελεκοτέ που είναι φωτογράφος και σχεδιάστρια, τον Ράντο Μιχαλιάνου που είναι σκηνοθέτης και έχει τιμηθεί ε, αλλά έχει συμμετάσχει και στην Επιτροπή Απονομής του βραβείου Λουξ που ξεκίνησε το 2007. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να καλέσουμε του συμπολίτε μα ώστε να ανακαλύψουν εκ νέου τη σημασία τη Ευρωπαϊκή πολιτιστικής κληρονομιάς της ταυτότητάς μας. Έχουμε πάνω από 3.000 χρόνια ιστορίας. Εκεί ανάγονται οι ρίζες μας και έτσι και έχει σφυριλατηθεί η κοινή μας ταυτότητα. Μπορεί το ξεχάσουμε αυτό. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλο αυτό τον πλούτο και θα πρέπει επίσης να ανατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Καταφέραμε μαζί να χτίσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση αυτών των κοινών αξιών και επίκεντρο είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ατόμου. Και αυτό το οφείλουμε πρώτα-πρώτα σε αυτή μας την ιστορία. Και έτσι γεννήθηκε η αυτοδιτά μας ε, στη, στα νησιά, στους, στους, ε, στις ακτές της Μεσογείου, στα ποτάμια, πρόκειτο για κάτι το οποίο αφορούσε τα αμφιθέατρα, ε, τα έργα της φιλοσοφίας, της σάτυρας στο θέατρο, κομικό, στην τραγωδία και ε, αυτά ξεκίνησαν από την Ελλάδα, την Ρώμη, στον Μεσαίωνα και έχουμε τα πρώτα πανεπιστήμια. Επίσης, είχαμε πάντοτε αυτά στους ελεύθερους ε, λιμένες ανοιχτούς ε, στο εμπόριο και ανοιχτούς προς την ε, ανακάλυψη νέων πατρίδων. Οφείλουμε επίση αυτό στην αναγέννηση, στον διαφωτισμό, τον ρομαντισμό, τη μοντέρνα σύγχρονη σκέψη, στο Δάντι, το Σάξπιρ, από τον Καραβάντζο μέχρι τον Ρέμπραν, τον Μολιέρο, Γκέτε, τον Καμίου Πυραντέλο, τον Βαγκόκ, τον Πικάσο και χάρη σε αυτή την ε, μοναδική διαδρομή ε, έχουμε την μισή κλωνία της UNESCO στην Ευρώπη. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και θα πρέπει να φοβόμαστε να αντιπαρατεθούμε σε άλλους ε, πολιτισμούς. Όσο πιο το ξέρουμε, τόσο πιο ισχυροί είμαστε και τόσο περισσότερο μπορούμε να συνομιλήσουμε με τους άλλους πολιτισμούς. Γιατί αυτός ο οποίος δεν έχει ταυτότητα, αυτός φοβάται τους ε, άλλους. Και χάρη σε αυτή την ιστορία η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία της ε, βιομηχανίας πολιτισμού, για τις δημιουργικές τέχνες ε, και εκεί έχουμε την ομορφιά, το design και πρόκειται για τους πιο δυναμικούς κλάδους που έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για τους νέους και για μία θέση απασχόλησης έχουμε 27 θέσεις απασχόλησης έμεσα. Και αυτό ενδεικτικά μόνο. Σχεδόν 8 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται στην ε, πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Η σημερινή μας συζήτηση αφιερώνεται σε όλες αυτές τις ε, προκλήσεις ε, της ψηφιακής εποχής, γιατί χωρίς ε, αποφασιστικότητα, τόσο ώστε να προστατεύσουμε την δημιουργικότητά μας, ε, τότε πρόκειται να πληγεί όλη η οικονομία της ε, Υπήρου. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε όσους νέους θέλουν να γίνουν συγγραφείς, σκηνοθέτες, μουσικοί, σχεδιαστές, μάγειρες και ο κόσμος μας κυριαρχείται από τους γέντες τεχνολογίας. Οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση πολιτικής προσφοράς για να μην υπάρχει ομοιομορφία. Οπότε θα πρέπει να βρίσκεται το Κοινοβουλίο στην πρώτη γραμμή για αυτή τη μάχη. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι, για όλα όσα κάνατε όσον αφορά την τροποποίηση τη οδηγία για τι ε, ε, οπτικοακουστικέ υπηρεσίε και τα μίντια. Και εδώ πρέπει να καλύψουμε και αυτέ τι ε, πλατφόρμες του Video On Demand. Επίσης έχουμε το βραβείο Lux και όλα αυτά βοηθούν στην πολυμορφία ε, της πολιτικής προσφοράς του κινηματογράφου. Αυτό νομίζω ότι χρήζει επενδύσεων και αφοσίωσης. Οπότε δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε η δημιουργικότητά μας να τροφοδοτεί απλώς τους γίγαντες του διαδικτύου. Πάρα συχνά έχουμε μουσική, έργα ή κείμενα δημοσιογράφων τα οποία διαδίδονται, αναδημοσιεύονται χωρίς ε, κάποιο είδους ε, αμοιβή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει εγγυήσει για την εύρυθμη λειτουργία της ψηφιακής αγοράς, να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού. Όπου πάμε σε όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι η Ευρώπη σημαίνει στυλ, σημαίνει γνώση, ε, σημαίνει ομορφιά και αυτό είναι η ισχύ μας είναι μια πρωτοπορία ε, αδιαμφισβήτητη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια κληρονομιά που δεν είναι δυνατόν να μετεγκατασταθεί έξω από την Ευρώπη. Οπότε ε, πρόκειται για μια νέα πολιτική και οικονομική αναγέννηση. Η επόμενη δεκαετία θα έχουμε διπλασιασμό των διεθνών ταξιδιωτών. Θα φτάσουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Σε μεγάλο βαθμό αυτό θα ωφέλεσε σε μια καινούργια άρχουσα τάξη ε, η οποία αναδύεται κυρίως από την Ασία, ε, οι οποίοι είναι αρκετά πλούσιοι και είναι αυτοί οι οποίοι ψάχνουν την ομορφιά, το στυλ, το design, την ε, μόδα και την κουζίνα της Ευρώπης. Οπότε βλέπουμε ότι θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τέτοιου είδου αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και για εξαγωγές. Όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για κάποιου σημαντικού κλάδου οικονομία, μεταφορέ, ε, κατασκευέ, εμπόριο, ε, μόδα, αγροδιατροφικά. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά ω πολυσυγκληνομιά είναι κλειδί για την οικονομία και για την ελκυστικότητα των πόλεων, των περιφερειών μα. Ε, πρόκειται για μια καινοτομία. Θα πρέπει να έχουμε μουσεία ψηφιακά, ψηφιοποιημένα τέλο πάντων και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε τα αρχαιολογικά μας αξιοθέατα, να προσέξουμε τον τουρισμό και όταν ολοκληρωθεί αυτή η τελετή έναρξης θα έχουμε ένα ρεπορτάζ από το Άρτε και θα έχουμε έτσι να δούμε κάποια παραδείγματα του πώς βοηθάει τα ψηφιακά στο να δώσουν νέα πνοή στην κληρονομιά μας. Έχουμε αυτό το, το, το, το όραμα, αυτό το project που λέγεται ε, η μηχανή του χρόνου της Βενετίας και εκεί μπορούμε να δούμε τη Βενετία ε, στο παρελθόν, στην ιστορία της, ε, τετραδιάστατα. Κυρίες και κύριοι, αυτή η πολιτιστική κληρονομιά ε, βοηθά και τις ρίζες μας, τις εκπροσωπεί, αλλά κυρίως εκπροσωπεί το μέλλον μας. Και αυτό είναι μια κοινή αίσθηση, μια κοινή πεποίθηση και ε, είναι κάτι πέρα από το κοινό νόμισμα, την οικονομία και την ασφάλεια, την κοινή. Είναι μια ευκαιρία. Δεν πρέπει να τη χάσουμε τόσο ώστε να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτή την, ε, την τρομερή πολιτιστική πολυμορφία η οποία βασίζεται σε αυτή την ευρωπαϊκή ε, πορεία, διαδρομή, περιπέτεια και μόνο όταν έχουμε επίγνωση όλων αυτών μπορούμε να αποφύγουμε το τέλος του ευρωπαϊκού όνειρου. Τώρα αυτό το όραμα, αυτή η διαδρομή περνά από κάποιες περίπλοκες ε, ε, στιγμές. Οπότε θα δώσω τώρα την ε, σκητάλη και τον λόγο στον πρόεδρο Γιούγκερ, ο οποίο ως Πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πάρα πολλά, ούτω ώστε να προστατευτεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αντώνιο, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτισμού, κύριε και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μου η χαρά που είμαι κοντά σας σήμερα. Άλλωστε πρέπει πάντα να το λέει κανείς αυτό. Αν και δεν είναι πάντοτε αλήθεια, σήμερα όμως είναι διότι έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για μια διάσκεψη που γνωρίζουμε ότι είναι σημαντική και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντώνιο που είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει στην ε, σημερινή εκδήλωση. Ο Ζαμονέ είχε πει μια φράση σύμφωνα με την οποία αν θα καλεί να ξαναρχίσει την ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα την άρχιζε αυτή τη φορά από τον πολιτισμό. Βέβαια, ποτέ δεν την είπε την φράση αυτή. Θα μπορούσε να την είχε πει όμω. Τόσο πολύ του ταιριάζει αυτή η φράση και τόσο πολύ δείχνει ανάγλυφα ένα ελάττωμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Είναι μεγάλη η ανάγκη να επιμείνει κανείς και να επιμένει διαρκώς κάθε μέρα σε αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή μας πολιτιστική κληρονομιά ανθρωπιά, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ μας είναι μέρος και της κληρονομιάς των ιδρυτών πατέρων της Ένωσης. Αυτή η αλληλεγγύη που χτίζεται και επινοείται καθημερινά από την αρχή. Αυτή η αλληλεγγύη που πολύ συχνά, ίσως υπερβολικά συχνά, τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί ρογμές. Και τώρα που σας μιλώ οι ρογμές συνεχίζονται και γίνεται όλο και πιο εύθραυστη. Ήδη καλούμεθα να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση του μεταναστευτικού. Συχνά λέω ότι αυτή η ρήξη της αλληλεγγύης συχνά αφήνει πληγές που επιμένουν και οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε καλά οι μεν τους δε. Όταν είχα παιδιά μικρά, παρακολουθούσα στο σχολείο τους, στο Λουξεμβούργο, το μάθημα της πατριδογνωσίας, που έχει σαν αντικείμενο τη γνώση της χώρας και των ιδιαιτεροτήτων της αυτή η ευρωπαϊκή χρονιά της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι κατά κάποιο τρόπο η πατριδογνωσία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την Ένωση μέσα σε όλη την ποικιλία της των χωρών και των λαών που είναι τόσο δεμένοι με τα εδάφη τους, με την επικράτειά τους, με τις παραδόσεις τους, αλλά που έχουν επιλέξει να συνεργαστούν, γνωρίζοντας ότι καθένας από αυτούς θα είχε πολύ περισσότερα να χάσει από το να κερδίσει εάν χωριζόταν από τους άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη είναι φτιαγμένη από όλη αυτή την ποικιλία και το σύνολο είναι πιο πλούσιο από τα μέρη του. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τους νέους. Και σε αυτούς πρέπει να αποδώσει η Ευρώπη που κατόρθωσε να δημιουργήσει την ειρήνη και να την κρατήσει σε μια ήπειρο που έχει τόσο υποφέρει από πολέμους. Και χάρη στην μεγαλοφία των γενεών που ήταν πριν από εμάς και που είχαν ευχηθεί και προσευχηθεί τότε όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος στη δεκαετία του 40 να μην ξαναγίνει ποτέ πόλεμος. Κάτι που ακόμα μέχρι τώρα εξακολουθεί να παράγει ωφέλη και ευεργετήματα. Είναι κάτι παραπάνω από μια μεγάλη αγορά, ωστόσο η Ένωση κάτι περισσότερο από την ενιαία αγορά ή τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μεν και των δε. Περισσότερο από το κοινό νόμισμα. Αρνούμε να συμπαρταχθώ με εκείνους που θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι μονάχα το χρήμα, το εμπόριο και τίποτε άλλο. Η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι κυρίως η καθημερινή συνεργασία των δυνάμεων όλων των Ευρωπαίων. Είναι αυτή η νεαρή μουσική που ακούσαμε πριν από λίγο. Είναι όλοι αυτοί που χάρη στο πρόγραμμα Erasmus Plus έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλες χώρες. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης αυτό το πρόγραμμα Erasmus Sin ή Erasmus Plus. Εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι και νεαρές Ευρωπαίες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό με άμεσο αποτέλεσμα ένα εκατομμύριο μωρά. Πρώτα-πρώτα από ζευγάρια που έγιναν ζευγάρια χάρη στα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής που επέτρεψε το Ερασμοσύν. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι και η καλύτερη απάντηση σε αυτή την ανοησία και την βλακεία των εθνικών εγωισμών, του κλεισίματος των εαυτών της κάθε χώρας. Όσο περισσότερο ταξιδεύουν οι νεαροί Ευρωπαίοι, τόσο περισσότερο θα γνωρίσουν τους άλλους, τις παραδόσεις, τα ρεφλέξ τους, το παρελθόν τους, την ιστορία τους, τις ελπίδες τους, αυτή την πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που έχει ανάγκη από την δύναμη των νέων. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό που δίνεται στο έρασμο ΣΥΝ στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. φέρνοντας το τελικό ποσό από 14,7 σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι κάτι, δεν είναι πεταμένα λεφτά, είναι κάτι που θα βοηθήσει το μέλλον της Ευρώπης. Δεν είναι λογιστικά ουδέτερος ο προϋπολογισμός. Κάθε προϋπολογισμός και ειδικά ο δικός μας είναι η μεταφορά σε αριθμούς των φιλοδοξιών μας. Και έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες για τους νέους και τις νέες που είναι το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες και για τον πολιτισμό ως έκφραση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας μέσα σε όλη της την ποικιλομορφία που συχνά οδηγεί και σε δημιουργία απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Μην δυσμονούμε ότι η πολιτιστική βιομηχανία, έκφραση που δεν μου αρέσει, ωστόσο δίνει δουλειά σε 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Γι' αυτό στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δηλαδή στους 7 επόμενους ετήσιους προϋπολογισμούς, προτείνουμε να αυξηθεί η δύναμη κρούσος, αν μπορώ να το πω έτσι, της δημιουργικής Ευρώπης, αυξάνοντας τις συνέργειες με άλλα προγράμματα, όπως για παράδειγμα το Horizon Ευρώπη, που θα στηρίξει ερευνητικές δραστηριότητες δραστηριότητες καινοτομίας στα μίδια και, στην, και στον πολιτισμό. Και το InvestU που θα στηρίξει και ιδιωτικές επενδύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργίας ή άλλο πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης που θα συμμετάσχει επίσης στην μετάβαση στο, στον ψηφιακό πλέον του πολιτισμού διότι πολιτισμός και ψηφιακή ε, εξέλιξη πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Όλη η καλλιτεχνική δημιουργοί, των οποίων η εργασία διαδίδεται online επιγραμμικά, πρέπει να αμείβονται δικαίως για το έργο τους. Γι' αυτό προτείνουμε έναν εξυγχρονισμό των ε, ευρωπαϊκών κανόνων των δικαιωμάτων του δημιουργού για να υπάρξει ισότητα δικαιωμάτων όλων των δημιουργών, διατήρηση της ελευθερίας έκφρασης και ευρωπαϊκές πλατφόρμες επιγραμμικές. Ελπίζω, αγαπητέ Αντώνιο, ότι ο συνομοθέτης του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το, και το Συμβούλιο θα συμβάλλουν στο να γίνει πραγματικότητα η προσπάθεια αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι τη στιγμή που η Ευρώπη για άλλη μια φορά γράφει το μέλλον της, οφείλουμε και θυμηθείτε την φράση του Ζαν Μονέ, πρέπει να αρχίσουμε από τον πολιτισμό. Τον ευρωπαϊκό πολιτισμό που συμβάλλει στην οικοδόμηση και στην προβολή της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. Ευρωπαϊκός πολιτισμός που αποτελεί και τον μισό παγκόσμιο πολιτισμό στην πραγματικότητα. Προωθώντας και σεβόμενοι τον πολιτισμό, σεβόμαστε τους ίδιους τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα σας υποστηρίξει σε αυτές τις προσπάθειες και για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, το Πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όλες τις πρωτοβουλίες υπέρ του πολιτισμού θα τις στηρίξουμε και υπέρ της νεολαίας. Ας περάσουμε τώρα στους προσκεκλημένου μας, ξεκινώντας από έναν διάσημο καλλιτέχνη, πολύ σημαντικό, τον κύριο Ζωμισελ Ζάχ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι Υπουργοί, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, αν και δεν ε, έχω την ε, συνήθεια να κάνω δημόσιες ομιλίες, πρέπει να σας πω ότι σήμερα είμαι, ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που έχω την δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσάς, σε αυτή την αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Ταγιάννη για την πρόσκληση να μιλήσουμε για την πολιτιστική κληρονομιά. Πολλέ φορέ, όταν μιλούμε για πολιτιστική κληρονομιά σκεφτόμαστε το παρελθόν, κτίρια ε, και έργα τέχνης στο παρελθόν. Είμαι γνωστός ε, ως πρωτοποριακός καλλιτέχνης κυρίως στην ηλεκτρονική μουσική που γνωρίζετε ότι είναι κάτι καινούριο, δυναμικό που κοιτάει προ το μέλλον. Πολλοί καλλιτέχνες ε, βρισκόμαστε παρόντε στη συνάντηση εδώ και ο λόγος που έχουμε έρθει δεν είναι μόνο για να μοιραστούμε μαζί σας ε, τις ανησυχίε των ανθρώπων του πολιτισμού, αλλά να σας μιλήσουμε για ανησυχίε οι οποίες αφορούν όλους μας. Γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές οικογένειες υπάρχει ένα παιδί, ένα ο του ή η αδερφή του μπορεί να ε, ονειρεύεται ότι θέλει να γίνει φωτογράφο, να ασχοληθεί με το σινεμά, να γίνει καλλιτέχνη. Και για να μπορεί να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα δίκαιο οικονομικό μοντέλο για τον 21ο αιώνα, για τον τρόπο με τον οποίο ε, δημιουργούμε πολιτισμό, τον διανέμουμε και ε, τον παρουσιάζουμε στους πολίτες. Με όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένου και του ίντερνετ. Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο το παρελθόν, αλλά πρέπει να ε, φροντίσουμε τον ε, πολιτισμό και στο μέλλον. Γι' αυτόν τον λόγο τα ζητήματα των ε, δικαιωμάτων, ε, των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού ε, είναι ένα ουσιαστικό θέμα. Ας σκεφτούμε τι επέτρεψε στον Βέρντι να ε, ζήσει ε, μια ζωή άνετη ενώ ο Μότσαρτ πέθανε στη φτώχεια. Ή ποια είναι η διαφορά. Ας σκεφτούμε αυτά τα πράγματα που έγιναν στο παρελθόν για να εμπνευστούμε για το τι πρέπει να συμβεί με τους ε, καλλιτέχνες μας. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και πάντοτε ακολουθούσαμε όλες τις εξελίξεις. Βεβαίως το τελευταίο αιώνα, στον 20ο αιώνα, το ίντερνετ είναι μια τεράστια επανάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις του ίντερνετ είναι ο εχθρός μας. Αντιθέτως, θα πρέπει να γίνουν εχθρος μας Αντιθέτω. θα πρεπει να γινουν εκεινες με τις οποίες συνομιλούμε. Οι δημιουργοί συμμετέχουν σε αυτήν την ε, ψηφιακή ε, πολιτιστική κληρονομιά. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να έρθουμε σε διαπραγματεύσεις με πλατφόρμες όπως το YouTube, το οποίο ε, ορίζει τον εαυτό του ως ένα αρχείο, ως μια πλατφόρμα αποθήκευσης. Και γιατί αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ε, του δίνεται, δίνεται τη δυνατότητα να μην πληρώνει τα αντίστοιχα δικαιώματα στους δημιουργούς. Είναι ένα κενό στην νομοθεσία το οποίο εξοπλίζει και χρόνια. Έχουμε αναπτύξει ε, καταπληκτικά τρομερά εργαλεία στο ίντερνετ και αυτές οι εταιρείε έχουν, ε, γίνει, έχουν γιγαντωθεί χωρίς όμως να έχουν αντιληφθεί ότι αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τα οποία πραγματικά χρειάζονται ρύθμιση σήμερα. Βεβαίως πρέπει να προασπίσουμε την ελευθερία της έκφρασης στο ίντερνετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσουμε στην ίδια παγίδα που με εκείνου που αρνούνται τον κώδικα δικής κυκλοφορίας όταν είχε πρώτα ανακαλυφθεί το αυτοκίνητο. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή οι εταιρείε του πολιτισμού, της πολιτιστικής βιομηχανίας έχουν τεράστια κέρδη, έχουν τεράστιο τζίρο ενώ οι καλλιτέχνες δεν αμείβονται στο σωστό επίπεδο. Πέρα λοιπόν από τα παραδοσιακά μέσα, τις εφημερίδες, τον, τον έντυπο, την έντυπη διανομή ή την τηλεόραση, πρέπει να μιλήσουμε για τα νέα μέσα της διανομής. Υπάρχει λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί και το οποίο πάντοτε υπήρχε, έτσι ώστε να επιτρέψει στους καλλιτέχνες να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους και μέσω των νέων μέσων. η σχετική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε και το θεωρούν οι καλλιτέχνε ολόκληρο τον κόσμο ότι θα έχει αποτελέσματα ντόμινο. Είχαμε πολλέ δυνατότητε να το αποδείξουμε αυτό. Γιατί αν δεν το πράξουμε αυτό, αν δεν το προστατεύσουμε αυτό, ο επόμενο Αλμοδοβάρ, οι επόμενοι σημαντικοί καλλιτέχνε του μέλλοντο θα χαθούν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, επιχειρήματα ε, τα, οποία δεν πείθουν και τα οποία ακούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόμα ε, και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρήματα παροχημένα. Είναι προφανές ότι τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού θα πρέπει να προστατευτούν για, ανεξαρτήτως του μέσου διανομής. Γιατί είναι δικαιώματα τα οποία προστατεύουν το έργο και όχι το μέσο με το οποίο διαδίδεται. σε καμία περίπτωση επίση δεν θα έπρεπε να υπάρχει η εικόνα, η ψευδή ότι εμεί οι δημιουργοί αντιτιθέμεθα στην ελευθερία τη έκφραση ή στι νέε τεχνολογίε. Δεν μπορεί τίποτα άλλο να είναι πιο ψέμα από αυτό. Εμεί ήμασταν πάντοτε πρωτοπόροι στι τεχνικέ, τι νέε και τι σπρώξαμε προ ε, νέε κατευθύνσει. Ε, και προσωπικά μπορώ να αποτελέσω παράδειγμα για αυτό όταν, ε, όταν πειραματίστηκα με τις τεχνολογίες της μουσικής. λένε ορισμένοι ότι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να είναι ε, ε, μια επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης. Και αυτό είναι ψέμα. Ακριβώς το αντίθετο είναι. Είναι ε, μια προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης του καλλιτέχνη. Θα πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να αγωνιστούμε για την ελευθερία της έκφρασης και στο ίντερνετ και να φροντίσουμε να μην καταδικάσουμε τις μικρές επιχειρήσεις του πολιτισμού ή τους καλλιτέχνες τους αυτόνομους ε, σε έναν αργοθανάτο. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα ουσιαστικά έχουν σχέση με την ευάλωτη στην θέση στην οποία βρίσκονται οι καλλιτέχνες. Ε, χρειάζονται τους νομοθέτες για να προασπίσουν την πατρότητα του έργου τους και τα δικαιώματά τους. Έχουν ανάγκη από εσάς λοιπόν το, τα δικαιώματα των δημιουργών είναι θεμελιώδου σημασία. Όπω μπορούσε κανεί να πει για την οικολογία πριν από 20 χρόνια, αντιληφθήκαμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρί τη φύση και ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο μα. Αντιστοίχω, πρέπει να, να αντιληφθούμε ε, τη σημασία του πολιτισμού. Θυμάμαι όταν είχε ο πρόεδρος της Google επισκεφθεί ορισμένες ε, ευρωπαϊκές ε, πρωτεύουσες τη συζήτηση για, τις, για τη φωτογραφία. Και θυμάμαι και είχα την ε, ε, εντύπωση ότι αυτό ήταν κάτι αντίστοιχο με τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι που ε, κατέκτησαν την Ήπειρο την Αμερικανική έδιναν καθρεφτάκια. Θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την πολιτιστική απεικιοκρατία για να μην καταλήξουμε στη δυστοπία που περιέγραφε ο Orwell. Τις προκλήσεις τις βλέπουμε όλοι μπροστά μας. Η Αφρική και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμα πιο ευάλωτες από εμάς, από την Ευρώπη, όσον αφορά την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η Αφρική, η Κίνα έχει καλλιτέχνες ε, και στην Αμερική το ίδιο, οι οποίοι κοιτούν να δουν τι θα συμβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχετε ευθύνη έναντι όλων αυτών, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πολιτισμός είναι μια έκφραση του σεβασμού της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση λοιπόν να τον υποβαθμίσουμε, να τον αποδυναμώσουμε. Γιατί έτσι προστατεύουμε την ταυτότητά μας, τις γλώσσες μας, την πολιτιστική μας ε, ε, κληρονομιά. Τα έργα, τα καλλιτεχνικά δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Και τέλο, υπάρχει και το ερώτημα που πρέπει να θέσει κανεί τελικά ποιο είναι εκείνο που επιβάλλει τη λογοκρισία, εκείνο που έχει την εξουσία να το πράξει. Σίγουρα όχι οι καλλιτέχνε που δημιουργούν. Οι πλατφόρμες του ίντερνετ προσπαθούν να έχουν και την, το μονοπόλιο να ορίζουν τι είναι cool, τι είναι στο πνεύμα των καιρών. Με αυτόν τον τρόπο όμως υποβαθμίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά, την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. Αυτό σίγουρα δεν είναι cool σίγουρα δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα των καιρών. Το ίντερνετ έχει ήδη 20 χρόνια στην πλάτη του. Είμαστε στα πρώτα τα βήματα, φυσικά στην προ, προϊστορία αν θέλετε. Το ίντερνετ σήμερα ίσως να, είναι, ε, το, να ήταν το Far West, αλλά τώρα πια έχει, έχει περάσει αυτός ο καιρός. Χρειάζεται λοιπόν αντίστοιχη ρύθμιση. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείε θα είναι αμερικανικές ή ασιατικές. Δεν μπορεί η ασιατικε δεν μπορει η ευρωπη να χάσει αυτή τη μάχη του περιεχομένου ε, ε, και να μην προβάλλει το DNA τη υπήρου μας μέσω αυτή. Εξάλλου το πρόβλημα με το YouTube δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις ή το YouTube είναι το πιο γνωστό από αυτές τις πλατφόρμες και φυσικά περιμένει να δει τι θα συμβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώς μπορεί να λάβει το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Ορισμένοι ίσως σας έχουν πει ότι η ρύθμιση μπορεί να σκοτώσει την ψηφιακή αγορά. Αυτό είναι ψέμα. Το να δημιουργήσουμε μια δίκαιη αμοιβή ε, δεν είναι ε, κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο εταιρείε οι οποίε έχουν κέρδη δισεκατομμυρίων. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι πώ μπορούμε να, να υπάρχει μια δίκαιη αμοιβή για αυτού που πραγματικά έχουν παράξει το περιεχόμενο. Και αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση λογοκρισία. Κλείνοντα. Το μήνυμα είναι πολύ απλό. Δυστυχώ βασιζόμαστε σε ένα παροχημένο νομοθετικό πλαίσιο και προσπαθούμε μέσω αυτού να ρυθμίσουμε το ίντερνετ. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται να μα δώσετε τα, τα, τα μέσα έτσι ώστε να καθίσουμε σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι ω Ευρωπαίοι δημιουργοί με ισότιμου όρου απαιτώντα δίκαιη αμοιβή για τη δημιουργία για τις μας και για τη διανομή τους. Και ας μην ξεχνούμε ότι το smartphone έχει την ευφυή του πλευρά ακριβώς εξαιτία ημών των δημιουργών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζουάρ. Και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ντανιέλ Μπάρενμποϊμ. Κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη και Γιούνκερ, εξοχότητες, ε, κυρίες και κύριοι, είναι Μεγάλη μου τιμή να ομιλώ ενώπιόν σας σε αυτή την εκδήλωση για το 2008 το έτος της ε, πολιτικής κληρονομιάς. Γιορτάζουμε το κοινό μας παρελθόν και ελπίζουμε ότι μαζί θα οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον. Πρόκειται για έναν εορτασμό ο οποίος έρχεται ακριβώς την πιο σωστή στιγμή μια που είναι πάρα πολύ μεγάλες ε, οι απειλές στην κοινή μας ευρωπαϊκή ταυτότητα. 75 χρόνια έχουν περάσει από το τέλος του πολέμου και έχουμε επικίνδυνους εθνικισμούς και λαϊκισμούς οι οποίοι έχουν φουσκώσει παντού στην ε, Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να παρακάμψουμε αυτές τις απειλές, θα πρέπει να ενισχύσουμε και πάλι την ιδέα μιας Ευρώπης που να είναι ειρηνική. Να, ποιο είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Μεγαλύτερη από ποτέ και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με όλα τα μέσα τα οποία μπορούμε να επικαλεστούμε. Οπότε έτσι θα πρέπει να γυρίσουμε σε κάποιον πολιτισμό ε, των γεγονότων, των πραγματικών περιστατικών. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, το οποίο έχει αφήσει πολλά περιθώρια για ψευδή αφηγήματα. Ο πιο φασαρτζής κερδίζει πόντους. Και αυτά τα οποία λέει μπορεί να είναι αλήθεια ή ψέματα. Οπότε αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και στο πεδίο της πολιτικής και του πολιτισμού. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι αυτό το οποίο έχει δώσει αρκετά στην Ευρώπη είναι ο πολιτισμός και είναι πολλές οι χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν αναπτύξει το δικό τους διαφορετικό πολιτισμό αλλά ανέκαθεν ναι, αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι η σημασία που αποδίδουμε στον ε, πολιτισμό. Η απαριθμίση είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Σοφοκλής, ε, Πλάτων, Καρτέσιος, Δάντε, Γκέτε, Μπετόβεν, Μότσαρντ, Ντεμπισί, Λονάρντο Νταβίντσι κλπ. Ποια άλλη ήπειρος θα μπορούσε να διεκδικήσει, θα μπορούσε να, να, να προτάξει τέτοιου είδους ε, πλούτο και πολιτισμό. Η άνοδος του εθνικισμού είναι ως επιτοπλίστων αποτέλεσμα του ότι ο κόσμος πολλές φορές δικαιολογημένα είναι δυσαρεστημένος από την παγκοσμιοποίηση η οποία έχει ε, ένα αποτέλεσμα ομοιογενοποίησης του πολιτισμού αυτού που είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα που είναι η υπέροχη πολυμορφία μας αλλά ο εθνικισμός δεν είναι η απάντηση σε αυτά ο πατριωτισμός είναι περηφάνεια για την ανήκει σε κάποια χώρα ο εθνικισμός πολλές φορές αποκλεί τον πατριωτισμό και αν ε, κανείς δεν έχει αξίες ε, τότε δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους δεν μπορεί να εκτιμήσει τον πολιτισμό του άλλου να τι θα πει ε, πνεύμα παγκόσμιο και διεθνιστικό να αυτό είναι ε, το, η καλή πλευρά της παγκοσμιοποίησης και αυτό πρέπει να μας ε, απασχολήσει γιατί επί πολύ καιρό έχουμε εστιαστεί μόνο στα οικονομικά ε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τον χώρο, τον χώρο του πολιτισμού, τον κοινό, ε, που τον έχουμε παρα, κάπως παραμελήσει και αυτά είχαν κατά νου Κόλ και Μιτεράν όταν κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου ε, ενώπιον ε, ενός αγήματος γαλλογερμανικού από στρατιώτες και έτσι επομένως ε, γνωρίστηκαν οι λαοί με, με ε, τον πολιτισμό με τον Μπετόβεν, τον Τόμας Μάν, τον Ντεμπισί, τον Μποντλέρ και ως μουσικός πέρασα τη ζωή μου προσπαθώντας να καταλάβω άλλους πολιτισμούς και άλλους λαούς μέσω της μουσικής, κάτι το οποίο ήταν ένα προνόμιο, αλλά αυτό θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε προς κάθε Ευρωπαίο. Θα πρέπει όλοι αυτό να το δοκιμάζουν. Και ένα από τα θετικά τη παγκοσμιοποίηση είναι ότι τώρα είναι φυσιολογικό, είναι δυνατό να φάει κανεί σε τελικό φαγητό τη Δευτέρα στην Ιαπωνία, το στο Μόναχο Ιαπωνέζικο φαγητό την Τρίτη και γερμανικό φαγητό στο Λονδίνο την Τετάρτη, ή άντε στο Παρίσι. Γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη διαδρομή και πρώτα για αυτή την πολυμορφία η οποία μας δίνει την πολυμορφια η οποια μα δινει την δυνατοτητα να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τους άλλους πολιτισμούς, τους άλλους λαούς και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε θετική επίδραση ο ένας επί του άλλου. Με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να σας εκφράσω τη θλίψη μου, τη στενοχώρια μου, γιατί η μουσική παιδεία δεν εμφανίζεται στην ύλη των σχολείων. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Η μουσική είναι από τους καλύτερους τρόπους τόσο ώστε να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος των ε, ανηλίκων αλλά και ο συστηματικό του κόσμος. Δυστυχώς στον σημερινό κόσμο κάποιος μπορεί να είναι καλλιεργημένος χωρίς να έχει καμία επαφή με τη ε, μουσική, χωρίς να παίζει κάποιο μουσικό όργανο ή χωρίς να ακούει μουσική. Μα δεν υπάρχει ε, λόγος να μην θεωρούμε ότι είναι ένα ακόμη μάθημα η μουσική, όπως είναι τα μαθηματικά, όπως είναι τα φιλολογικά, όπως είναι η γεωγραφία. Αυτό θα συζητηθεί κατά αυτή τη ε, διάσκεψη που κάνουμε και ελπίζω ότι θα δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν και έτσι θα ξαναγυρίσουμε στην αρχική ιδέα για το τι είναι εκείνη η Ευρώπη. Πάντως είναι μια πρόκληση είναι το ότι συνεχώς αλλάζει το ψηφιακό τοπίο και σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αναδείξουμε την αξία της μουσικής και της τέχνης, τους δημιουργούς των έργων ε, τέχνης. Επίσης η καταγραφή των έργων τέχνης είναι κάτι που συνδέει μέλλον με παρελθόν για μας. Και συμπαθάτε με και θα είναι προσωπικό το παράδειγμα που θα επικαλέσω. Εγώ έκανα την πρώτη μου ε, εγγραφή πριν από 64 χρόνια. Το 54. Εγώ δεν, και δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Και εκείνη η εγγραφή και καμιά δεκαριά άλλα εκατομμύρια εγγραφών τώρα είναι προσβάσιμα. Ε, αυτό είναι τρομερό. Και τη στιγμή που κάνει κάποιο μουσικός δημοσιοποίηση κάποια συγγραφή στο έργο του, τώρα είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε παγκόσμια εμβέλεια. Φοβερό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μα, ούτω ώστε να αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό, ούτω ώστε να μπορέσει να περάσει στι επόμενε ε, γενίε, να περισσωθεί. Και είναι μεγάλο ο προβληματισμό στους δημιουργούς μουσικής το ότι πάρα πολλοί τρόποι μέσω του ίντερνετ αδικούν τη μουσική δεν αδικούν την αξία της και έχουμε τώρα το δίκαιο copyright είναι κάτι το οποίο τώρα το καταστρώνει και το αναθεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε να ε, πώς μπορούμε να φροντίσουμε ακόμα ένα σύνδεσμο του παρελθόντος με το μέλλον. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κενό αξίας όσον αφορά την ε, μουσική στο ίντερνετ. Και εμείς στην ε, κοινότητα της ε, μουσικής ενατενίζουμε τις δικές σας προσπάθειες. Εσείς ως νομοθέτες για να εξασφαλίσετε το ότι η τέχνη, η μουσική, ε, από πάση απόψεις και εμπορική θα προστατεύονται τη σημερινή ημέρα, την ημέρα της ψηφιακής εποχής. Και γιατί θα πρέπει αυτό να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάθαρους λόγους και πάρα πολλούς. Αλλά ο βασικός λόγος είναι η ευθύνη μας να περισσώσουμε για το μέλλον τον πολιτισμό που έχουμε και που σήμερα τιμούμε. Ιδάλλως καταστρέφεται αυτός ο σύνδεσμος, αυτός ο κρίκος. Και πριν λίγο ακούσαμε την ε, ορχήστρα των ε, νέων και να, η καλύτερη απόδειξη για αυτό το οποίο επιβαρέται να γίνει το διαδίκτυο μας δίνει πάρα πολλά πλέον σε όλους, νέους μουσικούς και μεγαλύτερους στην ηλικία όπως ο υποφαινομένος. Και άκουσα τόσες ιστορικές ηχογραφήσεις και πάρα πολύ πρόσφατα άκουσα μια ηχογράφηση του Falstaff του Βέρντι από το Ζάλτσμπουργκ του 36 και διευθυντής ήταν ο Αρτούρο Ήταν μία από τις πιο υπέροχες παραστάσεις που έχω παρακολουθήσει. Και οι νέοι μουσικοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, το YouTube και άλλες πλατφόρμες και μπορούν από εκεί να αναδειχθούν. Πρέπει να έχουν όμως δίκαιη αμοιβή. Ιδάλλως, δεν έχουν κάποιο εισόδημα το οποίο είναι τόσο σημαντικό για οποιονδήποτε καλλιτέχνη. Και θα πρέπει επομένω να στηρίξουμε την επόμενη γενιά καλλιτεχνών, γιατί αυτοί θα δώσουν μορφή στο κοινό μέλλον, τον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό μας. Ειρήνη, ενωμένη Ευρώπη με κοινό πολιτισμό. Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια ελκυστική ιδέα. Είναι μονόδρομος για το μέλλον και εκείνοι που πέρασαν τη φρίκη των δύο παγκοσμίων πολέμων ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σκεφτεί την πολιτιστική ένωση, την ιστορία του κάθε λαού να αναδείξει, αλλά και την κοινή ιστορία και έτσι να προχωρήσουμε για το κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας προς εμένα αλλά και προς τη μουσική μας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάρενμποεμ. Ακολουθεί η Πέτρα Κάμε Εβέρτ, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει το λόγο κυρία ε, Κάμε Εβέρτ. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κύριε πρόεδροι, αξιότιμη κύριε επίτροπε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και για μένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μπορώ σήμερα να σας απευθύνω χαιρετισμό υπό το αξίωμά μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευκαιρία το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού. Λίγες άλλες πρωτοβουλίες του πρόσφατου παρελθόντος έχουν τέτοια αξία που να μπορούν να φέρουν το σύμβολο ευρωπαϊκός. Από τη μια μεριά ε, όμως αξίζει στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι ξεκίνησε και η πορεία του αρκετά δύσκολα, όπως γίνεται συχνά στην Ευρώπη, και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της χώρας μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια και με την υποστήριξη πολλών φορέων της ε, κοινωνίας των πολιτών, για να καταλήξει να γίνει πραγματικότητα. Και έκφραση αυτής της προσπάθειας είναι η σημερινή πρωτοβουλία με την παρουσία ε, σημαντικών προσωπικότητων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου του πολιτισμού. Από την άλλη μεριά αξίζει να φέρει το ευρωπαϊκό έτος τον χαρακτηρισμό ευρωπαϊκό και λόγω των φιλοδοξιών που επιδιώκει διότι μιλεί πέρα από τα γλωσσικά και τα εθνικά όρια για έναν πολιτισμό που είναι εκείνος ο δεσμός που ενώνει όλους τους λαούς της Ευρώπης. Γιατί μπορεί κανείς να μιλήσει για μια πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό ισχύει και από άποψη χρόνου, διότι σημαίνει μια, ένα κεντρικό σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Εκεί δηλαδή όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον. Η τέχνη και ο πολιτισμός που ε, δημιουργούνται σήμερα είναι πολιτιστική κληρονομιά της αύριον. Διαμορφώνονται όμως σήμερα. Έτσι λοιπόν η σημερινή συνάντηση είναι αυτή που προσφέρει την ευκαιρία όλοι μαζί ως καλλιτεχνική δημιουργή, ως πολιτικοί και ως πολίτες να στοχαστούμε γύρω από τις διάφορες πτυχές και λειτουργίες της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός ρόλου του πολιτισμού μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική διότι αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδέστηση η ελπίδα ότι δήθεν μόνο η οικονομική πτυχή θα αρκούσε για να αναπτύξει τέτοιες συνθετικές δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που να επιτρέψουν ταύτιση των πολιτών με την Ευρώπη στο διηνεκές. Για να μην μιλήσω καν για τη συναισθηματική ταύτιση των ανθρώπων με την Ευρώπη. Όμως για την ανάπτυξη του πολιτισμού δεν αρκεί κανείς να πιστεύει αφελώς σε, στη δύναμη του πολιτισμού θεωρώντας ότι θα είναι η πανάκια για όλα τα προβλήματα της Ευρώπης και του κόσμου. Πρέπει κανείς να έχει διαρκώς υπόψη την αμφισημία του πολιτισμού διότι μπορεί ο πολιτισμός να λειτουργήσει και συνδετικά αλλά και διαλυτικά. Συχνά όταν ο πολιτισμός χρησιμοποιείται ως όχημα εθνικισμών, αποκλεισμών ή δυσφήμιση του άλλου εντό εισαγωγικών, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα υπερβολικά συχνά. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Δανίλ Μπάρνμποιμ που μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα σε εθνικισμό και πατριωτισμό. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει σήμερα και το έτος του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι η αυτοκριτική αντιμετώπιση του κοινού μας, του κοινού ευρωπαϊκού πολιτιστικού πλούτου. Ελπίζω ότι αυτό το έτος ευρωπαϊκού πολιτισμού θα οδηγήσει και σε μια νέα όθηση μιας νέας ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής στην Ευρώπη και στις χώρες μέλη. Και πάλι ευχαριστώ εδώ ιδιαίτερα τον Ντάνιελ Μπάρενμποιμ που τόνισε και πάλι πόσο σημαντικό είναι να επενδύσει κανείς στην πολιτιστική παιδεία η επίσκεψη σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε ένα μουσείο δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να θεωρείται σαν αποχή από το μάθημα μόνο και μόνο επειδή δήθεν ο δάσκαλος δεν έχει καμιά καλύτερη ιδέα. Όχι, αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο μέρος των εκπαιδευτικών συστημάτων μας. Και πρέπει όλο και περισσότερο να δούμε πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και ιδίως να την εγγυηθούμε την πρόσβαση αυτή σε όλους. Συχνά θεωρούν πολλοί ότι ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της ε, ε, κοινωνίας όταν είναι ομοιογενής. Εγώ πιστεύω όμως ότι ιδίως στον πολιτισμό μπορεί να προκύψει μέσα από την ποικιλία, από την πολυφωνία ένα είδος ενότητας, διότι η πολυφωνία δεν είναι μονάχα, ως γνωστό, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολυφωνία είναι και ένα κεντρικό στοιχείο αυτού που θεωρούν στον κόσμο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Εμείς, ωστόσο, οι πολιτικοί πρέπει να κριθούμε από το πόσο σοβαρά εννοούμε αυτήν την πολυφωνία. και εν του ιστορικού, πολιτισμικού και γλωσσικού όπως το βλέπουμε σήμερα. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι η πολυφωνία μέσα σε μια εποχή αυξανόμενων αυταρχικών και λαϊκιστικών τάσεων δεν είναι εξασφαλισμένη. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε παρέτηση. Αντίθετα θα πρέπει να μας κινήσει, να μας οθήσει σε αποφασιστική δράση. Ας δουλέψουμε από κοινού και σκληρά ώστε ο πολιτισμός και κυρίως ο πολιτισμός βασισμένος στις θεμελιώδεις αξίες του σεβασμού και της ανεκτικότητας απέναντι στον άλλο να αποτελέσει τη βάση της πολιτικής δράσης για το καλό της Ευρώπης, για το καλό των πολιτών και των δύο φίλων, αλλά και πέρα από τα όρια της Ευρώπης για όλο τον κόσμο. Και σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ, Πέτρα. Τώρα θα δώσω το λόγο στο Ρούμεν Τιμητρόφ, αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Έχετε το λόγο. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε Ταγιάννη, κύριε Πρόεδρε Γιούνκερ, κυρία Κάμερεβερτ, κύριε Ναύρατσιτς, ξέρετε, Υπουργοί των Κρατών Μελών, Λοιποί εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, αγαπητοί φίλοι, κυρίε και κύριοι. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκομαι εδώ στην έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτου Πολιτιστική Κληρονομιά σε αυτή την διάσκεψη όπου συζητούμε πώ μπορούμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το μέλλον. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ταγιάννη για την πρόσκληση, καθώ επίση να ευχαριστήσω και όλου εσά που ήρθατε στην διάσκεψη αυτή, με την παρουσία σας αποδεικνύεται ε, την σημασία αυτού του εγχειρήματο. που αναφέρεται σε μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, την πολιτιστική κληρονομιά, που μας επιτρέπει να ε, οραματιζόμαστε και το μέλλον. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα κοινό αγαθό που γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την Ευρώπη για λόγους ε, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς προφανώς. Όταν κανείς ε, μετέχει ε, αυτού της κληρονομιάς, όταν συνεισφέρει στην πολιτιστική κληρονομιά, διευρύνει τους οριζοντές του και μπορεί να κοιτάξει τη ζωή, τον κόσμο με τρόπο διαφορετικό πολιτιστική κληρονομιά στέλνει και σταθερά μηνύματα. Μας επιτρέπει να δίνουμε νόημα στην ε, ζωή μας και στη, στην εμπειρία μας. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να την αποδώσουμε στις επόμενες γενιές. Βρισκόμαστε στο πλαίσιο μιας, ε, στο, στο να απόϊχο μάλλον μιας ε, μεγάλης οικονομικής κρίσης ε, η οποία μας έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια οικονομική ένωση, οφείλει να είναι μια ένωση αξιών και θεμελιδιών δικαιωμάτων. Σήμερα λοιπόν, για να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ευρωπαϊκό εγχείρημα, χρειάζεται να ανανεώσουμε τις, ε, τους δεσμούς μεταξύ μας και μεταξύ των κοινωνιών μας. Και ο πολιτισμός είναι ε, ένας τρόπος για να συμβεί αυτό. Είναι ένας από τους ε, τρόπους με τους οποίους ορίζει κανείς την ταυτότητά του, την ε, συμμετοχή του σε μία από τις κοινότητες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια κοινή αγορά. Αντιλαμβανόμενο όλα αυτά, κατέληξε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμπεράσματα ήδη από το 2014 για τον πολιτισμό και από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό σαυλάκι και επιλέγει το 2019 ως, ε, 2018 συγγνώμη, ως έτος πολιτισ, πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον Δεκέμβριο του 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά στο να οικοδομεί κοινότητες ε, που έχουν σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, καθώς επίσης και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να παίξει το ρόλο του τον οικονομικό και τον, και τον κοινωνικό ο πολιτισμός. Αξιοποιώντας και φέροντας στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό αναγνωρίστηκε και πάλι στα αντίστοιχα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μάιο. Ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα τη συζητήσεως στο Συμβούλιο ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων και όλων των εμπλεκομένων στο γιατί χρειάζεται να αξιοποιούμε την πολιτιστική κληρονομιά και γιατί αυτό είναι ένας τρόπος να ενθαρρύνει κανείς την καινοτομία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας ε, και γιατί μπορεί να συνεισφέρει επίσης και στην εδαφική συνοχή ε, την περιφερειακή συνοχή, μπορεί να βοηθήσει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους, προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για όλους αυτούς τους λόγους, το Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη-μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προώθησης του πολιτισμού και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, με τα οποία συγκεκριμένα μέτρα να αξιοποιούν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά ως ένα στρατηγική σημασία πόρο. Ε, συμφωνήθηκε επίση ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλα τα η επιτροπή μαζί για να έχουμε μια κοινή εικόνα, μια κοινή στρατηγική, ένα κοινό όραμα για το πώς αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που θέλουμε να δούμε να βγαίνουν από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σημερινή διάσκεψη έρχεται και σε μια στιγμή σημαντική στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε έχουμε αρχίσει να συζητούμε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και θα πρέπει να ε, ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση του προπολογισμού που προβλέπει για το πρόγραμμα Creative Europe για την ε, ε, υποβοήθηση της δημιουργίας στην Ευρώπη και το οποίο ανέρχεται πλέον σε ένα ύψος 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. για να, είναι για να είμαστε πιστικοί προς τους πολίτες μας θα πρέπει να συνεχίσουμε και να υποστηρίζουμε όλες τις δράσεις τις οποίες προανέφερα αλλά να αναλάβουμε και νέες. Ε, να αξιοποιήσουμε και άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς τα επόμενα χρόνια. Ε, για μένα αυτό είναι και η πιο δύσκολη πρόκληση να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις πιθανές ευκαιρίες και δυνατότητες για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον, τον πολιτισμό στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο των χωρών μας. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποια είναι η δυναμική που μας δίνει η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά επίσης και ποιες είναι όλες οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει κανείς για να, για να υποστηρίξει την πολιτιστική δημιουργία. με όλες αυτές τις αποφάσεις των συμβουλίων που σας παριέγραψα, τις πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αντίστοιχες με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το νέο, και το νέο ε, πρόγραμμα για τον πολιτισμό που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύμπνοια για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς χρειάζεται ε, συνεργασία ε, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν ε, οι δημιουργοί, οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και όλοι οι πολίτες. Μόνο με τέτοια συμμετοχική προσέγγιση, με μεγάλη συμμετοχή, θα μπορέσουμε να πούμε με ασφάλεια ότι και οι γενιές που θα μας διαδεχτούν θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να απολαύσουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τώρα βρεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα παιδείας, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είμαι μεγάλη μου χαρά να παρίσταμε σήμερα εδώ ενώπιον σα και θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο Ταγιάννη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι διοργάνωσαν αυτή την ε, εκδήλωση ούτω ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της υπόθεση τη Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ο πολιτισμός δηλαδή και η πολιτική κληρονομιά Όπω προαναφέρθηκε και ισχύει το ευρωπαϊκό όραμα ανέκαθεν αφορούσε τον πολιτισμό διότι πάνω απ' όλα ο πολιτισμό μα ενώνει και ε, η πολυμορφία του πολιτισμού μας ε, μας επιτρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε ένα τον άλλο, να αποδεχθούμε τις διαφορές μας και να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα κοινά μας στοιχεία. Οπότε γι' αυτό και υπάρχει η κριτική για το πώς καλύτερα θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη. Να υπάρχει ανθεκτικότητα, ε, στην κοινότητα και στις κοινότητες και για άλλη μια φορά τώρα να γνωρίζεται η αξία του πολιτισμού. Ε, επανήλθε ο πολιτισμός στην κορυφή του θεματολογίου μας. Ας εξασφαλίσουμε, ας σιγουρεύσουμε ότι θα παραμείνει και στην κορυφή. Η κληρονομιά μας αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και ήδη έχει βοηθήσει ούτω ώστε να δοθεί αυτή η όθηση που πρέπει τώρα να αξιοποιήσουμε και θα πρέπει να τάξουμε και τις φιλοδοξούς στόχους και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ό,τι χρειάζεται για να τους πετύχουμε. Επίσης τώρα έχουμε ε, αυτά τα οποία χρειάζονται, ούτω ώστε να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντό μα και υψηλή ποιότητα ο πολιτισμό. Ε, τώρα έχουμε περάσει το μισό αυτό έτος του πολιτισμού ε, και Είχαμε 2.500 εκδηλώσει σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Έτσι μπορέσαμε να επισημάνουμε την κληρονομιά μας, κάτι που θέλαμε να, να μπολιάσει την καθημερινή ζωή όλων στην κοινωνία μας και ε, συμμετέσχουν σε όλα αυτά ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι και οπότε μπορούσαμε να δούμε πώς θα έχουμε βιώσιμη πολιτισμό, τουρισμό, πώς θα ε, μπει στην καθημερινή ζωή των πόλεων ο πολιτισμό και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να γίνουν ε, γίνονται διότι όλοι βοηθούν τόσο ώστε η χρονιά αυτή του πολιτισμού να γίνει μια πραγματικότητα όλοι εμπλεκόμενοι, η κοινότητα των πολιτών, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι διοργανωτές και επίσης έχουμε και τις νέες χώρες μας και τους διεθνούς μας, ε, διεθνείς μας εταίρους να ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι οι ευρωβουλευτές είναι πρέσβης ε, για τον πολιτισμό ε, και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Κάμερα φέρετε την πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου. Να ευχαριστήσω επίσης ε, του, την κυρία Κώστα, τον κύριο Διακόνου και την κυρία Σόντροβα, σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής της πολιτικής αυτής επιτροπής να ευχαριστήσω και την Περιφερειακή Επιτροπή μάλλον των περιφερειών στην Ευρώπη ε, γιατί ε, θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η χρονιά ούτως ώστε ο πολιτισμός να είναι στην κορυφή του θεματολογίου μας και αυτό είναι το κλειδί του να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει ο πολιτισμός και επίσης έτσι θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα την ταυτότητα αυτή που δεν απειλεί αλλά εμπλουτίζει την περιφερειακή την τοπική και εθνικοί ταυτότητες. Οπότε γι' αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θεματολόγιο που καταρτήσαμε πριν από ένα μήνα και έχουμε τρεις πτυχές, κοινωνική, οικονομική και εξωτερική και έχουμε ε, τώρα ε, την εντολή προς να συνεχίσουμε γιατί έτσι ε, ενθαρρύνεται η συνεργασία για το μέλλον. Και ένα κεντρικό στοιχείο του νέου θεματολογίου είναι το σχέδιο δράσης για την πολιτική κληρονομιά. Αυτό θα σας παρουσιάσω περί τα τέλη ενεστώτος έτους. Με αυτό το πρόγραμμα δράσης βλέπουμε ποια είναι η κληρονομιά μας, το βλέπουμε πολλά, είναι χαρτί πορεία πορείας για το τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε, για να προωθήσουμε την κληρονομιά μας και έχει να κάνει με αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλη τη χρονιά σύμφωνα με το ότι θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα, προστασία, στράτευση και καινοτομία να καλύψουμε την αθλητισμό των νέων, την προσβασιμότητα στην κληρονομιά και σε δραστηριότητες ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο έργων τέχνης. Και επίσης θα πρέπει όλα αυτά να είναι προτεραιότητες και το πρόγραμμα δράσης θέλουμε να λάβει υπόψη τη γνώμη των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και άλλων, και άλλων εταίρων. Ε, αυτές οι απόψεις ε, που συζητήθηκαν στο Λονδίνο και την περασμένη εβδομάδα στην συνάντηση κορυφής. Αυτή η έκκληση αφορά την Γερμανική Επιτροπή για τα Πολιτιστικά που συντονίζει τις εκδηλώσεις στη Γερμανία και αυτή η κλονιά για φέτο μα δίνει μια ευκαιρία ούτως ώστε να ασκήσουμε επιρροή στην προβληματική για το μέλλον τη Ευρώπη. Τόσε απειλέ, τόσε προκλήσει για τι βασικέ μα αξίε. Αυτή η προβληματική δεν μπορεί να δοθεί γύρω από του άξονε τη πολιτική και τη ασφάλειας. Ο πολιτισμό θα πρέπει να είναι στην καρδιά αυτή τη προσπάθεια. Αγαπητοί κύριοι ευρωβουλευτέ, ήρθε η στιγμή να επιδείξουμε φιλοδοξία. Φιλοδοξία ε, θα πει και πρικοδότηση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο μετά το 2020 πρόκειται να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα προβληθεί και που θα υποστηρίζει ε, τον πολιτισμό. 1,85 δις θα διατεθούν για το Creative Europe δηλαδή σε εκατομμύρια παρά μόνο από όσα τώρα. Και έτσι θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και άλλα προγράμματα έρευνας, κοινωνική συνοχής, περιφερειακή ανάπτυξη. Οπότε, υπολογίζουμε στη δική σα βοήθεια. Να μας βοηθήσετε ο επόμενος προπολογισμό να στηρίξει τον πολιτισμό και την πολιτική κληρονομιά αποτελεσματικά με το Creative Europe και με κάθε άλλο τρόπο και η πολιτική είναι ξεχωριστές αυτές οι στιγμές επέστρεψε εκεί που ανήκει ο πολιτισμός ακριβώς στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ευρώπης τώρα υπάρχει ευρεία συνένεση ότι για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ανάπτυξη, συνοχή, ε, σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο, ε, το κλειδί είναι ο πολιτισμός και επίση κυρίως είναι η δύναμη που καθορίζει το ποιοι είμαστε και το τι μέλλον χτίζουμε. Οι κοινωνίε μα έχουν αντιμετωπίσουν πάρα πολλέ προκλήσει. Από μέσα και από έξω και έχουμε ε, τα κενά που μεγαλώνουν τι αποστάσει. Ε, οπότε ο πολιτισμό είναι το κλειδί για να ξανασυνδεθούμε. Οπότε α, έτσι θα καταλάβουμε τι έχουμε κοινό, έτσι θα καταλάβουμε τι πάει να πει να είναι κανεί άνθρωπο. Θα καταλάβουμε τι αξίε, θα καταλάβουμε τα συναισθήματα που είναι το θεμέλιο μας. Οπότε θα πρέπει με τον πολιτισμό να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία συμβίωση Ε, άρα θα πρέπει όλα αυτά να είναι στο επίκεντρο της δράσης μας εδώ ε, στην Ευρώπη. Στην καθημερινή μας ζωή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τίμπορ, για την ομιλία σου και για την συνεργασία φέτος. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα η Μόνικα Γκρούτερ, υπουργό ε, από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, είναι επίτροπος για τα τον πολιτισμό και τα μέσα μαγνητιστικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ αξιότιμε πρόεδρε Ταγιάννη, κυρίες και κύριοι. Ε, η Ενωμένη Ευρώπη ε, γράφεται ακριβώς ε, στο ασπρόμαυρο χαρτί των ευρωπαϊκών συνθήκων. Και είναι που πρεσβεύουν τα θεσμικά όργανα εδώ στην, Ευρω... στην Βρυξέλλες. Έτσι λοιπόν, μέσα στις συνθήκες του Μάστρικ και στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει το άσπρο. Έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα. Έχουμε ένα οικοδόμημα το οποίο μας μεταφέρει υλικά και άλλα αγαθά. Τις ε, ιστορίες, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Όλα αυτά χρωματίζουν την Ευρώπη και μας ενώνουν. Η μουσική, ας πούμε. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα των Νέων που είναι ακριβώς ε, για μας ε, αυτό που μας κάνει να ακούμε τον ήχο της Ευρώπης. Εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε στοιχεία που μας ενώνουν και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό τώρα παρά άλλες εποχές. Τώρα που οι εθνικιστικές ε, δυνάμεις μας θέτουν ενώπιον αυτών των ε, μεγάλων προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όπως η πολιτική ασύλου και να τα διαμορφώσουμε εκ νέου. Φέτος το 2018 θέτουμε τους πυλώνες ε, της Ευρώπης. Όχι μόνο δίνοντας μια ε, μαρτυρία για τις προηγούμενες εποχές, αλλά μιλώντας και για το μέλλον. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούμε και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους ε, σε πολλά φόρα και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν αλλά και γενικά για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από κάθε μεριά ώστε να υποστηρίξουμε αυτούς τους σκοπούς. Φέτος η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά είναι το αποκορύφωμα όλων αυτών των εκδηλώσεων. Έχουμε πάνω από 100 θεσμούς από όλη την Ευρώπη που την περασμένη εβδομάδα ήρθαν στο Βερολίνο και είχαμε πάνω από 400 εκπροσώπους για να μας τονίσουν, όπως ο Ζαν Μισελ ε, Μεζάν, πόσο σημαντικά είναι αγαθά όπως η πνευματική ιδιοκτησία, έτσι ώστε να μην ζουν εφήμερα τα έργα των δημιουργών. Αντιμετωπίσαμε, ας πούμε, το θέμα των αξιών, των αρετών, πώς όλα αυτά τα έχουμε διαμορφώσει μέσα από σκληρή δουλειά και πώς πρέπει να τα σώσουμε στην ψηφιακή εποχή. Στο Βερολίνο, στη Σύνοδο Κορυφή. επίσης διαπιστώσαμε πόσο σημαντικό είναι το κράτος και η κοινωνία των πολιτών. Είναι το Ευρώπα Νόστρα. Είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς να προωθήσει την κατανόηση μεταξύ μας ε, και να γιορτάσει τις αξίες ε, και τις αρετές. Έχουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματα τα οποία είναι κάτι παραπάνω από ότι μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ε, και από την εφαρμογή των κοινών συμφερόντων. Σε πάρα πολλούς τόπους δυστυχώς δεν ακούγεται αυτό και έχουμε ξανά τον εθνικισμό η υπερηφάνεια για την πολυμορφία και για την συνύπαρξη με άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες δεν ακούγεται τόσο. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι ακριβώς σε αυτούς τους καιρούς που έχουμε τόσους μεγάλους διχασμούς στην Ευρώπη ε, Είμαι πεπισμένη ότι η κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης θα μας βοηθήσει να τη διαμορφώσουμε ακόμα περαιτέρω. Έχουμε για παράδειγμα ε, συγκεκριμένα ε, σημάδια αυτού του πολιτισμού, ας πούμε την αρχιτεκτονική και άλλους τομείς που έχει υπάρξει ανταλλαγή. Ε, μετά από όλα αυτά, από όλα όσα έχουμε βιώσει στην Ευρώπη και τους πολέμους, έχουμε πια ένα πολιτιστικό κέρδος το οποίο είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτές τις εθνικιστικές βαρβαρότητες. Όμως οι οραματιστές της συνθήκης της Ρώμης, Ρώμης μας έδωσαν τη δυνατότητα πλέον εδώ να είμαστε σήμερα ως Ευρωπαίοι και να τα έχουμε καταφέρει να έχουμε βάλει πάνω από τους διχασμούς μας ε, την ενότητά μας. Έτσι λοιπόν έχουμε διαφορετικές ε, κουλτούρες ε, και θρησκείες, έχουμε μια παγκόσμια θεώρηση του κόσμου. Έχουμε μια ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία, μέσω της κατανόησης και αυτό κάνει την Ευρώπη όπως και η ειρήνη που είναι ε, στην καρδιά της κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό πρέπει να φέρουμε την πολιτική ευθύνη, για όλα αυτά και να είμαστε ξεκάθαροι σε τέτοιες εποχές συγκρούσεων σαν αυτές που ζούμε τώρα. Εμείς, ε, αν θέλουμε να αξιολογήσουμε μία κοινή ευρωπαϊκή λύση, να, δώσουμε, να της δώσουμε την αξία που έχει και να μην γυρίσουμε πίσω στις σκοτεινές εποχές. Αυτές είναι οι αρχές που χρειαζόμαστε σε αυτή την Ευρώπη για να μην ξαναβιώσουμε αυτές ε, τις ε, φρικαλαιότητες. Η ενότητα μέσα από την κατανόηση. Ναι, κάτι σημαντικό είναι προϋπόθεση της ευημερία. αλλά πάνω από όλα είναι η ετοιμότητα να συνεννοηθούμε και να είμαστε ανθρωπιστές, να μην δείχνουμε μόνο το δίκιο του δυνατότερου. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την ε, ευρωπαϊκή κατανόηση να κερδίσει έτσι ώστε να φανούν προς τα έξω αυτά που ενώνουν όλους εμάς ως Ευρωπαίους. Θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατική Ευρώπη και ισχυρές δημοκρατίες στην Ευρώπη. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό και είναι έμπνευση που θα υπάρχει και η μουσική συνοδεία σε αυτήν εδώ τη διάσκεψη. Θα πρέπει μέσα από αυτό να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε για περαιτέρω χρηματοδότηση όλων αυτών των πρωτοβουλειών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα των Νέων. Τέτοια πράγματα θέλουμε. Θέλουμε να ακούμε προσεκτικά ε, διάφορες φωνές, διάφορους ήχους, διάφορα χρώματα και συγχορδίες, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την αξία της πολυμορφίας, της ποικιλομορφία. Σας εύχομαι λοιπόν σε αυτή τη διάσκεψη ε, να υπάρχει δέσμευση για μια ενωμένη, δυνατή Ευρώπη, μια Ευρώπη της ειρήνης, ε, της ελευθερίας, ε, της δημοκρατίας, μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί από μόνη της να χτίσει το μέλλον της μέσα από την ενότητα. Ευχαριστώ. Thanks. A lot, Σας ευχαριστώ, Μόνικα, για αυτόν τον λόγο και που μιλείτε υπέρ του πολιτισμού. Και τώρα, Λιδία, η κυρία Λιδία Κονιόρδο, Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Your Excellency, Mr. President of the European Parliament. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεχότατε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αξιότιμη Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι υπουργοί, κυρίε και κύριοι. Τελεί τιμή για εμένα να παρευρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ταγιάννη για την ε, πρόσκληση του να συμμετάσχω σε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη. Αγαπητοί φίλοι, γνωρίζουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Φοβούμαστε όλοι ότι μπορεί η στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε αυτό που θεωρούσαμε πολύτιμο μπορεί να έχει έρθει, να έχει έρθει. και προετοιμαζόμαστε για ένα μέλλον αβέβαιο και θυμούμε το τίτλο ενός, μιας του ο Αγγελόπουλου το μετέωρο βήμα του πελαργού βρισκόμαστε σε μια στιγμή με διλήμματα και ουσιαστικές αποφάσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε και ατομικά αλλά πάνω απ' όλα συλλογικά. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα άλμα προς τα πίσω στον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία στην Αθήνα. Μια στιγμή στην πορεία της ανθρωπότητας όπου αναδύθηκε ο πολιτισμός και το πνεύμα από τον αρχαϊκό κόσμο στον νέο κόσμο, που έθετε ερωτήματα, που ζητούσε διάλογο, που, στην οποία υπήρχαν συγκρούσεις μέχρι και πόλεμοι, πλημμύ και ασθένειες, πανούκλες. Προσπαθούσαμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις παλαιές μορφές οργάνωσης, ε, την οικογένεια, τις πατρίε και να δημιουργήσουμε νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι τα σημαντικότερα έργα ποιητών και φιλοσόφων που σήμερα θαυμάζουμε γεννήθηκαν μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Σας, μιλώ για τις τραγωδίες, για τα, ε, το θέατρο που αναφέρονται στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναλογίες με τους καιρούς, του σημερινούς ο πολιτισμός μας ετοιμάζεται για άλλη μια φορά να κάνει ένα άλμα στην ιστορία του προς τα μπρος, προς ένα αβέβαιο και άγνωστο μέλλον και αυτό είναι ένα έφορο έδαφος αν θέλετε και ευκαιρίες, που δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες ε, εντελώς καινούριε και πρωτοφανείς σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο αντιλαμβανόμαστε πόσο αλληλένδετα είναι όλα, πόσο όλοι εξαρτώμαστε από, όλου, από όλους τους άλλους, πως όλοι αποτελούμε ε, μέλη αυτού του παγκόσμιου πλανητικού χωριού. Βέβαια, όπως θα περίμενε κανείς, αυτή η αβεβαιότητα γεννά και φόβο. Δημιουργεί ε, φυγόκεντρες τάσεις. Δημιουργεί ένταση της τάσεις μας να περιθεωρηποιούμαστε, να χαρακωνόμαστε. Για αυτή τη, στιγμή λοιπόν χρειάζεται να ανατρέξουμε στη σοφία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να αξιοποιήσουμε τα πολύτιμα υλικά αυτού της παλαιάς μας πορείας και να τα συνδέσουμε με το παρόν και το μέλλον, με τους νέους ανθρώπους, με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με την ε, ε, προστασία του περιβάλλοντος. χρειάζεται να χτίσουμε μια κυβωτό ως νέοι νόε για να προφυλάξουμε τον, τα πολύτιμα στοιχεία του πολιτισμού μας και να μην επιτρέψουμε να χαθούν εξαιτία της αίσθηση του επίγοντος και των τεχνολογικών αλλαγών. Θα πρέπει να συνδέσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά με τις σημερινές προτεραιότητες των καιρών μας, έτσι ώστε να μην τα σκεπάσει και να μην χαθούν εξαιτία αυτών των θορύβων και των, συζητήσεων άνευ νοήματος. Πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα για χρόνια σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι πλέον δεδομένα. Θα πρέπει να ξαναθέσουμε βασικά ερωτήματα στις, ε, για να λάβουμε αποφάσεις σε αυτό το σταδροδρόμι. να την μπορεί να προσφέρει ο πολιτισμός και η εκπαίδευση στους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα για να προφυλάξουμε αυτήν την εντυπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαιτερότητα. Τελούμε μια πολιτιστική νήσο με κοινέ αξίες, η οποία έχει ακτινοβολήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πολιτισμός είναι η συνδετική ουσία και χρειάζεται να υποστηρίξουμε τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες στις προσπάθειές τους, στην κινητικότητα τους. Πρέπει να ξαναθέσουμε τα βασικά ερωτήματα, αυτά τα βασικά διλήμματα και να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά με βάση τα, τις κοινέ μας αρχές και αξίες. Να λάβουμε συλλογικές αποφάσεις. Είναι δύο τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε. Η προσφυγική κρίση και το, τα, προστασία του περιβάλλοντος, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, τα οποία συνδέονται προσφυγική κρίση δείχνει τη, πόσο σημαντική είναι η ελληνική τώρα που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Εάν δεν δώσουμε τη σωστή απάντηση, έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος για να φουντώσει ο εθνικισμός, η ξενοφοβία. Όσον αφορά το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή μας δείχνει ότι η απάντησή μας θα πρέπει να είναι όχι μόνο οικονομική αλλά επίσης και πολιτιστική για να βρούμε πώς θα συνεχίσουμε να συνεπάρχουμε στο μέλλον. τη φίλοι, έχουμε κοινού μύθου και σύμβολα. Ορισμένα από αυτά έρχονται από την, ε, την αρχαία ελληνική μυθολογία, το Τροϊκό Πόλεμο, την ίδια. Πριν από λίγες μέρες, στην Σύνοδο του Βερολίνου για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά, προβήκαμε σε μια δήλωση για να δείξουμε τη δέσμευσή μας στην προστασία αυτή τη κληρονομιά, στην οποία συμμετέχουν ε, θεσμικοί παράγοντες, οργανώσεις από όλα τα, τα επίπεδα της κοινωνίας, που δήλωσαν ότι θέλουν να συνεργαστούν έτσι ώστε η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να προστατευτεί. Στη συζήτηση που έγινε εκεί, έφερα το εξή παράδειγμα, τα χωριά στο παρελθόν βοηθούσαν το άλλο, το ένα το άλλο, ε, για να ε, και έδειχναν αλληλεγγύη το ένα στο άλλο σε περιόδους λοιμών ή μεγάλων ασθενειών. Αυτό πρέπει να πράξουμε και σήμερα. Είναι ζήτημα κοινή λογικής. Απέναντι στα δύο μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να μάθουμε, να διδαχθούμε από το, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να ζητήσουμε από τους παλαιούς να μας βοηθήσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στο μέλλον. Και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν είναι απολύτω απαραίτητη η πολιτιστική κληρονομιά σήμερα. Δεν πρέπει κανεί να έχει την ψευδέστηση ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς αυτήν. Η ανάγκη ήταν για τους αρχαίους Έλληνε η πιο μεγάλη θεϊκή δύναμη. Ο πολιτισμός είναι αυτό που μας δίνει την ομορφιά, είναι επίσης η κοινή μας πηξίδα που μας δείχνει πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο πλοίο και να πορευόμαστε μαζί. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό για τη νέα γενιά που θα τους δείξει πώς θα μπορέσει και εκείνη να αφήσει το ίχνος της στο πλανήτη, στον κόσμο. Θα είναι εκείνοι που θα ζήσουν το μεγάλο, τη μεγάλη έκρηξη του πολιτισμού μας, είναι σε θέση, θα είναι σε θέση πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε τους νέους δρόμους προς την ευτυχία, την ελευθερία για όλη την ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα ζητήματα, αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ μεγάλα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κράτο ή οποιοδήποτε άτομο στην Ευρώπη ε, μεμονωμένα. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία επί τη βάση των αξιών μα, τη δημοκρατία, τη ε, αλληλεγγύη, τη ε, συμμετοχικότητα, τη φιλοξενία στο κέντρο των προσπαθειών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, Λίδια, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, οι τελευταίοι δύο μιλητές για αυτό το πρώτο πάνελ. Πρώτος, ο Υπουργός Πολιτισμού της Κροατίας. Ή Υπουργός, μάλλον, συγγνώμη, η κυρία Νίνα Ομπούλιαν Κόρτζινεκ. E, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. E, Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σήμερα παρίσταμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ομιλώ για αυτό το θέμα, γιατί ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί το θεσμικό όργανο. Είναι το θεσμικό όργανο το οποίο τόσες δεκαετίες έχει προλιάνει το έδαφος για τόσα θέματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα έχει εντάξει στο θεματολογιό του θέματα σχετικά με τον πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία μετά αναδέχτηκαν τα άλλα θεσμικά όργανα. Αγαπητοί φίλοι, η Ελληνίδα υπουργό. σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμια. Συμφωνούμε. Φυσικά και μας ε, σοκάρει η λέξη κρίση και γι' αυτό καλύτερα να μιλάμε για σταυροδρόμια. Γι' αυτό και σήμερα εδώ εορτάζουμε ε, την χρονιά της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μιλούμε για μια διαδρομή που πρέπει να κάνουμε οι Ευρωπαίοι όσοι πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό όραμα και που θέλουμε να είναι στέρεο, στεγανό και να βοηθήσουμε τους νέους Ευρωπαίους και έτσι να έχουμε μια κοινωνία οπότε οι δεσμοί αναμεταξύ μας να αναβαθμιστούν, να γίνουν πιο δυνατοί. Το ίδιο να ισχύσει και για τις κοινές μας αξίες και να δούμε τα θέματα που μας διαιρούν, που μας χωρίζουν, γιατί έχουμε διαφορετικά κράτη. Έχουμε τόσα θέματα επί των οποίων διαφωνούμε. Τη μετανάστευση, το ότι χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια, την Ευρώπη σε διάφορα επίπεδα, από διάφορε απόψει κλπ. κλπ. Αλλά έχουμε και τον πολιτισμό και η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα θέμα το οποίο μα ενώνει μας αποδεικνύει ότι όλοι είμαστε τμήμα αναπόσπαστο μιας οντότητας, ενός συνόλου. Κροάτης, Πορτογάλος, οτιδήποτε, ε, δεν αντιφάσκει αυτή η ιδιότητα με την ιδιότητα του Ευρωπαίου. Όλες οι ιδιομορφίες, οι ιδιοτυπίες, όλα αυτά ε, τα οποία μας κάνουν είμαστε τόσο κοντά στην ε, ταυτότητά μας, στην καταγωγή μας και είχαμε αυτή την συνάντηση κορυφής του ε, Βερολίνου την προηγούμενη εβδομάδα και γιορτάσαμε και εκεί το Ευρωπαϊκό του Κληρονομιάς και οπότε θα πρέπει σχετικά να ε, ευχαριστήσω την ε, Γερμανίδα ε, Υπουργό για την διοργάνωση αυτή και Ξέρετε, ως υπουργό, τι αισθάνθηκα στη συνάντηση κορυφή. Όλοι κάτι συμβάλλουμε σε αυτήν την υπόθεση, αλλά με μεγάλη είδαμε ότι υπάρχει ο πόθος του να ενατενίζουμε αυτά που μας ενώνουν, τα κοινά μας στοιχεία. Ο πολιτισμός δηλαδή και η πολιτιστική κληρονομιά. Όλα αυτά τα οποία κάνουν τους πολίτες να προσέχουν τον πολιτισμό, να μπορούν να καταλάβουν την κοινή ευρωπαϊκή διαδρομή. Όλοι όσοι έλαβαν μέρος σε εκείνη τη συνάντηση κατέληξαν στο ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα προγράμματα. Η καινοτομία είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για τον πολιτισμό. Επίσης, είπαμε ότι μας προβληματίζει το ότι κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα δεν προβάλλονται στις μικρότερες κοινότητες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να το καλύψουμε στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, ήταν ευρία η συνένεση και η υποστήριξη του θεματολογίου για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και ο Επίτροπος Ναύρασης το εξήγησε καλά. Για οπότε πρέπει να βρούμε ποια είναι η εύστοχη ισορροπία μεταξύ του να δούμε τι θα γίνει με τις προτεραιότητες που είχαμε τάξει στο παρελθόν και από την άλλη μεριά να περιλάβουμε τώρα κάποια νέα θέματα σε αυτό το θεματολόγιο των προτεραιότητων. Επίσης, κάποιοι από τους προλαλήσαντες το είπαν και εγώ το τονίζω το πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα δράσης για την πολιτιστική κληρονομιά. Ε, εννοείται ότι πρόκειται αυτό να είναι ε, το κληροδότημα ή ένα από τα κληροδοτήματα αυτής της χρονιάς για τον πολιτισμό. Τώρα, κάτι άλλο, κάτι άλλο το οποίο κατάλαβα στην συνάντηση κορυφής ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων, όλων των θεσμικών οργάνων μεταξύ των κυβερνήσεων μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον πολιτισμό. Να υπάρχει συνεργασία με τη των πολιτών. Γι' αυτό και εγώ νιώσα μεγάλη ικανοποίηση που διαπίστωσα ότι είχαμε δύο διάσημους παγκοσμίου βελληνικούς ε, καλλιτέχνες που ήταν εδώ κατά την ε, έναρξη της ε, σημερινής εκδήλωσης έχει φύγει βέβαια ο κύριο Ζώρα, αλλά μιλήσαμε πριν ε, μπει στην αίθουσα, πριν μπει στο ημικύκλιο και μου ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο που προσεκλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή εκδήλωση ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα αποφασιστεί γιατί όλος ο κόσμος συναντενίζει το τι κάνει η Ευρώπη στο τι έχει επιτελέσει η Ευρώπη στο μέτωπο του πολιτισμού και να δούμε τι ρότα θα πάρει η Ευρώπη γιατί είμαι πεπισμένος ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θεσμικό όργανο και σίγουρα ήταν πολύ σημαντική η συμβολή πρωταγωνιστική στα θέματα του πολιτισμού το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πολιτισμικό πλαίσιο που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Thank you very much, Nina. The last speaker. Ευχαριστούμε την Νίνα. Τελευταίο, τελευταία ομιλία από την Λετωνία, Υπουργείο Υπολιτισμού, Ντάσε Μελπαερντέ. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συμμετέχοντες ε, στη διάσκεψη. Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω την ε, παράδοση του τραγουδιού στις βαλτικές χώρες. Γι' αυτό θα σας μιλήσω για την ισχύ του πολιτισμού και τη δυνατότητα να φέρει θετικές αλλαγές. Γι' αυτό το λόγο θα σηκωθώ όρθια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 klausījās Σε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι από τη Λετανία, ε, Λετωνία λέει η τραγουδίστρια ότι διάλεξε ένα ψηλό σημείο έτσι ώστε η φωνή της ε, να ακούγεται μακριά πάνω από τα λιβάδια και τα όρη και τα βουνά. Έτσι και εγώ λοιπόν σήμερα στέχω, στέκομαι εδώ σε αυτό το ψηλό σημείο ντυμένη με την παραδοσιακή στολή της Λετωνίας του 18ου αιώνα για να σας δείξω την ισχύ της παράδοσης της χώρας μου. Στη... Το έθνος μας, ε, το τραγούδι, είναι η πιο ε, καλά φυλαγμένη παράδοση. Έχουμε πάρα πολλά φολκλωρικά τραγούδια και ε, έτσι ε, θεωρούμε ότι εδώ και πάνω από 150 χρόνια ε, η καλύτερη εκδήλωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι αυτά τα φεστιβάλ που κάνουμε με χορό και τραγούδι. Κάθε πέντε χρόνια γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Την Κυριακή έχουμε το 26ο φεστιβάλ. Μπορείτε να έρθετε λοιπόν. Φανταστείτε σε μια ανοιχτή σκηνή 16.000 τραγουδιστές να χρησιμοποιούν τη μέθοδο καπέλα για να τραγουδήσουν ε, μια σειρά από τραγούδια με τα παραδοσιακά όργανα της Λετωνίας ε, σε ένα τεράστιο διεθνές ε, στάδιο. Επίσης, πέρα από το τραγούδι, η παράδοση ενώνει τους ανθρώπους από όλες τις περιοχές, τη διασπορά μας, το εξωτερικό, αλλά και τους φιλοξενούμενους μας από όλο τον κόσμο. 40% του πληθυσμού της χώρας άμεσα εμπλέκονται στη, στην διάσωση της κληρονομιάς μας και πάρα πολλοί από αυτούς εμπλέκονται σε αυτό έμεσα. Τα φεστιβάλ που κάνουμε με τραγούδι και χορό γίνονται παντού και η μοναδικότητά τους αναγνωρίστηκε το 2003 όταν η UNESCO μίλησε για το συμβολισμό των χωρών και των του τραγουδιού στην Λετωνία και την Εστονία και στις βαλτικές χώρες. Είναι κομμάτι της άειλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και αυτό ακριβώς μας θυμίζει το τραγούδι και ο χορός στις βαλτικές χώρες, ότι το τραγούδι και ο χορός μας ενώνουν όλους εδώ στην Ευρώπη. Μπορούμε να βρούμε ε, στις ρίζες αυτών των εορτασμών με τραγούδι και χορό τις κοινέ πηγές της ευρωπαϊκής ε, ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Μαρτίνος Λούθυρος ακριβώς έφερε αυτή την αναμόρφωση στην θρησκεία. Η οι διάφορες ε, παραδόσεις ε, που ε, προέρχονται από την περιοχή της Μοραβίας επίσης μας δείχνουν έναν αντίστοιχο δρόμο. Έτσι λοιπόν η παράδοση στη Λετωνία πέρασε μέσα από τα φεστιβάλ, από τους εορτασμούς από το 19ο αιώνα μέσα από τους μετανάστες από τη Γερμανία και την Αυστρία. Για πάνω από 150 χρόνια αυτή η παράδοση με τους εορτασμούς έπαιξε πολύ κεντρικό ρόλο στην διαμόρφωση του έθνους ε, και της ταυτότητάς μας ως ε, κράτος. Μας έσωσε κοινωνικά και πολιτικά. Είναι μια συμβολική πνευματική έκφραση της ταυτότητάς μας, ε, της ενότητάς μας ως έθνος. Έγινε λοιπόν ένα ισχυρό εργαλείο της μη βίαιης αντίστασης κατά την Σοβιετική κατοχή και ε, είχαμε και την ε, αντίστοιχη επανάσταση μέσω τραγουδιού στα βαλτικά κράτη ε, μαζί με την Λιθανία και την Λετωνία θα γιορτάσουμε την, τα 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν η ισχύς του τραγουδιού μας ξαναέφερε εδώ στην ευρωπαϊκή κοινότητα για να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές ε, κουλτούρες και πολιτισμοί. Μόνο δική μας κουλτούρα και πολιτισμός υπάρχει που μας ενώνει ε, όλους ε, στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Thank you very much. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε εντυπωσιακοί, Υπουργό. Avant de descendre πριν να κατεβούμε για την οικογενειακή φωτογραφία, θα ήθελα να σα ενημερώσω λίγο για τι εκδηλώσει που προβλέπουμε για απόψε. Μετά τη φωτογραφία θα δούμε το ρεπορτάζ του ARTE Άρτε σχέση με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τον πολιτισμό, τη χρονομηχανή της Βενετίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο Πρόεδρος, τους διερμηνείς που θα διερμηνεύσουν το βίντεο με βάση τους υποτίτλους. Ε, ευχαριστούμε. Οπότε και τώρα ξεκινούμε στη συνέχεια το πάνελ, το οποίο πρόκειται να το προεδρεύσει η κυρία Σιλία και έχουμε επίσης ε, ως προσκεκλημένο τον ε, μαέστρο Έτζιο Μπόσο, τον οποίο ευχαριστώ. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ο οποίος πέραν των άλλων ε, ταλέντων είναι κάποιος που είναι πάντοτε χαμογελαστός και δίνει σε όλους ε, κουράκι μας έχει δείξει το πώς κερδίζονται οι μάχες Καλώς όρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο go downstairs for the picture, exactly for the family photo. Thank you very much. Τώρα θα βγάλουμε την οικογενειακή φωτογραφία, λέει ο πρόεδρος.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 Εδώ και χρόνια μετά την ψηφιακή επανάσταση αρχίσαμε να συλλέγουμε χιλιάδες, δισεκατομμύρια δεδομένα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας και ξεκινήσαμε να τα συλλέγουμε σε μεγάλα δίκτυα, τα οποία σήμερα φιλοξενούν αυτό που ονομάζουμε big data, μαζικά δεδομένα. Μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι αυτή η ψηφιακή επανάσταση αναφερόταν μόνο στο, στο παρόν και το μέλλον, χωρίς να προσπαθούμε να περάσουμε το σύνορο προς το παρελθόν. Συλλέγετε τις πληροφορίες από το παρελθόν και τις συγκρίνετε με εκείνους του παρελθόντος. Και ε, δημιουργείται κάτι το οποίο μοιάζει με μανιτάρι. Έχουμε τα μεγάλα δεδομένα του παρόντος από στο πάνω μέρος και προς τα κάτω έχουμε τα δεδομένα που αφορούν στο παρελθόν. Είναι πολύ σημαντικό τα δεδομένα του παρελθόντος να είναι εξίσου προσβάσιμα με εκείνα που αφορούν στο παρόν. Για να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή, μια συνεργασία μεταξύ του Πολυτεχνείου της Λοζάνης και του Πανεπιστημίου Καφουσκάρη στην Βενετία έκανε ένα project πολύ ε, φιλόδοξο, τη χρονομηχανή της Βενετίας ένα ε, σύστημα με το οποίο προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε 80 χιλιόμετρα αρχείων στη Βενετία. Το κράτος της Βενετίας πριν την κατάρρευση του 1797, ήταν ένα από τα κράτη με την καλύτερη δημόσια διοίκηση, διοίκηση ε, στην παλαιά Ευρώπη. Οι Βενετσιάνοι ήταν το Google του Μεσαίωνα θεωρούσαν ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορεί κανεί να βρει από πού έχει προέρθει οποιαδήποτε πληροφορία και δημιουργούσαν τεράστια αρχεία προ αυτό. Με αυτό το σύστημα λοιπόν, με αυτό το αρχείο, έχουμε στη διάθεσή μας χιλιάδες δεδομένα, μία μηχανή η οποία μας επιτρέπει να πάμε 10.000 χρόνια πίσω. Έχουμε μια τεράστια βάση δεδομένων, όμως πρέπει να αξιοποιηθεί, πρέπει να την, ε, να, την κάνουμε λειτουργική. Η χρονομηχανή της Βενετίας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ε, τετρατιστιάστατα μοντέλα της ιστορίας. Δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες υποδομές. Οι δυνατότητε που μα δίνουν αυτά τα συστήματα προκαλούν ήλιγκο. Μα δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Είναι εξαιρετικά πυκνά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η τεχνολογία αλλάζει, αλλά σε λίγα χρόνια αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούμε θα είναι παροχημένα, όμως οι ιδέες είναι, ε, παραμένουν και θα, το ζήτημα είναι να, παρα, να ε, παραμείνουν προσβάσιμες με τρόπο δημοκρατικό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά κυρίως για την κοινωνία. Now... Ο πρόεδρος. Και τώρα, καθίστε παρακαλώ. Sit down. Now we start with the panel number one, cultural heritage. Με τώρα το πρώτο πάνελ για την πολιτική κληρονομιά, την ευρωπαϊκότητα θα προεδρεύσει η Σίλβια Κώστα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τον πολιτισμό δηλαδή. Συνεχίζω στα Ιταλικά Πρόεδρε και πότε φορέστε τα ακουστικά σας να ακούσετε την μετάφραση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ γιατί έχουμε το, την εκδήλωση του Μιλάνου. Είναι μια μεγάλη ε, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο. Ούτω ώστε έτσι να κλείσουμε την Ευρωπαϊκή Χρονιά της Κοινωνίας επίσης. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που μιλήσαμε εδώ Έχουμε τον κύριο Γιούγκερ και έχουμε όλους τους εκλεκτούς εδώ προς μα μας και θέλω να σας πω κάποια σημαντικά για την σχέση μεταξύ πολιτικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της ε, ηλικής και άειλης και επίσης την ε, αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη. Γιατί είπαμε ότι θα θεσπίσουμε αυτή τη χρονιά. Θα είναι αφιερωμένη στον ε, πολιτισμό. Τώρα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, την ευρωπαϊκή πορεία, θα πρέπει τώρα να δούμε το ότι το ευρωπαϊκό όραμα της ελευθερίας, της ανάπτυξης, της δημοκρατίας έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Αλλά όμως ε, επίσης ένα αμφιβόλο έχουν τεθεί και οι ρίζες, η ταυτότητα, ο κοινός, ο κοινός προορισμός της Ευρώπης που αφορά και εμάς και όσους ενατενίζουν την Ευρώπη και έρχονται σε αυτήν και δεν βρίσκουν πάντοτε την ε, αλληλεγγύη που επιβάλλει η ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και ρωτήθήκαμε, γιατί όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλή αυτή η ερώτηση, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Μα τι άλλο, αν όχι η τέχνη, ο πολιτισμός, η πνευματικότητα, η αρχιτεκτονική, οι εκκλησίες μας, η μουσική, η φιλολογία, το θέατρο και το σινεμά δίνουν αναγνωρισιμότητα στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και δημιουργούν αυτή την αίσθηση του ανήκειν στους Ευρωπαίους. Τι άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει θεμέλιο του ευρωπαϊσμού, την περισσότερη συνειδητοποίηση αυτού, γιατί έχουμε αυτήν την ενότητα, στην πολυμορφία. Είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο, αλλά έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Πέρασε μέσα από τραγωδίες, διαιρέσεις από τη μία γενιά στην άλλη. Και σε σχέση με αυτές τις τρεις ε, έννοιες, αδελφότητα, ισότητα, ελευθερία, μα τι είναι περισσότερο ελευθερία από το να υπάρχει καλλιτεχνική δημιουργία, ισότητα στην ε, συμμετοχή, περισσότερη αδελφότητα, από το να μπορεί κανείς να μοιραστεί την ομορφιά και την αρμονία. Ξέρουμε περισσότερο από όλους οι καλλιτέχνες ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της ε, πολιτιστικής πληρομορφίας και της επιβεβαίωσης της κοινή ευρωπαϊκής ταυτότητας που βασίζεται στις κοινέ αξίες όπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελληνική, το κράτος δικαίου. έτσι αναγνωρίζεται η δημιουργικότητα, δίνεται μια δίκαιη αμοιβή ε, και δίνεται επίσης και η ελευθερία στη δημιουργία για τους καλλιτέχνες. Σήμερα έχουμε γίνει οραματιστές και άλλα και μάρτυρες όπως ε, ε, αποδεικνύουν όλα αυτά τα προγράμματα γιατί έχουμε τώρα τους συνομιλητές μας της κοινή προσπάθειας όπως είδαμε για το φόρουμ του Μιλάνου αλλά και για τις έντες του Βερολίνου και έτσι θα κλείσει και με κάποια διακοινοβουλευτική εκδήλωση αυτό το έτος. Θα συμμετάσχουν όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. Να το κληροδότημα αυτής της χρονιάς. Είχαμε πολύ επίπεδη και καλύψαμε όλους στη διαχείριση και διακυβέρνηση αυτής της χρονιάς. Υπάρχει πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ πολιτικής κληρονομιάς και του ανήκειν στην Ευρώπη. Κοινέ εμπειρίες, ρόλοι και διαφορετικές χώρες. Πρώτα-πρώτα. Όμως, επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλώς όριζε κάποιος ξεχωριστός καλεσμένος. Ο μαέστρος, ο διευθυντής ορχήστρας, έτσι όπως ένας πάρα πολύ σπουδαίος διευθυντής ορχήστρας, είναι συνθέτης αλλά και μουσικός. Έχει διευθύνει σπουδαίες ορχήστρες έχει δουλέψει διεθνώς αλλά και την ε, London Symphony Orchestra έχει διευθύνει αλλά και φέτος στην Ιταλία έχει αναδειχθεί και θα πρέπει να του δώσουμε τον ε, λόγο. Είχαμε πάντως πριν από λίγες μέρες μία συνέντευξη που είπατε κάτι εντυπωσιακό ότι ένας μουσικός αναγκαστικά γεννιέται Ευρωπαίος γιατί η μουσική κουλτούρα ορίζει την ε, Ευρώπη ε, ακριβώς όπως η οικονομία τα κρατεί. Οπότε θα πρέπει να δώσω τώρα το λόγο και να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Hello. Hello. Ciao. Scusate, ma paura. <laughs> Sono abituato a star di schiena a fare musica facile. Vedete, ah, c'è Υπάρχει κάτι για τη μουσική, εκεί που ανήκω. Τη μουσική, την κλασική. Είναι κάτι που τη συνοδεύει. ένα βρέφος. Είναι σαν να το συνοδεύει παντού η μουσική, ένα βρέφος Ευρω... την Ευρώπη. Αγγίζει για τα βρέφη μουσική. Είτε προέρχονται από τη Γερμανία, την Αυστρία, την ε, Γαλλία. Να, ποιος. Ο Ντεμπισί, ο Μπραμς, ο Μέντελσον. Δεν υπάρχουν όρια και σύνορα. Η μουσική είναι κάτι που διαπερνά όλους. Είναι κάτι που ξεπερνά τα σύνορα. Εδώ και αιώνες. Έκανε κάποιος 100 χιλιόμετρα για να ακούσει τον ε, Μαρτσέλο ή του, του Μπαχ ή του Σούμπερτ που έδωσε την τελευταία του δεκάρα για να πάει να ακούσει Παγκανίνη. Και, και όχι επειδή ε, ήταν ε, Ιταλός ο Παγκανίνη, αλλά για να ακούσει το βιολί του Παγκανίνη. Να, έτσι θα κάνουμε την υπέρβαση. Με την ταυτότητά μας. η ορχήστρα την οποία διευθύνω είναι μια Ιταλική ορχήστρα αλλά ο πρώτος βιολιστής, το πρώτο βιολί είναι Ρουμάνος, ένας πιο άλλος είναι Ούγγρος οπότε τελικά πρόκειται απλά για μια ορχήστρα έτσι θα το πράγμα, είμαστε αφελείς γιατί πολλές φορές αργούμε να ανακαλύψουμε τα πράγματα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε αγωνιστεί και αυτό περνάει από το μυαλό μου. Να γιατί ο Μπετόβεν έγραψε μουσική για την Ευρώπη, την οδή στη χαρά. Και από την άλλη μεριά, ενώ μαθαίνουμε λέξεις τόσους, συγγνώμη, γλώσσες τόσους αιώνες, τελικά η μουσική μιλάει όλες τις γλώσσες. Φρόιντε, χαρά. Αυτό θυμίζει και τη λέξη φίλος. Συνύπαρξη. Δηλαδή, Οπότε η οικοδόμηση αυτή είναι ο αρχιτέκτονας της Ευρώπης, της, του οράματος. Μέντελσον είδε την Ιταλία και έγραψε την συμφωνία στην οποία περιγράφει τη χώρα. και ο Τσακόφσκι το ίδιο. Είδε τον παράδεισο στην Ιταλία και εμπνεύστηκε από όσα είδε. Να, η διαφορά στην Ευρώπη τόσο σημαντική και άρα θα πρέπει να φροντίζουμε να προστατεύουμε την πολιτική μας κληρονομιά. Είναι οι ευρωπαϊκές ρίζες και κυρίως η μουσική καταργεί τα σύνορα, όλα τα σύνορα. Και προβάλλει την Ευρώπη σε όλο τον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να θυμηθούμε για κάποιον άλλον, Κλάουντι Άμπαντα. 40 anni fa Έχουμε τώρα την ορχήστρα των ε, νέων. Η νέα ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτοί μας μαθαίνουν ότι είμαστε μια ορχήστρα. Η Ευρώπη είναι μια ορχήστρα. Και οι ρίζες για τις οποίες ε, μίλησα δεν είναι κάτι μονολυθικό, κάτι μονοδιάστατο, είναι κάτι που απλώνεται και πάει βαθιά. Γι' αυτό σας λέω. Και σκεφτείτε πώς λέγεται αυτό το μέρος που βρισκόμαστε. Κοινοβούλιο, παρλαμέντο. Ε, άρα ο λόγος είναι το πιο σημαντικό. Ο λόγος τον οποίο πρέπει να ακούμε. Να ακούει ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα προβλήματα. Αυτό είναι η ευκαιρία που δίνεται με τη μουσική. Πιστέψτε με, πιστέψτε στην Ευρώπη, πιστέψτε. Penso, grazie, grazie maestro. Η κυρία Κώστα, ευχαριστούμε. Μα συγκίνησε όλους. Δύο κοβέντες μόνο για στιγμή για να δώσουμε στο άλλα μέλη του πάνελ το λόγο. Απλώς για να ανέδειξω κάτι. Ίσως θα πρέπει πιο συχνά να το λόγο καλλιτέχνες να μιλούν για την Ευρώπη. Γιατί λένε πράγματα πολύ σημαντικά. Σας έχει ανάγκη εσάς τους καλλιτέχνες ε, η Ευρώπη. Εσείς, οι άνθρωποι της δημιουργίας, οι διανοούμενοι. Είσαστε η φωνή, είσαστε η εκδήλωση του τι είναι και τι μπορεί να γίνει η Ευρώπη. Έχεις δίκιο. Εδώ είναι το, το Παρλαμέντο, εδώ είναι το Κοινοβούλιο, εδώ που θα πρέπει να ακούει ένα τον άλλο. Το, la parola, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, που μείνατε μέχρι τώρα. Πρέπει τώρα να αποχωρήσετε. Δίνουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Έχουν θέματα πολύ σημαντικά, ενδιαφέροντα. Θέματα πολιτιστικά, είναι και πανεπιστημιακοί. Ε, πρώτα πρώτα ο Χέρμαν Πάρτσιγκερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ιδρύματος για την ε, προσική πολιτική κληρονομιά. Εκείνος με το Ευρωπανόστρα οργάνωσαν την εκδήλωση του Βερολίνου και ήταν υπέροχη αυτή η πρωτοβουλία που αναλάβατε. Αυτό το call to action κάτι σαν ψήφισμα που όλοι το προσυπογράψαμε ιντερνετικά. Όλη η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της χώρας σας, όλοι οι υπουργοί, πρόκειται για ένα κάλεσμα, μία πρόσκληση. Να μην ολοκληρώσουμε αυτά που κάνουμε τον Δεκέμβριο φέτος. Απλώς αυτό να είναι η απαρχή μιας νέας φάσης για την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική. Yeah, thank you, Ευχαριστώ Σίλβια, μέλη του Κοινοβουλίου, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούσαμε ακριβώ ε, όλα αυτά τα πράγματα που άκουσαν και οι υπουργοί την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο. Το είπε ο Επίτροπος, το είπαν ε, οι υπουργοί της Ελλάδος, της Κροατίας. Ε, Οπότε, να συνεχίσω λέγοντας ότι η διεκδήλωση του Βερολίνου είναι ε, μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση γιατί θέλει να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Και όντω ήρθαν 1500 άτομα, πάνω από 100 θεσμικά όργανα, κυβερνητικά όργανα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών ε, και συμμετείχαν σε 70, διαφορετικά, ε, σε 70 διαφορετικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ε, και τα λοιπά. Επίσης είχα εγώ ως εκτελεστικός διευθυντής της Ευρώπα Νόστρα και ως πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Πολιτιστική Κληρονομιά, του Προσικού μάλλον, ε, ήμουν εκεί ε, ως ο αμφιτρίωνας. Είχαμε λοιπόν πολλά θέματα. Καταρχάς να παρουσιάσουμε την πολιτιστική κληρονομιά και από την άλλη να, το, να τη χρησιμοποιήσουμε ως όπλο για την πολιτική την πολιτιστική κληρονομιά έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια κόλλα, ένα συνδετικό κρίκο για την Ευρώπη. Να χτίσουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες μετά από την οικονομική κρίση, την κρίση των προσφύγων, το λαϊκισμό, δείχνει ξεκάθαρα ότι η οικονομική ευημερία είναι η βάση της καθημερινής ζωής, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό. Ε, το πράγμα που θα πρέπει να μας ενώνει. Ειδικά σε μια περίοδο κρίσης η ίδια Ευρώπη προσπαθεί να επιβιώσει και να μείνει ε, ενωμένη. Όμως χρειαζόμαστε κάτι άλλο για να μας ενώσει. Νομίζω η πολιτιστική κληρονομιά και ο πολιτισμός αυτό ακριβώς το δυναμικό ε, έχουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα από την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης. Ε, το ακούσαμε και στο Βερολίνο. Παρακαλώ, α υπογράψουμε όλοι. Είναι εύκολο στο ίντερνετ να υπογράψουμε για την προτεραιότητα που έχει η πολιτιστική κληρονομιά. Ε, για το πώ μας βοηθά να συνδέσουμε τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών. Η πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές είναι η ενσωμάτωση. Είναι διπλό το πρόβλημα. Ε, ενσωμάτωση και ολοκλήρωση σε επίπεδο Ευρώπης μεταξύ ημών και ταυτόχρονα έχουμε και τόσο κόσμο που έρχεται απ' έξω. Εμείς που μένουμε εδώ πρέπει κάπως να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Διπλή μορφή ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης. Η εκπαίδευση, η πολιτιστική κληρονομιά είναι κατά κάποιο τρόπο υλοποιημένη ιστορία. Αν θέλεις να δεις τι είναι η ιστορία θα δεις τα μνημεία, τις εκκλησίες. Αυτό ακούω από πολλές χώρες. Η εκπαίδευση και η ιστορία στην τέχνη στον πολιτισμό είναι ένα θέμα παντού. Η προσβασιμότητα, η συμμετοχή μέσω του ίντερνετ οι αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες και τέλος ε, οι πολλές οπτικές γωνίες. Όλοι πρέπει να υποφεληθούμε από το γεγονός ότι ως Ευρωπαίοι μπορούμε να υποφεληθούμε από διαφορετικές δράσεις και συμβάντα της ε, ιστορίας, να μάθουμε από την οπτική των άλλων. Έτσι λοιπόν για μένα το να αντιμετωπίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά είναι κομμάτι της ειρήνης και είναι το μόνο μέλλον που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει σχετικά το χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας από του επόμενου. Αλλιώ δεν θα τα καταφέρουμε. Οπότε ευθύς να δώσουμε το λόγο στην Αν που είναι η Γενική Διευθύντρια του καναλιού Αρτέ. Προογάγει τον πολιτισμό μέσω των προγραμμάτων ε, εκπέμπει σε έξι γλώσσες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει ήδη βρισκόμαστε στην τρίτη χρονιά. Και έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα ε, που σας αφορά, που είναι η Δημιουργική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη σημαντική ημέρα, συμβολική. Και Έχω την χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτω από το βλέμμα της Σιμών Βέιλ και να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις σημαντικών καλλιτεχνών καθώς επίσης και των πρόεδρων των θεσμικών οργάνων. Και επίσης ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει οργανώσεις με τις οποίες υπερασπίζονται την πολιτιστική μας κληρονομιά και ακούσαμε επίσης ότι θα αυξηθούν και τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον για τον πολιτισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καλό νέο. Βλέπετε λοιπόν την σημασία της πολιτικής πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι, πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Το Άρτε από πάντοτε θεωρούσε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος του πολιτισμού. Είμαστε δηλαδή από τη δική σας τη μεριά, από την μεριά εκείνων που είναι πεπισμένοι ότι ο πολιτισμός μπορεί να αξιοποιήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες για να απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πράγμα ήδη εδώ και 26 χρόνια ως κανάλι έχουμε δει προσπαθήσει να επιδείξουμε όλη τη διαφορετικότητα που υπάρχει στην Ευρώπη μέσω των προγραμμάτων μας, τα οποία διανέμονται σε όλη την Ευρώπη και ε, δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αναφέρει στην έκθεση που ενέκρινε πριν από δύο εβδομάδες σε σχέση με τα δομικά συστηματικά εμπόδια που υπάρχουν στον χρηματοδότηση και που περιορίζουν την διάδοση του πολιτισμού. Αναφέρει λοιπόν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε να υποστηρίξουμε την πολυγλωσία. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινήσαμε εδώ και κάποια χρόνια στο Άρτε μια υποστήριξη στην πολυγλωσία προσπαθώντας να ε, μεταφράσουμε τα προγράμματά μας σε διάφορες γλώσσες και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και την ψηφιακή ε, τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή έχουμε από το 2015 διάφορα κανάλια στα αγγλικά, στα ισπανικά και από το 2016 στα πολωνικά και προετοιμάζουμε και την έκδοση του Άρτε στα Ιταλικά. Με αυτόν τον τρόπο απευθυνόμαστε στο 70% των Ευρωπαίων πολιτών στην ε, μητρική τους γλώσσα. Επίσης ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε και την πολιτιστική κληρονομιά, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτού του ε, προγράμματος για λόγους χρόνου, όμως όπως ε, τα ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Μπάρεμποϊμ, όπως έλεγε και ο Μιτεράν, έχει τεράστια σημασία για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο πολιτισμός. Και προσπαθούμε να συνεχίσουμε να είμαστε το ευρωπαϊκό ε, κανάλι το οποίο επιτρέπει να έρχονται πιο κοντά οι, οι λαοί της Ευρώπης, όλο και πιο κοντά, όπως αναφέρουν και οι συνθήκες. Σας ευχαριστώ. Λυπούμε. για να καταλάβετε πώς ε, δυσκολευόμαστε. Καμιά φορά μέσα ένα λεπτό ή δύο λεπτά για να μιλήσουμε. Βλέπετε, ε, άρα μπροστά σε αυτό τα δύο λεπτά είναι πάρα πολλά. Ε, γιατί είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω για το χρονοδιάγραμμα και έχουμε ακόμα ε, δύο πάνελ και τώρα έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, τον Ρικάρντο Ριβέρο Ορτέγα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Μπορούσαμε να δούμε ακριβώς τι ρόλο διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη για την επιδίωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τόσο ώστε να μεταλαμπαδευτεί σε επόμενες γενιές. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο. Ε, χαιρετίζω όλους όσους ήρθαν εδώ στο πάνελ. Ε, κλείνουμε 800 χρόνια. Εργαζόμαστε για να μεταναμπαδεύσουμε, όπως είπατε, τον πολιτισμό. Θα πρέπει να μάθουμε στους νέους τι πάει να πει η Ευρώπη, ποια είναι η πολιτική κληρονομιά. Επίσης όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Να το προσέξουν οι νέοι. Έχουν πολλά να μας πούν και πολλά να μας δείξουν. Είναι ο πλούτος μας, είναι η νεολαία, οι δυνατότητές τους για το καινούργιο. Έχουμε προτάσεις που ξεπηδάνε από τα πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο ήταν πάντα η πηγή της αιώνιας νεότητας. Δεν είναι θέμα ηλικία. Δεν είναι θέμα του πόσα χρόνια γράφει η ταυτότητα. Είναι θέμα μυαλού, νοοτροπία, πνεύματο. Πάρα πολύ αρχαία. Παλιά Ευρώπη, αλλά αισθάνεται νέα. Θα πρέπει ο πολιτισμός να ξυπνά το συνέστημα. Είδαμε πόσο εύλογα μας τα είπε ο κύριος Μπόσο. Μουσική, φιλολογία, ποίηση και το πανεπιστήμιο τα κάνει όλα αυτά. Οπότε θα πρέπει βεβαίως να μεταδίδει τις αξίες, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Μας το υπενθυμίζουν τα θεσμικά όργανα, αλλά εμεί ανέκαθεν ε, πιστεύαμε στο έρασμος. Κινητικότητα 800 ετών για φοιτητέ και για καθηγητές. Ε, θυμάμαι πριν από 20 χρόνια ήμουν εδώ. Πήγα στο 10ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στο Φράιμπουργκ. Επομένω, κινητικότητα για διανοούμενου πνευματικού ανθρώπου, άντρε, γυναίκε και αξίε έτσι αναδεικνύονται η κληρονομιά, το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει η Ευρώπη να ανανεώνεται, να προσαρμόζεται τις βασικές ιδέες, τις αναπαλωτρίωτες, όπως η ισότητα ανδρών γυναικών και είχαμε εδώ και 500 χρόνια την πρώτη καθηγήτρια και παρά την τότε απαγόρευση ήρθαν να σπουδάσουν πρώτες γυναίκες. Έτσι ξανοιγόμαστε στις ε, πραγματικότητες και δεν θα ήταν η Ευρώπη αλλιώς αυτή που είναι το κέντρο, το επίκεντρο της δημιουργίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που τρίσατε το χρονικό ε, περιορισμό, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, όπως τα λέτε, όπως τα λέτε για το πνεύμα και πώ πρέπει να ξυπνάει. Και τώρα έχουμε την Κωνσταντζη που είναι η διευθύντρια του μουσείου που ονομάζεται 20 Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι ανανεώνονται οι ευρωπαϊκές αξίες με τέτοια μουσεία. Πέστε μας την εμπειρία σας. Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι φιλοξένομοι, θα ήθελα να μιλήσω ε, και να αναφέρω τρία σημεία σχετικά με την έκθεση στο δικό μας ε, οίκο για την πολιτιστική κληρονομιά. Πώς σώζουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, πώς ένα μουσείο μπορεί να συμβάλλει σε κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος επαφών. Πολλές μικρές πολιτικές οντότητες συνεπάρχουν σε μια πολύ μικρή ήπειρο. Αυτό δημιούργησε πολλές ε, ε, δυνατότητες και για σειράξεις αλλά και για επαφές με ταξί ανθρώπων από διαφορετικό εθνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων μονάδων. Έτσι λοιπόν στην πρώτη μας ε, έκθεση ακριβώς αυτό δείξαμε πώς ε, η Ευρώπη διαμορφώνεται από το περιεχόμενό της. Αυτό που βλέπουμε ως κοινή η ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι προϊόν και αμοιβαίας επιρροής. Η ε, πολιτιστική κληρονομιά έχει μια ισχυρή υπερεθνική διάσταση. Ακόμα και αν ε, περιγράψουμε τον πολιτισμό σε ένα ε, τοπικό φαινόμενο, δεν υπάρχει κανένα κομμάτι που να μην είναι και διαπολιτισμικό, διεθνικό. αυτό που θέλουμε να διατηρήσουμε είναι το παρελθόν, γιατί για να έχουμε ένα μέλλον. Υπάρχει συνένεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινή Κληρονομιά. Η μόνιμη έκθεσή μας, λοιπόν, θέτει μία πρόταση σχετικά με το τι είναι ακριβώς αυτή η κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ζητάμε από τους ε, επισκέπτες να φτιάξουν ακριβώς, ε, να δώσουν τη γνώμη τους. Η, Ευρώ, η Ελλάδα, η Ρώμη, ο χριστιανισμός, ε, αλλά και η απεικιοκρατία, η σκλαβιά, οι γενοκτονίες είναι πράγματα που παρουσιάζονται. Τα μεν πιο εύκολα τα αποδέχεται κανείς, τα άλλα όχι. Όμως η Ευρώπη θα πρέπει να αποχωριστεί το δινηρό της παρελθόν και να μιλά για μια κληρονομιά η οποία είναι ε, πιο επικοδομητική. Ως μουσείο λοιπόν θέλουμε μια ε, σκέψη να δημιουργήσουμε σχετικά με, την ευρω... με την εξευρωπαϊσμό της κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν έχουμε στοιχεία στη συλλογή μας από 37 χώρες, από περιφερειακές συλλογές που ξαναμπαίνουν σε άλλο πλαίσιο και έτσι παίρνουν νέο νόημα και γίνονται οι εκπρόσωποι ενός υπερεθνικού ιστορικού φαινομένου. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλαπλές ερμηνείες. Έχουμε για παράδειγμα το θέμα του 1918 Κάποιοι από τους καλλιτέχνες ε, το ερμήνευσαν σύμφωνα με την εθνική ε, ιστορία, την οικογενειακή ιστορία ή και την ιστορία της Ευρώπης. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να συνδυάσουμε το τοπικό, το περιφερειακό και το ευρωπαϊκό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή κληρονομιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο. Όλοι γνωρίζουν τον Πολ Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μποζάρ. Και αναγνωρίζουμε ότι το έργο σου ε, είναι κάτι το οποίο το κάνεις ε, ακάματα για τις τέχνες και τα πολιτιστικά. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε. Βρισκόμαστε μαραθώνιο. Θα σας μιλήσω ως διευθυντής της, του Μποζάρ που έχω την δυνατότητα μέσω της της θέσης να παρακολουθώ τον παλμό και της δημιουργίας στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Την συντήρηση των έργων και την καινοτομία. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν για τη σημασία του πολιτισμού σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο και η, η διακήρυξη της UNESCO μας αναφέρει αυτό και το, από το 2013. Το Ποζάρ έχουμε προσπαθήσει να βρούμε μια σωστή ισορροπία από την ίδρυσή μας το 28 και προσπαθώντας να αναδείξουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες, τους δημιουργούς και τους εκείνου που λαμβάνουν τι αποφάσει. Γνωρίζουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να θεωρείται στατική και ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή, να μιλάει σε όλου. Βεβαίω, η Ευρώπη ανακάλυψε την έννοια τη πολιτιστική κληρονομιά και την απέδωσε στον κόσμο και την έχει διαδώσει με τρόπο ε, πολύ αποτελεσματικό. Όλοι άλλοι όμως βλέπουν διαφορετικά την κληρονομιά. Τη βλέπουν πολύ περισσότερο τυπικά, τοπικά. Λιγότερο κεντρική. Με πιο μικρές πρωτοβουλίες τοπικές. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο άϊλο παρά στο υλικό. βλέπουμε δημιουργούς στην Ευρώπη να προσπαθούν να το κάνουν αυτό, πώς προσπαθούν να δημιουργήσουν μια συλλογή που να όπως ο Μπάνοφ. Στο, συγγνώμη, ο σταθμό στο Βερολίνο. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια πολιτιστική κληρονομιά από τη βάση και όχι κεντρική. Αυτό είναι ουσιαστική σημασία για να δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό ήθο που να απευθύνεται στους Ευρωπαίους πολίτες. Αποκέντρωση λοιπόν, αν θέλετε, της διαχείριση του πολιτισμού και δημιουργία συνεργασιών μεταξύ πολιτιστικών οργανισμών. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Εράσμου. Πολύ περισσότερες συνεργασίες δηλαδή μεταξύ πανεπιστημίων. Κανείς δεν μπορεί να εξερευνήσει την Ευρώπη ή και τον κόσμο εάν δεν συζητήσουμε και το θέμα της αποαπικιοποίησης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό. Εάν δεν το πράξουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό ήθος, σε μια κοινή αντίληψη. Η πολιτιστική κληρονομιά απευθύνεται σε όλους και αφορά και το παρελθόν την, και, το, και το παρόν, το ευρωπαϊκό μοντέλο για το περιβάλλον, για την κοινωνία. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε δημόσιους χώρους στην Ευρώπη, δημόσιους χώρους πολιτισμού, όπου η πολιτισμός και η οικολογία συναντώνται. Το συμπέρασμά σας, λέει η Πρόεδρος, στην διακήρυξη του Νταβός, του 2018 αναφέρεται ότι πρέπει όλο και περισσότερο η σύγχρονη αρχιτεκτονική να συνδεθεί με το σχεδιασμό των πόλεων με μια ολιστική προσέγγιση στην σχέση κοινωνίας και πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κλείνοντας, αφού όλοι ψάχνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή ε, κληρονομιά, τον 21ο αιώνα και η υλική κληρονομιά και η άειλη κληρονομία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερη, με περισσότερη συμμετοχή των πολιτών με σεβασμό της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και της έκφρασης. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Α, δείξαμε μια γενεοδορία προς τον ε, Πολ. Ε, ελπίζω να μην καταχραστούν τις γενεοδορίες μας και οι άλλοι. Τώρα στον τρέχουμε τον Ιωάννης Έμπερτ, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Γκέτε και εκείνος επιτελεί σπουδαίο έργο. Μια, μια καινούργια φάση στην Ευρώπη. Και το έχει τιμηθεί από την Μογκερίνη, από το Κοινοβούλιο, όσον αφορά τον πολιτισμό, τις διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης. Έχουμε την Έουνικ και αυτό στο οποίο βοηθάτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα με εντύπωση, γιατί πραγματικά ό,τι λέμε μεταφράζεται σε 23 λόγες ε, και 23 φορές, ε, είτε αργά είτε γρήγορα, ακούς το δικό σου κοντσέρτο στην ευρωπαϊκή σου γλώσσα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και βλέπω πόσο καλή δουλειά κάνουν οι διερμηνείς. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να μιλήσω σε τόσο πολλές γλώσσες. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα και χρήσιμο για μας γιατί η UNESCO λέει ότι η γλώσσα είναι ο φορέας της άειλης κληρονομιάς μας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι' αυτό να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διεμηνείς. Αυτή τη στιγμή ε, που μιλάμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ε, έχουμε μιλήσει για την ευρωπαϊκή ατζέντα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και συγκεκριμένα υπάρχουν πολλές διαστάσεις του πολιτισμού, αλλά η κοινωνική είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Ακριβώς ε, το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι ένας τρόπος με τον οποίο αποκρισταλώνεται η κοινωνική ε, συνύπαρξη, ε, τα ζητήματα και η ταυτότητα της Ευρώπης. Άνθρωποι από διαφορετικές ε, κοινωνίες και από διάφορες τάξεις έρχονται και στο ΓΚΕΤΕ μέσα στα πλαίσια του UNIC και σε συνεργασία με τους συναδέλφους από την Ευρώπη Πήγαμε ε, στο Μαρόκο και εκεί ε, μιλήσαμε με αρχιτέκτονες ε, για να δούμε πώς εκεί εξελίχθηκε η αρχιτεκτονική κληρονομιά μια Μεδίνα. Έτσι λοιπόν η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι κάτι το οποίο συνήθως διηγούμαστε μέσω από την ευρωπαϊκή ιστορία. Υπάρχουν κάποια έργα ε, της ευρωπαϊκής ιστορίας, ας πούμε, ε, έχουμε κάποια ε, αυτούς τους κύβους με τη ζάχαρη που είναι μια συνεργασία μεταξύ τριών χωρών που αυτό, αυτή η εφεύρεση. Ε, είναι πολλές οι ιστορίες λοιπόν που μπορούμε να διηγηθούμε νέοι οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά ξανά στη ζωή με ένα νέο τρόπο. Σε 20 δευτερόλεπτα μιλάμε για το θέμα της ενσωμάτωσης που για εμάς την ε, Γερμανία είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς έχουμε 800.000 μετανάστες και έχουμε και μια δική μας ταυτότητα που φτιάξαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με την ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Πρέπει λοιπόν τώρα να φέρουμε κοντά μας μια νέα ομάδα ανθρώπων που έχει μεγαλώσει με μια άλλη αφήγηση, με μια άλλη κληρονομιά και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας τα πολιτιστικά ιδρύματα. Είναι μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ταυτότητα της Ευρώπης και η ολοκλήρωση είναι θέματα που για μένα είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτιστική κληρονομιά. Σας ευχαριστώ. Συμφωνούμε 100% λέει η κυρία Σίλβα όσον αφορά την ενσωμάτωση, την κοινωνική και την ε, πρόκληση για την κοινωνία μας. Ξέρετε ότι εμείς στην Ιταλία ε, τι γίνεται, ότι πόσο μόνοι έχουν προσπαθήσει όλα αυτά να τα καλύψουμε και ε, υπάρχουν και έχει πηγαίνει και αυτή η στροφή που έγινε στην Ιταλία για να μην έχουμε τόσο μεγάλη απόσταση από άλλες πιο γενναιόδορε χώρες όπως η Γερμανία. Τέλος πάντων πρώτα η Ευρωπαία και μετά η Ιταλία. Και τώρα ο Σταύρος Μπέος για λόγο, ο οποίος είναι πρόεδρος του φορέα Διάζωμα που αφορά τους ε, καλλιτέχνες, δημιουργούς και τοπικές αρχές. Μιλήστε μας για την συνέργεια, για το τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε χάρη στην καλλιτεχνία. Δύο λεπτά. Θέλω να δεχθείτε μια θερμή καλησπέρα από την Ελλάδα και από τα εκατοντάδες μέλη του διαζώματος. Κυρίες και κύριοι, έχω μπροστά μου ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτό το ψήφισμα, το διάζωμα, το έχει κάνει ειδική έκδοση γιατί είναι μια τομή πραγματικά για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Λες και έχει συγκεντρώσει όλο το βίωμα και όλη την πνευματική παραγωγή της Ευρώπης, των θεσμών της και των πολιτών της. Αυτό το κείμενο έχει στο υπόστρωμά του ένα υπέροχο αξιακό φορτίο που θέλω να το συνοψίσω με δύο μόνο λέξεις. Συνέργειες. Κυρίε και κύριοι, το απόθεμα, το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό, μας χρειάζεται όλους. Όλους. Όχι μόνο τις δομές της δημόσιας, αλλά και τις ιδιωτικές. Και μια αυθεντική συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αυτό το κείμενο έχει και κάτι άλλο που μας απελευθερώνει πνευματικά. Μιλάει επιτέλους για το απόθεμα το περιβαλλοντικό και το πολιτικό ότι είναι κοινό αγαθό. Δεν είναι κρατική περιουσία των κρατών μελών. Είναι περιουσία όλων των πολιτών του κόσμου. Αλλά κάνει και κάτι άλλο. Δέστα και τη στη θεωρία. Μας δίνει και έναν βραχίωνα επιχειρησιακό. Το ΕΣΠΑ 2014-2020. Και μας σωθεί να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού. Τις πολιτιστικές διαδρομές και τα αρχαιολογικά πάρκα. Όλα αυτά που σας περιέγραψα αποτελούν και το γενετικό υλικό και τη μεγάλη αποστολή του διαζώματος, κυρίες και κύριοι. Το διάζωμα λοιπόν δουλεύει στη χώρα μας σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, βλέπω απέναντί μου την κυρία Κονιόρδου και με όλους τους θεσμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι μια συμμαχία δηλαδή που περιλαμβάνει πόλεις, περιφέρειες, την κοινότητα των αρχαιολόγων, διανοούμενους, πολίτες, όλο το τραπεζικό σύστημα, όλα τα ιδρύματα της χώρας. Και έχει και ένα θεσμό καινούριο. Το θεσμό των εταιρικών μελών συμμετέχουν και οι κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας. Ο πρώτος καρπός αυτών των συνεργειών του διαζώματος, που είναι και ο πρώτος καρπός αυτού του ψηφίσματος πανευρωπαϊκά, είναι η πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Υπήρου, την οποία θα δώσουμε στις 20 του Οκτώβρη, μαζί με την Υπουργό, την κυρία Κονιόρδου, στην τουριστική οικονομία, στην παγκόσμια τουριστική οικονομία και θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλα τέτοια προϊόντα. Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω έκκληση. Να μην είναι σήμερα μια μέρα πανηγυρική, αλλά να είναι μια μέρα αγωνίας και μια μέρα υπόσχεσης ότι αυτή την παραγωγή μας θα την υπερασπιστούμε. Και θα φέρουμε τα μνημεία, το απόθυμα, δηλαδή το περιβαλλοντικό και το πολιτικό της Ευρώπης, στο κέντρο της ζωής, στο κέντρο της οικονομίας και στο κέντρο της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα λίγο να διασφαλίσω ότι εφόσον είμαστε και στην Επιτροπή... Είναι τελικά οριζόντιο αυτό το θέμα και έτσι και το βλέπουμε και εμείς. Θεωρούμε ότι θα πρέπει ο πολιτισμός να πάει παντού, στην έρευνα, στα ψηφιακά, στα διαρθωτικά, και επίσης τις ε, πολιτικές όπως της καινοτομία. Όλα αυτά θα πρέπει να εμπλέκονται τα κρατή, μέλη, όλη, όλη η καλλιτεχνική κοινότητα να υποδείξει αυτά και τα ε, ψηφιακά όπως είπα. Και ε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε αυτό το οποίο λέγαμε, να έχουμε δηλαδή ερώτα απαντήσει γιατί έχουμε τώρα τα άλλα πάνελ, αλλά έχουμε μία-μία εξαίρεση για τις δίθια στην αρχή κάποιος που κάτι μπορεί να μας πει. Πρόκειται για την πραγματικότητα. Θα δώσω το λόγο μόνο σε εκείνον. Και μετά έχουμε την ε, μουσική. Έχουμε τα παιδιά τόση ώρα εδώ, να σεβαστούμε την αναμονή τους και κατόπιν έχουμε το επόμενο πάνελ. Και τώρα... Future for Religious Heritage. Το μέλλον της θρησκευτική κληρονομιάς η Λίλιαν που από την αρχή είχε ζητήσει τον λόγο και θα τη τον δώσω. I am here, I'm here. Ε, εδώ. Yes, yes, yes, I'm here. Σας εδώ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μάλιστα τώρα σας είδα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με το οποίο ασχολείστε. Έχετε μόνο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα. Μας δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθούμε. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ και να αναδείξουμε την πρωτοβουλία μας. Θέλω να ζητήσω από όλους σας, όλοι όσοι είστε εραστές του πολιτισμού να συμμετάσχετε σε, αυτόν τον, σε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε για την πολιτική μας κληρονομιά. Πρόκειται εδώ για ένα ε, μπαούλο με θησαυρό που πρέπει να ανοίξουμε. Πρόκειται για κληροδότημα. Αυτό αφορά τα πάντα, ακόμα και μια ζωγραφιά. Να Κοιτάξτε αυτό το κουτί τώρα που σηκώνει η ομιλήτρια. Ε, στην είσοδο θα βρείτε ε, τα σχετικά φυλάδια για το τι χρειάζεται να γίνει. Σα ευχαριστούμε για την πολυμορφία στην Ευρώπη. Όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, όλοι είμαστε μια ορχήστρα. Ο καθένα παίζει το δικό του σκοπό, αλλά τελικά, όπω είπε και ο Ιταλός μαέστρος, έτσι θα πρέπει να δουλεύει η Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε εμεί. Είναι αυτή σα η πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική είναι ένα από τα υπερσυνοριακά, διασυνοριακά ε, προγράμματα της ε, Ευρώπης. Πολύ όμορφη και η άκρο συμβολική πρωτοβουλία σας. Οπότε τώρα, κοιτάξτε, έχουμε ταυτόχρονα αυτό το βίντεο που εξηγεί τι είναι το Europa in Canto. Είναι ε, κάτι καινοτόμο αφορά 50.000 παιδιά 3 έως 14 και ε, που σπουδάζουν την ε, όπερα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα του πώς κανείς μπορεί να σπουδάσει μουσική. Ε, παίζουν πολλές όπερες κάθε χρόνο σε πάρα πολύ σημαντικά ε, κτίρια όπως ε, στην ε, Ρώμη, Νάπολη, Τρεβίζο και πρόκειται για μια, τροπο, μια πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί στο να διαδοθεί η όπερα. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και τους ενήλικες. Πρόκειται για χιλιάδες γονέων, δασκάλων που έχουν εμπλακεί. Και όταν βλέπει σε μια Ιταλική όπερα, σε ένα Ιταλικό θέατρο να παίζεται μια όπερα, έχουμε δύο-τρεις ε, παραστάσεις κάθε μέρα και πάντα είναι το θέατρο γεμάτο. Στα πλαίσια και του Ευρώπα Όπερα, ένα χειροκρότημα για τον διευθυντή ε, τον Τζερμάνο, Δεν θυμάμαι. Πάλι τόσο μου δεν έχει σημασία. Και το πιο σημαντικό που να θυμόμαστε είναι ότι έτσι πλησιάζουν, εξοικειώνονται τα παιδιά. Ε, το κάνουν σαν παιχνίδι. Γιατί το δράμα, το μελόδραμα και αυτό είναι κομμάτι του πολιτισμού και άρα έτσι ε, βλέπουμε με φρέσκια ματιά την όπερα. Έχουμε εδώ κάποιους ε, γονείς. Και ε, υπάρχει και CD. Και έτσι οι γονείς κάνουν καραόκε. Συνοδεύουν τα παιδιά και τραγουδούν την ΑΕΔ με αυτόν τον τρόπο. Να πώς γίνεται η εκπαίδευση και πώς μεταδίδεται η κουλτούρα και ο πολιτισμός από τη μια γενιά στην άλλη. Grazie. Just... Κυρία Κώστα, ευχαριστώ. Θέλω το εξή να σας πω. Βάλτε τα ακουστικά σας. Είναι δύο σχολεία από την Ρώμη. Και έχουμε και ένα σχολείο, μια σχολή τέλο πάντων που προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια εμπειρία που ενώνει, γιατί εδώ έχουμε και κάποια παιδιά τα οποία είναι κοφάλων. Μάλλον έχουν κοφόντα τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ σημαντική γι' αυτό το λόγο αυτή η εμπειρία.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 Thank you so much. Η κυρία Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν φανταστική αυτή η μπράβο στους νεαρούς μουσικούς, στους νεαρούς τραγουδιστές, τον διευθυντή σε όλους σας. Και τώρα, με τη μουσική ολοκληρώσαμε αυτό το πάνελ και θα δώσουμε τη θέση μας στο επόμενο πάνελ. Αυτό το οποίο θα προεδρεύσει ο Μητσέα Διακόνου. Ο εισηγητής μας για το έτος πολιτικής κληρονομιάς του Κοινοβουλίου. Μίρτσε, έχεις το λόγο.

work. Yeah. Please sit down. Παρακαλώ. Παρακαλώ καθίστε. Thank you. Good afternoon. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Since we are here... Επειδή σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να συζητήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η γλώσσα είναι κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επίσης, η δυνατότητα να ακούσε την κάθε εθνική γλώσσα είναι η ίστατη έκφραση της ε, ποικιλομορφίας. Και επειδή το να μιλάς μια γλώσσα είναι μορφή πολιτιστικής κληρονομιάς και η στη μορφή πατριωτισμού, θα μου επιτρέψετε να ε, μιλήσω στη γλώσσα μου τα ρουμάνικα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο πως αυτή η διάσκεψη αποτελεί μία γιορτή, ένα πανηγύρι. Έχουμε ιδικούς προσκεκλημένους και όλοι μας, από όπου και αν προερχόμαστε, πρέπει να αποτίσουμε πόρο τιμής σε αυτό που μας ορίζει, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών και αλληλεγγύης από την Επιτροπή ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Πολιτισμό, σύσσωμη την Επιτροπή και να την ευχαριστήσω. Είχαμε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ε, σταθερή. Ε, ο βασικός μου στόχος λοιπόν ήταν αυτός ο εορτασμός ε, να γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεκτός και να γίνει αποδεκτός και σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ήταν δύσκολο αλλά έγινε, έγινε πραγματικότητα καταφέραμε γιατί η πολιτιστική κληρονομιά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού ιδεώδους που πρέπει να φέρουμε ε, στους λαούς ε, της Ευρώπης. Πρέπει αυτό το έργο να μην έχει τέλος. Ας πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Καλό τον Τερίμαξ. Σεφ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, ε, αγαπητοί Ευρωπαίοι φίλοι. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί είμαι από μία γειτονιά του Ανατολικού Παρισιού όπου δεν έχω συχνά την ευκαιρία να μιλώ σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Ε, ε, μιλάμε πλέον σήμερα για την πολιτιστική κληρονομιά. Επειδή από νωρί ε, στο σχολείο κατάφερα να μάθω ότι υπάρχει δυνατότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης για να μπορέσει κανείς ε, να απελευθερώσει τις δυνάμεις του, έγινα ζαχαροπλάστης και μέσα από αυτό μπορώ να γιορτάσω την κληρονομιά. Την κληρονομιά που είναι αυτό που μας άφησαν οι πατέρες μας. Κάτι σημαντικό, ένας διαφωτισμός, ε, είναι αυτό που μας δείχνει το δρόμο. Έτσι λοιπόν, ε, μέσα από αυτό είδαμε πως δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της παράδοσης και της καινοτομίας. Αυτό που μετράει είναι μεταφορά της γνώσης. Αυτό έμαθα λοιπόν από την καριέρα μου ε, και από την ιδέα της ε, κληρονομιάς ποια θα είναι η γαστρονομία στα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ε, ευρωπαϊκό ε, κοινό εγκέφαλο, ο οποίος ε, θα εργαστεί για την βιοτεχνία, για τις επιστήμες, για τη γεωργία, για να διασφαλίσουμε καλά προϊόντα, για να διασφαλίσουμε σωστές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και ποιο είναι το όπλο, είναι ακριβώς η τέχνη μου. Έτσι λοιπόν Πάμε από το πολύ μικρό στο, στο απείρος μικρό στο απείρος μεγάλο. Φτιάχνουμε μια ιδέα η οποία γίνεται ένα πιάτο και στην ουσία επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την ίδια ιδέα ε, που, για την οποία μιλάμε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του ωραίου και του χρήσιμου. Η Ευρώπη έχει την εξή δύναμη, την ποικιλομορφία της. Είμαστε όλοι μαζί και ο ένας με τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Euh, και εμεί ευχαριστούμε, κυρία Ματίλντα Κοτέ, φωτογράφου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κύριε και κύριοι Υπουργοί, κύριε και κύριοι Επίτροποι, κύριε και κύριοι αγαπητοί φίλοι Ευρωπαίοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Αντώνιο Ταγιάννη που μου έδωσε την ευκαιρία να εκφράσω πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη τη κληρονομιά μας, τη Ευρωπαϊκή δημιουργία των Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Αισθάνομαι βαθιά Ευρώπη. Έχω γεννηθεί στις Βρυξέλλες, ζω στο Παρίσι, έχω γεννηθεί εδώ στο Ιξέλ. Ε, τότε ήμουν ήδη ε, πεπισμένη Ευρωπαία από νωρίς ε, τότε φάμε. Τρώμε χάμπουργκερ, κασουλέ, κουσκούς ε, τρώγαμε τα πάντα, όλα τα φαγητά της Ευρώπης Αισθάνομαι βαθιά Ευρωπαία στα γονίδια μου. όπως είμαι και καλλιτέχνη. Αισθάνομαι Ευρωπαία καλλιτέχνη. Είμαι περισσότερο μια γυναίκα της εικόνας, ε, όχι τόσο ε, των λέξεων. Έφτιαξα λοιπόν μια ταινία που εκφράζει τη δουλειά μου, τις πεπιθήσεις μου, τη δημιουργία μου με τη φωτογραφία. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte. J'ai été reporter pendant 10 ans. Ανέκαθεν ε, ήμουν φωτογράφο, ήμουν ρεπόρτερ για 10 χρόνια. Ζούσα στο Λο Άντζελε που εργαζόμουν για γαλλικά περιοδικά. Έχω εργαστεί για διάφορα θέματα. Στην περιοχή του Λο Άντζελε. όταν ε, γύρισα στη Γαλλία, Δούλεψα για τον Αλάν Κάσε. έψαξε κάποιο φωτογράφο που να μην είχε ασχοληθεί με τη γαστρονομία. Εγώ προσέγγισα τα ζητήματα αναδεικνύοντας ε, την υφή τους, ε, την αξία τους. Αυτό μου επέτρεψε να δούμε με ένα νέο τρόπο. Για μένα ένα αυγό Σολομού μοιάζει με έναν πλανήτη. Ότι παράγει η γη μοιάζει με τη γη την ίδια. Έπαιξα με αυτό το πάρα πολύ μικρό και το πάρα πολύ μεγάλο με συγκεκριμένα πράγματα, με υλικά που χρησιμοποιούμε στις συνταγές. Ε, ε, δημιουργώ κάτι αφηρημένο, εικόνες που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Και αναδεικνύοντας ε, την ύλη, την προστατεύω. Μου επέτρεψε να βγάλω δηλαδή τη μαγειρική από τη μαγειρική. Διηγήθηκα ιστορίες σε ένα πλαίσιο συναισθηματικό δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο, σε ένα βιβλίο ή σε ένα χώρο, με μια διαφορετική διαδικασία, μια διαφορετική προσέγγιση που αποδεικνύει πόσο ξεχωριστό είναι. Δημιουργεί ένα διαφορετικό συνέστημα. Το 2001, όταν έφτασα στον κόσμο της γαστρονομίας, ε, γεννιόταν ένα νέο κίνημα στην Ευρώπη. Η μοριακή γαστρονομία ο Φεράν Αντριάν στην Ισπανία και ο Τιχέρη Μάρξε στη Γαλλία και ο στον Κομεντάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο την εισήγαγαν και παράλληλα με αυτή την εξέλιξη στη μαγειρική παγκοσμίω ε, γινόταν μια επανάσταση στον κόσμο της φωτογραφία με τι πρώτε ψηφιακέ μηχανέ. Εγώ πρέπει να πω ότι υποστηρίζω την πρόοδο και αμέσως ε, υιοθέτησα αυτή την τεχνολογική πρόοδο που εκδημοκράτησε τη φωτογραφία, βοήθησε την κοινοποίηση ταχύτερα των φωτογραφιών και των πληροφοριών μέσω της εικόνας. Λίγο νωρίτερα, το 1994, χάρη στην Alliance Française, οργάνωσα μία κινητή έκθεση που έδειξε ε, τη δουλειά μου στις μεγαλύτερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκτοτε δεν κατάφερα να ξαναταξιδέψω τις εικόνες μου, που τόσο ασχολούνται με ένα οικονομικό ε, θέμα, το φαγητό είμαι ακτιβίστρια ως φωτογράφος, υπερασπίζομαι τη γη. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων. Ε, λόγω έλλειψης μέσων, έλλειψης υποστήριξης, έλλειψης ενός ε, ε, ισχυρού ευρωπαϊκού οργανισμού που να με βοηθήσει μέσω του διαδικτύου, του Instagram, κατάφερα όπως πολλοί καλλιτέχνες να διαδώσω την τέχνη μου. και έτσι μπορούμε να κρατήσουμε με την ψηφιακή φωτογραφία ένα μεγάλο ποσοστό των φωτογραφιών μας σε μικρές συσκευές, αλλά εγώ έγινα φωτογράφος λόγω του ε, πρωτόγνωρου συναισθήματος που ένιωσα την πρώτη φορά που είδα το φυσικό φως να φωτίζει ένα τεράστιο έργο αφοσιωμένο σε αυτήν. Γι' αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα δημιουργού στην Ευρώπη και πέραν τη Ευρώπη. Είναι κρίσιμη σημασία σε ευρωπαϊκέ χώρε να ενωθούν, να συγκεντρώσουν τα μέσα του ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε καλλιτέχνε και δημιουργού να εκθέτουν στην Ευρώπη και πέρα των σύνορων μα. Γι' αυτό για μένα ελπίζω ότι η Ευρώπη μας θα συνεχίσει να υπάρχει. Ε, και τώρα η κυρία Μάριο Νάκερμαν, Γενική Διευθύντρια των ε, Κρατικών Γενικών Συλλογών Έργων Τέχνης στη Δρέσδη. Τα ευρωπαϊκά ε, πολιτιστικά ιδρύματα ε, υφίστανται μεγάλες πιέσεις και μεγάλες απειλές για τη δημιουργία. Θα πρέπει να λάβουμε μια θέση και να σπάσουμε τα ταμπού και τη διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στα μουσεία και την καθημερινή ζωή, την υψηλή και τη χαμηλή τέχνη. Θα πρέπει κανείς να βιώνει τις ε, ύλες, ε, τα υλικά, τη χειροτεχνία για να συμφιλειωθεί ε, ο δημιουργός με εκείνο που απολαμβάνει το έργο τέχνης. Η γνώση και η εμπειρία είναι βίωμα, δεν είναι απλώς θεωρητική γνώση ο καθένας μπορεί να γίνει παραγωγός και δημιουργός της πραγματικότητας και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Το 1560 ιδρύθηκε ε, το μουσείο μας στη Σαξονία και έκτοτε παράγει τα μέσα και τις επιστημονικές ε, δυνατότητες ε, που έχουμε στη συλλογή μας. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερη χαρά ε, να έχουμε πάρα πολύ πολύτιμα ε, ε, έργα που επιβίωσαν στην Ανατολική Γερμανία, ιδιαίτερα στη Σαξονία. Έχουμε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 294 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι το 8% της παραγωγής στην ε, Ανατολική Γερμανία, επειδή δεν υπήρχαν καταναλωτικά αγαθά, η χειροτεχνία είχε πάρα πολύ ψηλή θέση και προστατευόταν. Σήμερα όμως ε, το dumping, οι χαμηλές τιμές και ε, οι ανταγωνιστικές εταιρείες πολυεθνικές πιέζουν προς τα κάτω την χειροτεχνία και την παραγωγή. Μπορούμε να εξυγχρονίσουμε ε, και τη χειροτεχνία και να ανοίξουμε προοπτικές για το μέλλον, ας πούμε. Για την ανοικοδόμηση ε, του ανακτόρου στη Δρέστη ε, χρησιμοποιήθηκαν και ανακτήθηκαν παλιές τεχνικές, παλιά χειροτεχνία και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας. Τα μουσεία είναι και μνημή αλλά και ενεργοποίηση της γνώσης. Το θέμα δεν είναι να επιβάλλεις τη μνήμη αλλά να δημιουργείς μνήμη η διεθνής ε, η διεθνής νοοτροπία ε, αποκτά νέες δεξιότητες, νέες ε, δυνατότητες και αυτό φαίνεται όλο και περισσότερο στη Δρέσδη. Από που ξεκίνησε η ακροδεξιά λαϊκιστική ρητορική. Είχαμε και την ομάδα καλλιτεχνών την Μπρούκε στο 19ο αιώνα, γέφυρα, και τώρα έχουμε πρόοδου στα φωτοβολταϊκά και σε άλλες τεχνολογίες. θα πρέπει να σπάσει επίσης ε, αυτός ο διχασμός ανάμεσα σε μεγάλου πόλεις και ε, ε, περιοχές της υπαίθρου. Αυτό θα δημιουργήσει πλούτο, θα φέρει πιο κοντά διαφόρους ανθρώπους από τη Γερμανία, από την Ευρώπη που δημιουργούν ταυτότητα ευρωπαϊκή. Θα πρέπει να σταματήσει η ιεραρχική αυτή αντίληψη ε, ότι άλλο η τέχνη, άλλο η χειροτεχνία. Αυτό μπορεί να έρθει από τις περιφέρειες, ε, από κάτω προς τα πάνω και να επαναφέρει ε, εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη χειροτεχνία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να τα προάγουμε. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να πω το μαγικό. Δύο-τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με και μένα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε καλά αυτή τη συνάντηση. Τώρα το λόγο έχει η Φρανς Δεμαρέ που είναι η ευθύντρια προγραμμάτων και ανάπτυξης του Διεθνού Συμβουλίου Μουσείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε σήμερα ότι ο πολιτισμό είναι αυτό που μα κάνει ανθρώπου, είναι αυτό που μα διακρίνει από τα άλλα είδη. Θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι δεν είναι ανάγκη να πείσουμε κανέναν για τη σημασία που έχει η προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά. Όμω, δεν είναι αλήθεια. Πρέπει. Γιατί σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά περισσότερο από ποτέ, είτε πρόκειται για ακίνητη, είτε πρόκειται για ηλική, για άειλη. Δέχεται επιθέσεις, λαιλασίε, καταστροφές, επίτηδες ή όχι επίτηδες, εξαιτία τη αμέλεια, εξαιτία ε, λαθρεμπορίου παντό. είδου. Όμως, ακριβώς αυτό είναι, είπαμε, που μας διακρίνει από τα άλλα είδη. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φροντίζει για την προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά για την πρόθεσή τη, για την ποικιλομορφία της και για το ρόλο που έχει να παίξει στην κοινωνία. Ελπίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι δεν προστατεύουμε μόνο αντικείμενα όταν προστατεύουμε την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά μαρτυρίε, μαρτυρίε του παρελθόντος, πυλώνε τη ανάπτυξή μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια το έχει καταλάβει αυτό και εγώ το έχω καταλάβει αυτό από πρώτο χέρι όταν η Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η πρώτη που πίστεψε στο διεθνέ Παρατηρητήριο για την αποφυγή λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών που δημιουργήθηκε το 2012. Κάνω λοιπόν έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να βοηθήσουν τι συνέργειε, τη συμπληρωματικότητα, τη συνεργασία με δύο λόγια. Κανεί από μόνο του, είτε πρόκειται για θεσμό είτε πρόκειται για χώρα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του αυτό το πρόβλημα. Η προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά είναι το έργο ε, πάνω στο οποίο πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε, να φροντίσουμε να βρούμε βιώσιμε αποτελεσματικέ λύσει. Όταν ε, ξεκίνησα να προτείνω τον κατάλογο με την πολιτιστική κληρονομιά που κινδυνεύει, διαπίστωσα ότι αυτό θεωρείται απλώς ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τα πολιτιστικά αντικείμενα. Μόνο μια χούφτα ανθρώπων ε, νοιάζεται πραγματικά τα πράγματα βέβαια σιγά σιγά αλλάζουν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ξεκάθαρο ότι εδώ διακυδεύεται κάτι πολύ περισσότερο γιατί υπάρχει μαζική καταστροφή, λαιλασίες, απειλές που ακυρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ιστορίας μας και την κοιτίδα του πολιτισμού και αλλού στον κόσμο. Άρα κατέληξε να είναι θέμα όχι μόνο ανάπτυξης, είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα επιβίωσης. Η προστασία του πολιτισμού συνδέεται τώρα και με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλοι είμαστε αλληλένδετοι μεταξύ μας, Οπότε, όποιοι και είναι οι λόγοι, όποια και τα επιχειρήματα που μπορεί να έχει κανείς για να θέλει να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά, το βέβαιο είναι ότι προστατεύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, προστατεύουμε τις ευκαιρίε μας για ένα καλό μέλλον στις χώρες μας αλλά και στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμαρέ. Το Ρακάουντ Ροντόλφο Ντελόσο Κορσβάρεμ, πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ιστορικών Οίκων. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη. Το έχω κάνει πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλά θέλω για άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά μας άνοιξε τις θύρες του δικού τους οικού, που είναι όμως και δικό μας και που πολύ αγαπάμε. Ήρθαμε εδώ, έχουμε πολλούς φίλους θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και του ανθρώπου που βοήθησαν ώστε το 2018 να καταστεί το έτο τη πολιτιστική κληρονομιάς. Έχω φίλου επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού. Αλλά και μεταξύ των επικεφαλή κρατών και κυβερνήσεων έχουμε φίλου, Γιατί από μόνη τη Επιτροπή, χωρί το Συμβούλιο, δεν θα μπορούσε να έχει πετύχει το ε, έτο αυτό πολιτισμού το 2018. Θέλω επίση να ευχαριστήσω πάρα πολύ και φίλους από την Ευρώπα Νόστρα και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πολιτισμού. Πρόκειται για 40 ενώσεις συλλόγους, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα λοιπόν είναι ιστορική σημασία αυτή τη στιγμή που είμαστε όλοι μαζί, ανθίζουμε. Είμαστε σε ένα δέντρο που έχουμε ρίζες, έχουμε κορμό, έχουμε τα κλαδιά, έχουμε τα φύλλα, έχουμε το άρωμα. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει από τις ρίζες και τον κορμό. Ε, είναι λιγάκι σαν μια λυσίδα με κρίκους. Μερικές φορές υπάρχουν και αδύναμοι κρίκοι, γιατί αυτή η ιστορική οίκη μερικές φορές είναι απομακρυσμένη από τα πάντα. Είναι ψυχροί, κλειστοί, κάνουν επισκευέ και αυτοί που τους διαθέτουν νομίζουν ότι είναι πλούσιοι, αλλά δεν είναι απαραίτητα πλούσιοι σήμερα. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Και γι' αυτό είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ. Τι θα μπορούσα να σας πω ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι πιο σημαντικός ως έσοδα για τους πολιτικούς από το έτος πολιτισμού, από την αυτοκινητοβιομηχανία, το ξέρετε αυτό, αλλά και από τη χημική βιομηχανία. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να κλαίμε. Αντίθετα, πρέπει να είμαστε ευτυχεί, να χειρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ και που έχουμε ένα μικρόφωνο μπροστά μα για να μπορούμε αυτό να το πούμε, να το φωνάξουμε και να το ακούσουν όλοι. Τέλος, θέλω να σας ε, μιλήσω και για κάτι για το οποίο δεν μιλάμε συχνά στους πολιτικούς χώρους. Για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έξω από τις μεγάλες πόλεις, στην Ήπεθρο. Να σας μιλήσω για τους ανθρώπους που δεν βλέπουμε, που δεν περιλαμβάνονται στο τοπίο. Έχουν και αυτή μεγάλη σημασία. Και τέλος, πρέπει να ξέρετε ότι εμεί δεν θέλουμε να ευχαριστήσουμε μόνο αυτού που έρχονται και επισκέπτονται τα μουσεία, του ιστορικού οίκου κτλ., αλλά και τι πεταλούδε, τι μέλισσε, τα πουλάκια, γιατί είμαστε σε πάρκα, σε κήπου που αποτελούν το κλαμπ Μεντιτερανέ όλων αυτών των ζωντανών που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε κι εμεί. Οπότε, όταν λέτε κρίμα για τις πέτρες και τα τούβλα, σκεφτείτε και όλη αυτή την όμορφη φύση που έχουμε γύρω μας και που πρέπει να φροντίσουμε να διασώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ολύμπια Μπράτσι Μερμορό, ε, καλλιτεχνική διευθύντρια στην Ένωση Πικολοτέατρο Μάργα Σεργάντη. Κύριε Πρόεδρε, ομιλητέ, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που με καλέσατε να σα παρουσιάσω την πολιτιστική κληρονομιά που κληρονόμησα από τη γιαγιά μου, τη Μάργα Σεργάντη, και πώ προτίθεμαι να προωθήσω το πολιτιστικό τη έργο, το οποίο αποτελεί ένα στο κομμάτι του Νεδρυθέντο Πίκολο Θεάτρο Μάργκα Σεργάρντι. Η κληρονομιά απτή και άειλη, σύμφωνα με την ταξινόμηση τη UNESCO, είναι ένα κληροδότημα από το παρελθόν, κάτι με το οποίο ζούμε σήμερα και το οποίο θα δώσουμε στι επόμενε γενιέ. Το μικρό θέατρο αυτό δημιουργήθηκε από τη Μάργκα Σεργάρτη Μάρμόρο. Έφερε στη Σιένα και στο Παλάτσο Σεργάρτη τη θεατρική γνώση που απόκτησε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ήταν νέα κοπέλα στους κήπους της Βίλα Κατινιάνο έξω από τη Σιένα, εκεί που μεγάλωσε όπου έδινε διάφορες ρουστικ παραστάσεις και με αυτόν τον τρόπο δίδαξε στα παιδιά των ε, το ντόπιον πώς να παίζουν στο θέατρο και διεύθυνε έργα για τα παιδιά. Στι αρχέ του 50 η Μάργα μεταφέρθηκε στο Παλάτσο Σεργκάρτη και ίδρυσε το μικρό θέατρο Σιένα δημιουργώντας ε, ένα θέατρο Εκατοθέσεων θέσεων ε, που λειτουργούσε απόλυτα και ήταν απόλυτα εξοπλισμένο στο... και όπου δημιουργήθηκε ένα κέντρο εκπαίδευσης και κέντρο θεατρικών παραγωγών. Αυτές οι δύο παράλληλες δραστηριότητες του μικρού θεάτρου ε, δοκίμησαν για περίπου μισό αιώνα. Σήμερα είναι δική μου επιθυμία να ακολουθήσω τα βήματά της. Εγώ ως καλλιτεχνική διευθύντρια με τον Τζαραρντο Μανφέη στη νέα ένωση που έχουμε δημιουργήσει, ε, σκοπός της οποίας είναι μεταξύ άλλων ένα θέατρο, ε, ένα κέντρο ε, τεχνών σαν αυτό, να προωθήσει την ηλική και άειλη η πολιτιστική μας κληρονομιά, διαδίδοντας τις παραδοσιακές δραστηριότητες διδασκαλίας, δημιουργώντας συνεργασίες σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και δημιουργώντας νέα ε, νέες σύγχρονες ε, καινοτόμες ε, θεατρικές παραγωγές. Πριν κλείσω, ήθελα να σας πω ότι είδα το όραμά μου να αντικατοπτρίζεται στα λόγια δύο επιφανών ανθρώπων. Ο καθηγητής Κλάμορ λέει ότι η έρευνα, όπως κάθε διαδικασία ανάπτυξης, αποτελεί ε, ένα, μια πολιτιστική συνιστόσα για να φέρει την αλλαγή. Οι τέχνε λοιπόν, ο πολιτισμός μπορούν να προωθηθούν ως σημαντική συνιστόσα της ανάπτυξης και της επιτυχίας της. Η ίδια η UNESCO πρόσφατα προώθησε την ιδέα των δημιουργικών ε, τομέων ως ε, τρόπου ανάπτυξη. Αυτό σκοπεύει να γίνει το Πίκολο Θέατρο Μάργα Σεργάρντι, ένας τομέας δημιουργίας. Στο μέλλον το ανθρώπινο, το κοινωνικό και το δημιουργικό κεφάλαιο είναι αυτό που θα επιτυγχάνει τα περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο η τέχνη ο πολιτισμός είναι κάτι αναγκαίο. Καμία άλλη προσέγγιση δεν έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στο να άρει τα εμπόδια, να συνδέει τις πολιτιστικέ μας διαφορές ε, και να θέτει από κοινού τι κοινέ μας αξίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κοινή ηγεσία, ώστε να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη ως κάτι αναγκαίο, όχι ως κάτι απλά όμορφο. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μαρία Τερέζα Σκετίνο, ε, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Τάζο εγώ τελαντικήτε. Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή να ανοίξουμε το μικρόφωνο σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να παίρνω το λόγο εδώ στο ημικύκλιο, πρώτον και κυρίως ως εκπρόσωπος ε, της ε, γαλλικής και ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας που ανέκαθεν ε, μελετούσε και ε, μετέφερε ε, την πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα της αρχαιότητας. Επίσης είμαι συγγραμματέας των État Généraux de l'Antiquité, που είναι ένα δίκτυο ενώσεων με το όνομα Antiquité Avenir, αρχαιότητα και μέλλον. Τελευταία φορά συνεδρίασε στη Σορβόνη 8 και 9 Ιουνίου υπό την αιγίδα μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική αξία της κληρονομιάς που η αρχαία Μεσόγειος μας έχει κληροδοτήσει. Πρώτα απ' όλα είναι μια άειλη κληρονομιά, όπως οι γνώσεις που αφορούν τη φιλοσοφία, τις γλώσσες, ε, τα νομικά και τα επιστημονικά ζητήματα. Αλλά υπάρχει και η υλική κληρονομιά, όπως είναι τα ιστορικά κτίρια και οι αρχαιολογικοί χώροι. Αυτή η κληρονομιά εμοδοτεί ε, την σύγχρονη μας ε, πολιτιστική πραγματικότητα και ε, είναι και το τοπίο των πόλεων μας. Προτείνω να δημιουργηθεί ένα, μια διαδρομή που να βασίζεται στην αρχαιότητα, στη Μεσόγειο, υπό την αιγύδα της Ευρώπης και της UNESCO. Να είναι λοιπόν μια πολιτιστική κληρονομιά που να συνδέεται με την ειρήνη και θα πρέπει να ενώσει τις διάφορες όχθες της Μεσογείου. Και όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά να χρησιμοποιηθεί και σε ένα διπλωματικό εργαλείο. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που θα δώσετε και θα δείξετε για την πρότασή μας. Παραμένω στη διάθεσή σας για να το συζητήσουμε και ενδεχομένως να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci. Σας ευχαριστούμε. Τώρα, Σνέσκα Μιχαηλοβίτς από την Ευρώπα Νόστρα. Γενική Γραμματέας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουν υποθεί τα πάντα. Εγώ θέλω να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα ευτυχή και πολύ περήφανη, γιατί όλοι ζούμε ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ότι καθόμαστε εδώ, σε αυτή την αίθουσα τη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Είμαστε στα μέσα του πολιτισμικού αυτού έτους και το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Και πώς έγινε αυτό, γιατί συνεργαστήκαμε όλοι με ενθουσιασμό και βάλαμε όλοι πολύ ενέργεια σε αυτό το όνειρο. Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει και η Ευρώπη. Και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Να πω ότι χρειαζόμαστε συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις, συμμαχίες στην Ευρώπη. Και γι' αυτό ο συνάδελφος Ρόντολφο Ντελός Κοσβάρμι το είπε. Όταν αρχίσαμε το 2011 δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το 2018 θα συγκεντρωνόμασταν εδώ πέρα για να γιορτάσουμε το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Ελπίζω να έχουμε ακόμα κάποιου ευρωβουλευτέ εδώ στην αίθουσα, να έχουν παραμείνει. Πάντω θα έλεγα ότι αυτή η συμμαχία πολιτισμών θα προχωρήσει μέσα από επιτροπές, μέσα από πολιτικά κόμματα και θα προωθηθεί ακόμα περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί πράγματι είμαστε δυνατοί αν είμαστε ενωμένοι. Επιτρέψτε μου να το πω και στη δικιά μου γλώσσα, λέει ομιλήτρια, στα σερβικά. Θα ήθελα να έχει ακουστεί και αυτό εδώ. Το όνειρο λοιπόν γίνεται πραγματικότητα. Ακούσαμε πριν όπερα εδώ, στην αίθουσα Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορχήστρα, τα ακούσαμε. Ο Πλάστο Ντομίκο δυστυχώ είπε ότι λυπάται πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά υποσχέθηκε ότι την επόμενη φορά θα έρθει. Γιατί και γι' αυτόν θα είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Και αυτό ακριβώ είναι το σημαντικό στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ότι είχαμε όπερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν είχαμε περισσότερη μουσική και περισσότερη ερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των πολιτών, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο την Ευρώπη. Ακούσατε πάρα πολλά για την έκκληση του Βερολίνου που προωθήσαμε, υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα Υπάρχει. Να, εδώ έχω ένα αντίγραφο και υπάρχουν και πολλά αντίγραφα. Εδώ αν θέλει κανεί, είμαι γεμάτη από αυτό, ποιος θέλει να έρθει να το υπογράψει, έρθει να με δει. Και θέλω σας παρακαλώ να πω και κάτι τελευταίο στο μισό λεπτό που μου μένει. Τώρα πρέπει να δράσουμε, μαζί πρέπει να δράσουμε, να αλλάξουμε την απόχρωση, να αλλάξουμε τη ρητορική, να αλλάξουμε την οτροπία μας για το μέλλον της Ευρώπης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Big Bang πνεύματος στην Ευρώπη. Η Λίνα Κονιόρδου μίλησε πριν για αυτό το Big Bang που έγινε στην Αθήνα πριν από 1500 χρόνια. Μπορεί να ξαναγίνει και όχι μόνο στην ε, Αθήνα, στις Βρυξέλλες ή σε μια μοναδική πόλη, όχι, σε όλες πρέπει να επαναληφθεί το παράδειγμα αυτό. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τον πολιτισμό και από την πολιτιστική μας ευρωπαϊκή κληρονομιά. Σας ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητή Σνέσκα, να ξέρεις ότι εδώ στο κοινοβούλιο άλλοι τραγουδούν, άλλοι δεν τραγουδούν καλά. Ο κύριος Φαράτζε είναι γνωστός τραγουδιστής εδώ, αλλά τραγουδάει λίγο φάλτσα. Δεν το ξέρετε. Okay. Ε, λοιπόν, ε, περνάμε στη συζήτηση. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε σύντομες ερωτήσεις ε, συνοπτικά. Όχι πολλές και με μεγάλη ακρίβεια γιατί θα ήθελα να μπορέσουμε να καλύψουμε τουλάχιστον 20 λεπτά καθυστέρηση που έχουμε σωρεύσει λόγω των μεγάλων ομιλιών που είχαμε στην αρχή της ημέρας. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Στέφανο Μπονφιά. Έρχομαι από την Oxford Sustainable Development, μια επιχείρηση που λειτουργεί εδώ και 15 χρόνια στην Oxford, στο Ρωμανό Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε κάτι που σχετίζεται με τη Μεσόγειο και θέλουμε να το συζητήσουμε περαιτέρω με την καθηγήτρια την κυρία Σκετίνο. Αφορά την έννοια της μεσογειακής κληρονομιάς Προσπαθούμε τώρα να υλοποιήσουμε κάτι που σχετίζεται με κύβους δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη για πουλμάν και τουρισμό. Αυτό που λείπει εδώ είναι οι στρατηγικές. Ε, αυτή η έννοια αναφέρατε για τα ε, διάφορα προβλήματα, τι απάτες, την ανάπτυξη. Αν δεν τα βάλετε όλα μαζί σε ένα οικοσύστημα, ξεκινώντας ε, από όσα γνωρίζουμε από την πραγματικότητα, βασιζόμενοι σε αυτή, δεν θα πάμε πουθενά, διότι το βασικό πρόβλημα στις μεσογειακές χώρες είναι η οικονομική ανάπτυξη. Η καινοτομία και ο πολιτισμός θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και τα μεγάλα δεδομένα, η νέα αυτή η τεχνολογία θα συμβάλλει σημαντικά, θα ωφελήσει σημαντικά ένα τέτοιο οικοσύστημα σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς αναπτύσσουμε πιλωτικά έργα σε, ολόκληρες, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου θα, ήταν, θα θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος να απαντήσει. Παρακαλώ. Ε, Πρώτα απ' όλα, πράγματι πιστεύω και εγώ ότι ο πολιτιστικός τουρισμός ε, μπορεί να αποτελέσει μέσο συνειδητοποίησης της ιστορίας της Ευρώπης της ιστορίας της Μεσογείου και της αξίας ε, της ε, κληρονομιάς γενικότερα, ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη δική μου πρόταση ήθελα να προσθέσω δεν υπογραμμίζουμε μόνο τις τοποθεσίες αλλά και τις διαδρομές. Οι διαδρομές μας δείχνουν την ιστορία, μας δείχνουν τη συνοχή των κοινών μας πολιτισμών της κοινή μα ιστορίας. Ε, δεν ξέρω αν ήμουν σαφής, αλλά είμαι ευχαρίστος να το αναλύσω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αλβάνα Βόξε ε, και είμαι πρόεδρος ε, στην Αλβανική Βουλή της Επιτροπής Πολιτισμικών Υποθέσεων. Ξέρετε ότι είναι πολύ μικρή η χώρα η Αλβανία, αλλά έχει μοναδική ε, πολιτιστική κληρονομιά. Ε, έχουμε Έλληνες, Ρωμαίους, Οθωμανούς, Ιταλούς και τα λοιπά που πέρασαν από την Αλβανία. Ε, μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού ήταν πολύ φτωχή χώρα και ο προϋπολογισμός για τη διατήρηση, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Γιατί λοιπόν παίρνω σήμερα το λόγο. Μια ανησυχία θέλω να σας αναφέρω και ε, ε, ε, μία παράκληση. Η Εθνική μας Βιβλιοθήκη έχει πλημμυρίσει μετά από μία καταιγίδα και μπορούμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να χάνουμε πολύ σημαντικούς θησαυρού. Έχω εδώ επίσης φωτογραφίες από διάφορα γεφρί, γεφύρια. Ο Όστροβα, Οργόσκα και εδώ έχουμε ένα μοναστήρι πολύ παλιό, 300-400 ετών, στη Νότια Αλβανία και ε, χάνονται αυτοί οι θησαυροί, εξαφανίζονται ε, λόγω της αδιαφορίας των κρατικών αρχών. Αλλά αυτή, ε, αυτός είναι το κτίριο του αλβανικού, του ιταλικού κύκλου στην Αλβανία και επί 80 έτη ήταν το εθνικό μας θέατρο. Το έχει χτίσει ένας σπουδαίος Ιταλός αρχιτέκτονας. Είναι η τρίτη ε, κατά σειρά εβδομάδα που διαδηλώνουν εκατοντάδες καλλιτέχνες μπροστά από αυτό το κτίριο γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να το κατεδαφίσει. Ο πρόεδρος διακόπτη. Ε, κοιτάξτε, δεν έχετε χρόνο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εμείς μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα και θα θέλουν να προστατεύσουν οι καλλιτέχνες αυτό το θέατρο και η κυβέρνηση αποφάσισε να ε, το γκρεμίσει και να το δώσει σε ιδιώτες να χτίσουν πολυκατοικίες. Εντάξει, το είπατε, είστε σαφείς, πρέπει να σταματήσετε. Καταλάβαμε το μήνυμά σας. Ε, αυτές οι χώρες σαν την Αλβανία θέλουν βοήθεια. Poate, nu vă poate Δεν μπορώ ε, να σας απαντήσω εγώ. Ε, άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καταφέραμε να καλύψουμε τα 20 λεπτά καθυστέρηση που είχαμε. Βάζουμε εδώ μια τελεία και παρακαλώ τα μέλη του επόμενου πάνελ να έλθουν. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle, oui. Monsieur Radou, n'ayez pas... Η πρόεδρος, κύριε Ράντου, μη φοβάστε, ελάτε εδώ δίπλα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 Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, λέει η Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε αυτήν την όμορφη συνεδρίασή μας. Και είναι τιμή για μένα που προεδρεύω εδώ. Είμαι η Καρίνα Ντελή, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι η πιο νέα σε ηλικία πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εδώ και ειλικρινά είμαι συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη ευτυχία, αλλά θα επανέλθω. Αυτή η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για ένα θέμα τόσο σημαντικό όπω είναι ο πολιτιστικός τουρισμός για μένα που είμαι πρόεδρος, όπως σας είπα, τη επιτροπή αυτή, βλέπετε, έχω τη θέση του κύριου Ταγιάννη εδώ πέρα και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Λέτε να σημαίνει τίποτα ότι κάθομαι στη θέση του. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πολιτιστικό τουρισμό είναι ένα επιθυμητό, ε, ευχαίος, ε, ε, είναι κάτι που βοηθάει στη συνοχή, είναι ένα τουρισμός, ο πολιτιστικό που λαμβάνει χώρα όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με δραστηριότητες πολλές και διάφορες. Όταν μιλάμε για τουρισμό, μπορούμε να μιλήσουμε για φαγητό, μπορούμε να μιλήσουμε για θρησκευτικό τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα μνήμης επίσης. Γιατί οι τοποθεσίες οι τουριστικές μας μιλούν για την ιστορία, για το παρελθόν. Επίσης πρόκειται και για μυρουδιές, για ομορφιά, για τοπία. Όλα αυτά σας τα λέω για να σας πω ότι πρέπει να σεβόμαστε τους τουριστικούς προορισμούς. Σήμερα έχουμε περάσει από έναν τουρισμό για τις ελίτ, δηλαδή στον οποίο δεν είχαν πρόσβαση όλοι, και έχουμε φτάσει σε ένα τουρισμό πολύ πιο προσβάσιμο με 40% επισκέψεις ε, του κόσμου σε διάφορες τουριστικές ε, περιοχές και ο τουρισμός θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος για να κάνει τουρισμό θα διαφέρουν όλο και περισσότερο και ο αριθμός των επισκεπτών επίσης θα αυξηθεί είτε έρχονται από την Ινδία, είτε έρχονται από την Κίνα που δεν ε, τον ξέρουν τον τουρισμό όπως τον ξέραμε εμείς που πηγαίναμε το καλοκαίρι διακοπές και κάναμε τουρισμό. Για αυτούς τουρισμός είναι για όλη τη χρονιά, οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Συνεπώς, ο τουρισμός και ο πολιτισμός Μερικές φορές συνεπάρχουν δύσκολα. Υπάρχουν προβλήματα μαζικού τουρισμού που καταστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά. Μιλάμε για το κέντρο μερικών πόλεων με υπερβολικά πολύ τουρισμό. Μιλάμε για την απώλεια ταυτότητας. Μιλάμε και σωστά για τον τουρισμό marketing. Έτσι τον τουρισμό που είναι της μιας μέρας, μερικών ωρών. Μιλάμε για το φτηνό τουρισμό που δημιουργεί άλλα προβλήματα και όλα αυτά βέβαια για μας είναι μια μεγάλη πρόκληση γιατί είναι σαν να χορεύουμε πάνω σε ένα ηφαίστειο. Γιατί και ο τουρισμός με το κλίμα και τον πλανήτη μας έχουν άμεση σχέση. Οπότε μπορεί να είναι καλός για τον τοπικό πληθυσμό, για την οικονομία. Το δικό μου όμως το μήνυμα είναι ότι ο πολιτιστικός πολιτισμός έχει ένα πολύ καλό μέλλον μπροστά του. Αν βασίζεται στο σεβασμό της ιστορικής μας κληρονομιάς, θα εξελιχθεί, θα αποκτήσει νέες μορφές. Ακριβώς γιατί βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ψηφιακές εξελίξεις. Άρα θα γίνει πιο δημιουργικός ο τουρισμός αυτός, θα έχει μια σχέση με τον πολιτισμό πολύ πιο σύγχρονη. Σε τοπικό επίπεδο θα είναι πιο ζωντανή αυτή η σχέση και η ψηφιοποίηση θα παίξει επίσης σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του τουρισμού πρέπει να δούμε μεθαύριο τι επαγγέλματα θα έχουμε σε αυτού του είδους τον νέο τουρισμό, τον ψηφιακό. Μήπως δεν υπάρχουν ε, αρκετές ρυθμίσεις. Ξαφνικά τα Airbnb ξεφυτρώνουν παντού. Τι θα κάνουμε με αυτές τις πρακτικές. Πώς θα φροντίσουμε ο τουρισμός αυτός να μοιραστεί όλο το χρόνο πραγματικά. Πρόκειται για μια νέα οικονομία επίσης που έχουμε μπροστά μας, την συμμετοχική με συμμετοχή όλων. Αυτή η νέα οικονομία όμως μερικές φορές μας βάζει μπροστά σε προβλήματα. Σήμερα δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι ο τουρισμός των ελίτ είναι παρελθόν. Βελτιώνεται η κινητικότητά μας στην Ευρώπη, μπορεί οποιοδήποτε να ταξιδέψει σήμερα. Στο κάτω-κάτω αυτό δημιουργήσε και η Ευρώπη. Το Rail, για παράδειγμα, που επιτρέπει στην νεολαία να ταξιδεύει και να ανακαλύψει την Ευρώπη. Όμως θα πρέπει να δούμε και από πιο κοντά πώς έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος στον τουρισμό. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Οπότε λίγα θα πω ακόμα. Ο αυριανός τουρισμός είναι εκείνο ο οποίος θα βοηθήσει την δημιουργικότητά μας να ανθίσει, που θα βάλει τη φαντασία μας να δουλέψει, που θα μας επιτρέψει να μην φοβόμαστε το μέλλον, να μην λέμε ήταν καλύτερα παλιά. Όχι, ο αυριανός τουρισμός είναι ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε νέες εμπειρίες. Οπότε με ιδιαίτερη χαρά σήμερα σας παρουσιάζω εδώ εξαιρετικές προσωπικότητες που έχω δίπλα μου. Σας το λέω ειλικρινά. Είμαι συγκινημένη, πραγματικά πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι δίπλα σας. Ο κύριος Ράντου Μιχαηλάνου Πρέπει να ξέρετε ότι συγκινήθηκα από την ταινία σας το κονσέρτο. Και συγκινούμε πάρα πολύ γιατί είναι μια από τις πιο όμορφες ταινίες που είδα ποτέ η συναυλία. Είναι ειλικρινά μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι δίπλα σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Επίσης, Στο πάνελ αυτό έχουμε και συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Κριστιαν Έλερ για παράδειγμα. Εξ αριστερών μου. Ε, είσαστε συνεισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας έκθεσης η οποία αναφέρεται ακριβώ στην συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την, ε, τον κλάδο της δημιουργία, αλλά και για τις πολιτιστικές ε, διαστάσεις. Μπράβο που είσαστε μαζί μας, ευχαριστούμε. Έχουμε τον κύριο Μοργάνο επίσης και εσείς είσαστε ευρωβουλευτής, συνεισηγητής επίσης της ίδιας έκθεσης, συνεργάζεστε εσείς οι δύο για την έκθεση αυτή που αφορά τους κλάδους της δημιουργίας και την πολιτιστική πολιτική που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε επίσης μαζί μας τον Φρανσίσκο Μιλάν Μον. Καλώς ήρθατε στο πάνελ. Είσαστε συμπρόεδρος μιας διεκνουλευτικής ομάδας που ονομάζεται Ευρωπαϊκός Τουρισμός, η ανάπτυξή του, η πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι πρόκειται για μια ομάδα ευρωβουλευτών που προσκαλεί εμπειρογνώμονε τακτικά, έτσι ώστε η νομοθεσία μας να μην αποτελεί τροχοπέδι στην ε, πολιτιστική διάσταση. Επίσης, έχουμε την κυρία Κλάντια Ταπαρντέλ. Και εσείς είσαστε συμπρόεδρος της διαγνωριστική αυτής ομάδας και είσαστε και μέλος της Επιτροπής μου. Είσαστε μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, έχουμε και άλλη συγγήτρια. Εδώ είσαστε, κυρία Μικαέλα Σόντροβα. Είσαστε συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντισμού. Τι είναι, πώς ε, ορίζεται, θα μας τα πείτε. Ε, στο πάνελ αυτό έχουμε επίσης την κυρία Σάμαντιτς Μακκοβίτς. Πού είσαστε? Δεν είναι εδώ. Είσαστε εκεί. Είσαστε στην αίθουσα. Σηκωθείτε παρακαλώ για να σας δούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχουμε και τον Κιγιόμ Κίντς. που είσαστε από το Μουσείο του Λούβρου. Θα μας ε, τα εξηγήσετε κι εσείς. Ε, φτιάξατε και ένα κλιπ το οποίο δημιούργησε τεράστιο θόρυβο. Έτσι εγώ το έχω δει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε επίσης τον κύριο Χάρη Φερβέγεν από την Ευρωπαίνα, το Ίδρυμα Ευρωπαϊκή. Πού είσαστε? Α, εκεί είσαστε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχουμε και τον Σέμον Λίτλ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ε, Διαδραστικού Λογισμικού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και έχουμε και τον Λουίτζι Φούσκο Ζιράρ, που είναι πρόεδρος του προγράμματος Click. Σας ευχαριστούμε και σας. Α, συγγνώμη, λέει Πρόεδρος, συγγνώμη, συγγνώμη. Έχουμε και τον Δημήτριο Παντερμαλή μαζί μας, που είναι ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης. Είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Αγαπητά μέλη του πάνελ, θα σας δώσω χρόνο φυσικά για τις παρουσιάσεις σας. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα, μάλλον να σας δείξουμε ένα μήνυμα βιντεοσκοπημένο από την Επίτροπο που είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή τεχνολογία, από την Μαρέγια Γκάμπριελ δηλαδή. Οπότε, να το βίντεο. Αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσά στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης που έχει τεράστια σημασία ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι μια ευκαιρία για μας να επιβεβαιώσουμε, να περάσουμε και πάλι το μήνυμά μας που λέει ότι ο πολιτισμός δεν είναι θέμα επιλογή σήμερα, αντίθετα. Ο πολιτισμός είναι στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, που είναι ελεύθερη, ανοιχτή στον κόσμο και η οποία δέχεται επιθέσεις όχι μόνο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσα σε αυτή. Ο πολιτισμός μας προσφέρει πολλές αρετές. Πρώτα απ' όλα, μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον ε, πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά των άλλων. Έτσι δημιουργείται μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μας. Από την άλλη όμως προωθούμε και την δικιά μας ευρωπαϊκή κληρονομιά, κάτι το αποτελεί ένα καταπληκτικό μέσο για να δείξουμε ποιε είναι οι αξίες μας και να τις προβάλλουμε στη διεθνή σκηνή. Η πολιτιστική κληρονομιά λοιπόν έχει μια οικουμενική αξία για όλους μας ως άτομα, ως κοινότητα, ως κοινωνία. Είναι σημαντικό λοιπόν να την προστατεύσουμε και να την μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι στατικό που ανήκει στο παρελθόν. Στην πραγματικότητα όμω είναι κάτι που εξελίσσεται μέσα από την ε, δικιά μας προσοχή. Έχει πολλές και διαφορετικές ε, μορφές, απτές όπως είναι τα μνημεία μας, οι πόλεις μας, ε, τα έργα τέχνης μας, αλλά και άλλες μορφές όπως είναι η πρακτική, η λογοτεχνία, η γνώση. Σήμερα η ψηφιακή επανάσταση που βρίσκεται στην καρδιά των σύγχρονων κοινωνιών μας επιτρέπει να βάλουμε τον πολιτισμό στο κέντρο της ζωής όλων των πολιτών. Σύντομα θέλω να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα που έχουμε, που είναι τέσσερα βασικά και που δείχνουν τι πρόοδο κάνουμε. Η πρώτη πρωτοβουλία που θα αναφέρω είναι η στρατηγική μας Digital for Culture. Είμαι πεπισμένη ότι έχει μεγάλη αξία ο ψηφιακό κλάδο. Έτσι δημιουργείται και Ε, όλοι έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό και βελτιώνουμε την αξία της. Και είναι πολύ βασικό για τον πολιτισμό μας και αποτελεί και προτεραιότητα δικιά μου που είμαι επίτροπος υπεύθυνη για τα ψηφιακά. Βασίζεται σε έξι πυλώνες στρατηγική μας. Πρώτα απ' όλα διεύρυνση και δημοκρατισμός της πρόσβασης στον πολιτισμό. Δεύτερον, πρόθεση, εμπορία του, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τρίτον, παραγωγή και ψηφιακή διανομή. Τέταρτον, προσόντα, ε, ικανότητες. Πέμπτον, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Και τέλος, διεθνή συνεργασία προκειμένου να προωθήσουμε αυτήν την ήπια δύναμη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Η δεύτερη πρωτοβουλία που θα αναφέρω σήμερα είναι η ανανέωση της δέσμευσής μας υπέρ του οπτικοακουστικού κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ανταγωνιστικότητά του και την πολιτιστική ποικιλομορφία μέσα από το πρόγραμμα Europe Creative. Στα πλαίσια βέβαια του περιορισμένου προπολογισμού που έχουμε και ιδιαίτερα μάλιστα με το βάρος του Brexit, εγώ δεσμεύτηκα προκειμένου να στηρίξω ένα φιλόδοξο προπολογισμό για τον οπτικοακουστικό κλάδο και πρότεινα να επενδύσουμε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020 με 2027. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει αφενός την ιδιαίτερη αξία που έχουν τα οπτικοακουστικά έργα που αποτελούν και το άνισμα το πολιτιστικό που προτιμούν οι συμπολίτε μα και από την άλλη μεριά γινόμαστε και πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τι επενδύσει μα σε ένα χώρο αριστεία. Η τρίτη πρωτοβουλία που συνδέει την πολιτιστική ε, κληρονομιά είναι τα ευρωπαϊκά έργα, ένα, μια καταγραφή των ευρωπαϊκών έργων, κάτι το οποίο ανακοίνωσα στο Βερολίνο. Είναι κάτι το οποίο στηρίζουν πάρα πολλοί καλλιτέχνε και δημιουργοί έτσι ώστε τα έργα τους να γίνουν γνωστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο και στους επαγγελματίε και στον υπόλοιπο κόσμο και να προβληθούν περισσότερο, άρα να αξιοποιηθούν περισσότερο. Είναι μια απλή ιδέα η οποία διαρθρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα αναπτύξουμε μια βάση δεδομένων για τους επαγγελματίες που θα έχει τα χαρακτηριστικά της ε, διανομής και της εκμετάλλευσης των ε, ταινιών. Οι υπηρεσμοί μου συνεργάζονται με τον κλάδο και προχωράμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ήδη από το 2019. Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος είναι να διευρύνουμε την πρόσβαση στη βάση δεδομένων και τις πληροφορίες που περιλαμβάνει αυτή έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει σε όλους τους πολίτες. Προσφέροντας για παράδειγμα ε, ό,τι προσφέρεται online νόμιμα. Τέταρτη πρωτοβουλία, πολύ σημαντική, Υπενθυμίζω τη μοναδική αξία τη Ευρωπαϊνα, που είναι η μοναδική online πλατφόρμα που επιτρέπει την πρόσβαση σε πάνω από 51 εκατομμύρια έργα τέχνης, αντικείμενα, βιβλία, βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα που προέρχονται από 3.300 πολιτιστικά ιδρύματα από όλη την Ευρώπη. Είναι ο καλύτερο τρόπο για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Και πέρα από όλα αυτά τα συγκεκριμένα, θέλω να αποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία, παρακαλώ, για να υπενθυμίσω ότι όταν καταλήξουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα δικαιώματα ε, του δημιουργού, θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση για όλους μας όσον αφορά το ψηφιακό κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ε, πρέπει να είμαι σύντομη, οπότε θα τελειώσω υπενθυμίζοντα και επαναλαμβάνοντα την ε, υποχρέωση που έχω αναλάβει υπέρ των ψηφιακών ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι και το όραμα που έχω για την ψηφιακή τροποποίηση και ελπίζω να τα καταφέρουμε και να είμαστε έτσι στην υπηρεσία των πολιτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καρποφόρες εργασίες. Merci à notre... Ευχαριστούμε την Επίτροπό μας για το μήνυμα αυτό. Αρχίζουμε αμέσω. Από εσά, κύριε Μιχαηλεάνου. Μιχαηλεάνου. Μιχαηλεάνου στα ρουμανικά. Στα γαλλικά είναι Μιχαηλεάνου. Λοιπόν, είστε σκηνοθέτης, ε, κινηματογράφου, ποιητής, Γάλλος σεναριογράφος. Για όσους σας γνωρίζουν, Έχετε γράψει και μια ποιητική συλλογή. Ναι, πάρα πολύ παλιά, πάνω από 30 χρόνια πριν. Ε, ένα κύμα με ναυτία, λέει, για τη συλλογή αυτή. Διατελέσατε ε, και πρόεδρος ε, της Κριτικής Επιτροπής σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ και είστε και επίτιμος πρόεδρος του δικού μας κινηματογραφικού βραβείου Λουξ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσατε λίγο το μήνυμα της Επιτρόπου μας και είστε σκηνοθέτης, κινηματογράφο. Πώς μπορεί κανείς με τις ταινίε και με αυτό το πολιτισμό να προσπαθήσει να φτάσει στις ευρωπαϊκές αξίες. Και σας καλώ όλους να δείτε αυτή την καταπληκτική ταινία, ε, στην αυλία ε, για το πώς αντιμετωπίζετε και πώς προσεγγίζετε την ευρωπαϊκή μας κληρονομιά ε, σε σχέση με την καθημερινή τέχνη και τη δική μας αποστολή. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε, έχετε το λόγο. Καταρχάς, σας ευχαριστώ και εγώ. Είμαι και πρόεδρος μιας ε, ε, ένωσης που ονομάζεται ΛΑΧΚ και εκεί συμμετέχουν δημιουργοί, παραγωγοί, σκηνοθέτες από τη Γαλλία, την Ευρώπη και παγκοσμίως και υπό αυτή μου την ιδιότητα είμαι παρόν σήμερα. ΑΡΠ λέγεται η ε, Ένωση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωβουλευτές και τον Πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη, όχι απλώς για τη διεξαγωγή και τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης, που είναι πάρα πολύ σημαντική και σε σχέση με τη σημερινή πολιτική σκηνή που είναι αρκετά ανησυχητική η κατάσταση στην Ευρώπη και ελπίζω μέσω του πολιτισμού να καταφέρουμε να κάνουμε να υποχωρήσουν λίγο λαϊκισμός και όλοι οι φόβοι που κατακτούν σήμερα την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο μας βοηθήσατε να κερδίσουμε πολύ σημαντικές μάχες και πρόσφατα σε σχέση με την οδηγία για τα δικαιώματα του δημιουργού, τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι σε καλό δρόμο, ε, ε, ε, εδώ και καιρό ήταν σε κακό δρόμο. Επίσης, για την οδηγία SMA έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα επανέλθω για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή ε, πολιτιστική ποικιλομορφία. Και δεν θυμάμαι και ε, δεν ξεχνώ μάλλον μια πολύ σημαντική μάχη το 2013 που κοντέψαμε να χάσουμε ε, τη λεγόμενη πολιτισμική εξέλιξη στην Ευρώπη που προστατεύει τις ταυτότητες όλες αυτές τις ευρωπαϊκές δώσαμε μια μεγάλη μάχη όλη οι δημιουργοί και θα επανέλθω σε αυτή την πολιτισμική εξαίρεση γιατί είναι η βάση της νομοθεσίας μας που μας προστατεύει και που ε, θα μπορέσουμε όλοι μαζί να χτίσουμε την αυριανή πολιτιστική κληρονομία. Ποια είναι η σημερινή πρόκληση και το διακύβευμα πέρα από τα πολιτικά που σας ανέφερα. Βεβαίως πάντα είναι η ποικιλομορφία. Και ποια είναι η ποικιλομορφία. Όχι μόνο πολιτισμική, αλλά είναι η ποικιλομορφία και η ποικιλία της σκέψης. Η Ευρώπη είναι σήμερα σε θέση να υπερασπιστεί την ποικιλία των σκέψεων που δημιουργούν πρώτα δημοκρατία και στη συνέχεια ισορροπία. Σε ένα πλαίσιο σήμερα και μια συγκυρία που μας προβληματίζει, καθόλου το ψηφιακό. Ο ψηφιακός κόσμος για μας είναι θαυμαστό εργαλείο και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση στα έργα μας. Αλλά ε, η πολιτική συγκυρία είναι αυτή που σας έλεγα προηγουμένως και όχι μόνο αυτή. Σε αυτή την ψηφιακή εποχή και το ψηφιακό κόσμο υπάρχουν γίγαντες που έχουν δημιουργηθεί ε, της ε, πληροφορικής. Και τίθεται το ερώτημα τι εστί πνευματικό δικαίωμα και ποιο είναι το δικαίωμα του δημιουργού απέναντι σε αυτό που ονομάζεται copyright. Γιατί ε, όταν ο Μπομαρσέ και ο Βολτέρος μιλούσαν για πνευματικά δικαιώματα, ήθελαν να απελευθερωθεί η σκέψη από την ηγεμονία των ισχυρών πριν από δύο-τρεις αιώνες και τότε οι ισχυροί ήταν πανίσχυροι, τουλάχιστον έτσι έμοιαζαν, αλλά ήταν σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, ενώ τώρα έχουμε χίλιες φορές παγκόσμιους πανίσχυρους. Άρα θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μην υπερασπιστούμε τα πνευματικά δικαιώματα και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην αμοιβή του δημιουργού. Έτσι ε, οι καλλιτέχνες μπορούν να έχουν διαφορετική σκέψη, διαφορετικές ιδέες από τους ε, και τους ισχυρούς και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί βλέπουμε στις τηλεοράσεις ε, Netflix, Amazon, Disney, Fox ε, και Κινέζοι που θα καταφθάσουν να συνενώνονται και βεβαίως τους οδηγούν και τους βοηθούν μοιραία οι αλγόριθμοι και θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν στους δημιουργούς αυτό που εντός εισαγωγικών ζητεί η αγορά. Άρα υπάρχει μέγας κίνδυνος για την ποικιλομορφία και αυτό ε, σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να υπερασπιστείτε αυτή την έννοια που είναι ευρωπαϊκή και με αυτά τα όπλα θα κερδίσουμε ε, τη μάχη, την οπτικοακουστική, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική μάχη εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Σήμερα ε, ε, ε η νέα γενιά ε, μαγεύεται οπτικοακουστικά. Και παρόλο που κάνω ταινίε εγώ, διαβάζω πάρα πολύ, μου αρέσει και η τέχνη γενικότερα, η ζωγραφική, η μουσική, αλλά δυστυχώς ε, οι νέοι σήμερα πραγματικά καθυλώνονται από τα οπτικοακουστικά και κινδυνεύει η ίδια η δημοκρατία, ε, η ισορροπία, η αγάπη, ο έρωτας και η κατανόηση του άλλου. Τώρα, πώς θα υποφεληθούμε από τα ωφέλη της ψηφιακής οικονομίας. Τα ακούσαμε προηγουμένως. Με ρύθμιση. Γιατί η ρύθμιση, καμιά φορά τρομάζει. Γιατί κανείς νομίζει ότι θέλει να περιορίσει την ελευθερία του. Όχι. Όταν είναι καλά σχεδιασμένη η ρύθμιση και καλά κατερτισμένη, ε, είναι μια ισορροπία. Ένα δούνε και λαβίν. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακές χρειάζονται αγορές, δηλαδή χρειάζονται και θεατές και χρήματα. Δεν είναι καθόλου κλειστές ούτε εμεί είμαστε κλειστοί να έρθουν στην αγορά. Βεβαίω να υποφεληθούν από το δικό μα κοινό που είναι ε, καλλιεργημένο και χρειαστήκαμε αιώνε για να το καλλιεργήσουμε. Είναι ανοιχτή η αγορά μα, αλλά υπάρχει και ένα αντάλλαγμα. Ελάτε στην αγορά μα να έχετε πρόσβαση υπό τον όρο ότι θα συνεισφέρετε κι εσεί στη σημερινή και κυρίω στην αυριανή μα κληρονομιά δεν μπορείτε να επελάβνετε ως αρπακτικά, να έρθετε όλοι εσείς που είσαστε και ισχυροί ως συνεργάτες. Και υπάρχουν μηχανισμοί όπως η οδηγία SMA που είναι τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, 30% ε, ποσόστοση ε, ε, ευρωπαϊκών έργων στην προσφορά κάθε καναλιού και διανομέα και σε ό,τι αφορά το κύκλο εργασιών ε, μπορούμε να επιβάλλουμε ένα ποσοστό επενδύσεων στην προχρηματοδότηση των ταινιών για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπε προηγουμένως ο Jean-Michel Jarre, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που ονομάζεται μεταφορά αξιών, αυτό που σήμερα εγώ ονομάζω τη μεγάλη διανομή, το σούπερ μάρκετ του πολιτισμού. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες εταιρείες που προσελκύουν συνδρομητές ε, γιατί ε, λένε είμαι πιο φθηνός. Είδαμε όμως μετά από 30 χρόνια τι σημαίνει μεγάλη διανομή. Το φτηνό και το ακόμα φτηνότερο τελικά σκοτώνει τους γεωργούς, στη γη και τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Τελικά σκοτώνει και την ανθρώπινη υγεία. Χρειαστήκαμε 30 χρόνια για να καταλάβουμε ότι το βιολογικό ε, δεν είναι και πολύ κακό. Και τώρα ε, ε, θα χρειαστούμε 30 χρόνια για να δούμε ότι θα έχουν καταστραφεί ο πολιτισμός, η παραγωγή, οι καλλιτέχνε και τα σχολεία για να γίνει ένα σούπερ μάρκετ η διανομή ε, του πολιτισμού και μετά θα ξαναγυρίσουμε στα βιολογικά. Προσοχή με τις ετικέτες, προσοχή στις ετικέτες, δεν μετράει η ετικέτα. Αξία έχει το περιεχόμενο και όχι αυτός που το πλασάρει. Θα πρέπει λοιπόν στην νομοθεσία να δούμε πώς θα έχουμε κατόφλια ε, κατώτατε τιμέ για τα έργα για να μην τα ξεπουλούν στο όνομα του φθηνού και να μην κερδίζει τελικά η μάρκα και η ετικέτα. Επίσης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα φαινόμενο που κινδυνεύει να αποκλείσει ορισμένους από την πρόσβαση στον πολιτισμό, ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν τα ε, υλικά μέσα. Μπορεί να βρείτε τον Κοντάρα, ας πούμε, στο Netflix στο μέλλον και για πάντα να είναι κλειστό, εκεί, Orson Welles στο Amazon και ο Τριφό δεν ξέρω πού. Και ένας νέος που δεν μπορεί να πάρει τη συνδρομή ε, ή όλες αυτές τι συνδρομές δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτή τη δημιουργία και δεν θα ε, μπορέσει να καλλιεργηθεί ε, καλύτερα. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε στο νομοθετικό πλαίσιο για να αποφύγουμε το γεγονός αυτό, να μην είναι φυλακισμένα τα έργα στον αιώνα των άπαντα σε ένα κανάλι. Ξέρω ότι έχουμε καθυστέρηση. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο την κυρία Μαρία Γκάμπριελ για αυτή την πρωτοβουλία. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τους ε, κινηματογραφιστές και σκηνοθέτες του ΑΡΠ να κάνουμε και μια μηχανή αναζήτησης. Υπάρχει ένας κατάλογος οπτικό-ακουστικό στην Ευρώπη που είναι ο πιο ενδιαφέρον ε, στον κόσμο και τώρα που είμαστε και στο παγκόσμιο κύπελο, άμυνα ξέρουμε, επίθεση δεν ξέρουμε. Ε, οι Αμερικανοί ξέρουν πολύ καλά να μας επιτίθενται, γιατί εμείς δεν πάμε ποτέ στο δικό τους γήπεδο. Και είναι εύκολο σήμερα λοιπόν με το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες αυτό το θαυμάσιο εργαλείο, να φτιάξουμε μια μηχανή αναζήτησης όπου όλα τα ευρωπαϊκά έργα ε, θα ε, συμπεριλαμβάνονται και στην Ευρώπη έχουμε ιδιοφυΐες και όχι μόνο, παράγουμε και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Και εμεί, οι Ευρωπαίοι είμαστε οι μόνοι που ε, έχουμε δικαιώματα ε, ε, από την Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία και ορισμένα από τη Βόρεια Αφρική, Αμερική, συγγνώμη. Ε, ε, να δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η μηχανή αναζήτησης και μετά ένα παγκόσμιο βίντεο on demand. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε για όλες τις ταινίε και να μπορούν παντού να προβάλλονται εκεί που δεν πουλούνται. Και υπάρχουν αριστουργήματα που κερδίζουν φεστιβάλ και νομίζουμε ότι διανέμονται παντού στον κόσμο. Ε, λοιπόν, μόνο σε 40 χώρες γίνεται αυτό. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να τα διανύουμε και να τα έχουμε στη διάθεση όλων των χωρών του κόσμου και για να προκαλέσουμε λίγο τους Αμερικανούς που μας στέλνουν όλες τις ταινίε τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί μερικές είναι αριστοργήματα. Καλό θα ήταν να υπάρχει και μια αμοιβαιότητα και να έχουμε και τεχνολογικά που μπορούμε τη δυνατότητα να στέλνουμε και τα δικά μας έργα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας. Ε, ήταν ε, πολύ ε, ηχηρά κάτι χαρακτηριστικό δικό σας. Μιλήσατε για την αμοιβαιότητα. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τους μεγάλους που να συνθλίβουν πάντα τους μικρούς. Και επίση είπατε κάτι σημαντικό. Τα δικαιώματα δημιουργού βοηθούν ε, στην επιβίωση των καλλιτεχνών. Και αυτό πρέπει να δούμε. Η δωρεάν δουλειά των καλλιτεχνών δεν είναι πια κάτι δυνατόν. Το να δουλεύουν δωρεάν σημαίνει το να τους βάζουμε φυλακή ουσιαστικά. Η αμοιβή τους απελευθερώνει από τον έλεγχο των δυνατών. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και θα τελειώσω με κάτι πολύ όμορφο που είπατε, προσπελάσιμο για την πλειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ε, διάδοση της δουλειάς σας, ε, πρόσβαση, να είναι προσβάσιμη. Αυτό που μαθαίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα τα εργαλεία τα οποία ε, βοηθούν ε, τους πολίτες μέσω των ταινιών, μέσω της τέχνης σας, ε, ώστε να δημιουργηθεί μια συνείδηση στους, στους πολίτες, μέσω των δικών σας αμέσων. Είναι πολύ δυνατά τα λόγια αυτά που είπατε εδώ, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αφού μιλάτε για τουρισμό, να σας θυμίσω ο πολιτισμός μου έφτιαξε τα πιο όμορφα ταξίδια που έκανα στη ζωή μου μέσω της υποκειμενικότητα των άλλων. Αυτό είναι ο πολιτισμό. Ε, είναι ένα όχημα ειρήνη, όχι πολέμου. Η δυνατότητα να ταξιδεύει ε, στο φανταστικό κανεί μέσω του πολιτισμού. Πρόεδρος, μπορούμε να σας χειροκροτήσουμε για αυτά τα πολύ καθαρά ηχηρά σας λόγια, σημαντικά λόγια που ακούσαμε εδώ, εδώ στο κοινοβούλιο που υπερασπιζόμαστε αυτές τι αξίε. Αξίε που όπω είπατε και εσεί ε, δεν μπορούμε να διαφημίζουμε το πουλάμε έτσι. On passe à vous, Monsieur Heller, notamment. Κύριε Έλερ, συνεισηγητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ε, πολιτική ευρωπαϊκή συνοχή για την πολιτιστική πτυχή και, τις, και ε, τους τομείς δημιουργίας. Σας δίνω το μικρόφωνο. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που έχετε παραμείνει εδώ. Το τίμημα είναι ότι αγγίζουμε λίγο πιο πολύ την πολιτική πτυχή της συζήτησης. Μου ζήτησε ε, ο συνάδελφος από την Επιτροπή Πολιτισμού, κ. Μόργανο, να αναφερθώ λίγο ε, στην εμπορική διάσταση του τομέα αυτού. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αποφύγω μια παρανόηση το Κοινοβούλιο το απέδειξε ότι εκτιμάμε συναισθηματικά συμφωνούμε μαζί σας. Μπορεί εσείς να μην το πιστεύετε σε ένα τέτοιο χώρο, αλλά εμείς εκτιμάμε αυτό που κάνετε εσείς. Την μη εμπορική διάσταση της πολιτιστικής ε, ε, κληρονομιάς. Και αυτό ήρθαμε εδώ να ε, γιορτάσουμε, να χαιρετήσουμε, να υπογραμμίσουμε ως κάτι σημαντικό. Δεν είναι όμως αντίφαση να δούμε και την εμπορική πτυχή. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κομμάτι του τομέα της δημιουργικότητας και του πολιτισμού στην Ευρώπη. Τομέας ε, που απασχολεί 2,5 φορές περισσότερους ανθρώπους από ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ε, οι άλλες, ε, η χημική βιομηχανία, πέντε φορές περισσότερο από ό,τι η χημική βιομηχανία. Για να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Μιχαηλεάνου, αν ψάξετε στο Google σήμερα το άρθρο των Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα ότι η Google δαπάνησε τρία ψηφιακά εκατομμύρια σε lobbying στις Βρυξέλλες κατά του copyright εκεί διαφαίνεται η εγγενής εμπορική ε, οπτική γωνία που αντιλαμβάνεται η Google αλλά που δεν καταλαβαίνουν συχνά οι πολιτικοί στην Ευρώπη Δεν το λέω για να δώσω πολιτική έμφαση. Αυτό δημιουργεί, ε, μας δείχνει τι γίνεται με τους ε, λομπίστες ε, και την πολιτική πλατφόρμα. Είναι κάτι επικίνδυνο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικά χρόνια στο τέλος της πολιτιστικής ε, πολυμορφίας στην Ευρώπη. Ναι, ε, υπάρχει αυτή η πολιτιστική διάσταση και η πολιτική και συνδυάζονται αυτές οι δύο και πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ συμβάλλει η πολιτιστική κληρονομιά ως κινητήριος δύναμη για τις τοπικές οικονομίες, ως ε, μηχανή έμπνευσης ε, των τομέων του πολιτισμού, του τομέα του πολιτισμού. Μας οδηγεί ξανά στο ερώτημα της συνοχής ε, στην Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την εμπορική του διάσταση Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε. Και γι' αυτό το λόγο, για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Βιομηχανίας και η Επιτροπή Τουρισμού, που συνήθω δεν είναι ε, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Για πρώτη φορά ευθυγραμμίστηκαν κάνοντας αυτή την έκκληση προς την Επιτροπή προς τη, στις Βρυξέλλες να υπάρξει μια ε, συνοχή στρατηγικής σε θέματα πολιτισμού και ε, τομέα της δημιουργικότητας. Βρισκόμαστε στην αφετηρία και αυτό είναι ένα καλό σημείο. Βρισκόμαστε στην αφετηρία ενό κρίσιμου ε, μια κρίσιμη συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες και θα δείτε ότι θα χρηματοδοτήσουμε ε, την πολιτιστική κληρονομιά και το, και το σχετικό κλάδο στην Ευρώπη ε, πέραν από το απλά να χρηματοδοτούμε ταινίε. Νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά κατανοητή αυτή η διάσταση σε αυτό το τομέα απασχολούνται οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Αυτό, σε αυτό τον τομέα, όχι σε άλλον. Ε, αυτό που σας λέω βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Εδώ απασχολούνται οι περισσότεροι και μάλιστα όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επανεκβιομηχάνηση. Πάντα συζητάμε για το χάλιβα και άλλα τέτοια, αλλά αν συγχωνεύσουμε τη δημιουργικότητα ε, με τις ε, τέχνες, αυτό θα οδηγήσει σε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν Δείτε τα πολυτελεία, δείτε μια τσάντα που παραγείται στην Βόρεια Ιταλία ή στην Γαλλία. Γιατί είναι τόσο σημαντική στην, στην Κίνα, στην Ασία, διότι περιλαμβάνει όχι μόνο στυλ, ε, αντιπροσωπεύει τη μοναδικότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό την καθιστά τόσο ελκυστική ως καταναλωτικό είδος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά πρέπει να το μεταδώσουμε κάπως αλλιώς ε, εδώ σε μια τέτοια συνάντηση απλά αναφέρουμε την ε, ε, πνευματική ανωτερότητα του θύματο. Δηλαδή, ξεπουλιόμαστε στην Google, δεν κάνουμε τίποτα σε θέματα έρευνα ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αυτό πιστεύω πρέπει να αλλάξει και εμεί θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Θα δείτε ότι θα χρηματοδοτήσουμε αυτήν την κληρονομιά. Θα υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ έρευνας και πολιτισμού. Θα πρέπει αυτή μας η κληρονομιά να ενσωματωθεί στο Ταμείο Συνοχής. αυτό το μάθημα πρέπει να ε, κρατήσουμε ότι έχουμε ε, λειτουργήσει απομονωμένα κάπως. Τώρα βλέπουμε τις δυνατότητες αλλά και τις απειλές και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε σήμερα. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το βαθμό στον οποίο η Google και οι διαφορές πλατφόρμες θα ε, μας απορροφήσουν. Στην αντίθετη περίπτωση, τι σημαίνει αυτό οικονομικά για την Ευρώπη, και για τις δημιουργικές δυνατότητες και την ε, πολυμορφία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε αγαπητέ συνάδελφοι. Λοιπόν, τώρα λυπάμαι για τους επόμενους ομιλητές, αλλά έχουμε, βλέπετε, καθυστερήσει πάρα πολύ, οπότε θα πρέπει να χειριστώ το χρόνο. Έχετε δύο λεπτό καθένας. Και έχω εδώ και ένα κουμπί μπροστά μου που κλείνει το μικρόφωνο, να ξέρετε. Λοιπόν, ο κύριος Μοργάνο, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι και προσκεκλημένοι πολλά υπόθηκαν. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος θα εστιαστώ στο γιατί είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά το οποίο έκφραση είναι ο τομέας της δημιουργικότητας ε, και του πολιτισμού. Πρέπει να αξιοποιηθεί διότι η δημιουργική Ευρώπη δημιουργεί αξία, εκφράζει την ψυχή της, την ιδιαιτερότητά της. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε, να αξιοποιήσουμε ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά γιατί είναι ε, ζωή, ε, είναι η φλέβα μέσω των οποίων η δημιουργικότητα, η φαντασία, η ικανότητα να δημιουργήσουμε συναισθήματα, να δημιουργήσουμε ομορφιά, την πραγματική δύναμη της, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη είναι το σημείο συνάντησης τεχνών, πολιτισμού, ε, δημιουργικότητας, δραστηριοτήτων διαφόρων που ε, χαρακτηρίζονται από μια διτή αξία. Τι θέλω να υπογραμμίσω εν συντομία. Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια πραγματική ε, στρατηγική για τον τομέα με συνοχή και μακροχρόνια. Να λαμβάνει υπόψη αυτή η στρατηγική τις σημερινές συνθήκες καθώς επίσης και την πρόσβαση σε πιστώσεις απαραίτητο και όπως ε, μας υπενθύμησαν εδώ να καλυφθεί το χάσμα αξίας, το value ΑΚΑΠ. να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, ε, την παραποίηση, την απομίμηση και να υπάρξει ε, προστασία του δικαιώματος του δημιουργού. Εμείς με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 έως το 2027 θα έχουμε νέα προγράμματα ειδικά από τη Δημιουργική Ευρώπη μέχρι το νέο εμβληματικό πρόγραμμα ε, Horizon. Αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία για αυτά τα προγράμματα και θα αποτελέσουν διάφορες ευκαιρίες που θα υλοποιηθούν με το χρόνο. Ζητούνται πολλά από τον πολιτισμό. Επιμένουμε πολύ στην πολιτιστική κληρονομιά. Για παράδειγμα, ένα εσωτερικό πρόγραμμα τέτοια δομή ε, για την κοινωνία χωρί αποκλεισμού και με ασφάλεια που θα περιλαμβάνει το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο τη ε, Επιτροπή ε, πολιτισμού που θα εξετάσουμε, εκεί θα πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Το λέω διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ευνοήσουμε νέες, νέα γλώσσα, νέες τεχνικές, πρέπει να συμπληρώνουμε την ε, πολιτιστική κληρονομιά, όχι απλά να την διατηρούμε. Θέλω να αναφερθώ στην εικονική πραγματικότητα, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην ολογραφία. Όλα, για όλα αυτά χρειαζόμαστε μια Ευρώπη ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και πιο δημιουργική και πιο ενημερωμένη. Πιστεύω και ελπίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας ριζοσπαστικής προσέγγισης που θα είναι καθοριστική για το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοργάνο. Μια Ευρώπη με τη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμού, ζωντανή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν πρέπει όμως μόνο να το λέμε, πρέπει και να το κάνουμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρανθίσκο Μιλανμόν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη, το είπατε, αποτελεί μια μεγάλη δημιουργική δύναμη, πολιτισμική, με τεράστιο δυναμισμό. Από παλιά ξέρουμε πως έχουμε διαμορφώσει στην Ευρώπη τον τρόπο σκέψης, διάφορους ε, παράγοντες που αναπτύχθηκαν από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, με διάφορες επιρροές βέβαια και εκτός Ευρώπης, που οδήγησαν σε διαφορετικά στυλ δημιουργίας και μια πολυμορφία σκέψης. Οι αλλαγές αυτές βέβαια έχουν περάσει τα εθνικά σύνορα και έχουν οδηγήσει σε ευρωπαϊκά στυλ. Υπάρχουν ε, τα μνημεία ιστορικής κληρονομιάς της UNESCO και τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Ευρώπη. Λοιπόν, η πολιτιστική κληρονομιά έχει τεράστια σημασία και πολιτισμική αλλά και αισθητική. Πρόκειται για στοιχεία πολύ ελκυστικά για τον τουρισμό, κυρίως στην Νότια Ευρώπη, για την οποία ο τουρισμός αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και την ιστορική κληρονομιά στην ανάπτυξη. Η αναπαλαίωση ενός μοναστηριού, ενός κάστρου, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό οικονομικό παράγοντα. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ειδικοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αναπαλαίωση των κτίριων. Η ψηφιοποίηση, το είπαμε ήδη, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Η αεροποάνα επίσης, η οποία αναφέρθηκε εδώ. Αλλά επίσης η πολιτιστική κληρονομιά έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη δημιουργία για την ε, διατήρηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε σε εποχές λαϊκισμού. Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των Ευρωπαίων και γι' αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρηθεί αυτή η πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι μόνο η κοινωνία των πολιτών, η περιφέρεια, η δήμοι, οι κοινότητες κτλ. Και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να κάνουν το δικό τους. Με προγράμματα, ε, με δράσεις, αλλά και με ειδική χρηματοδότηση από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Νομίζω ότι δύο λεπτά μίλησα, όχι παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που πήρατε το λόγο, <clears throat> κύριε Μιλάν Μον. Όντως, αναφερθήκατε στον τουρισμό, τον ιστορικό τουρισμό, το υπογράψετε τώρα. Κυρία Ταρταντελ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ και μιλάω εδώ από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η πρώτη φορά που θα ακούσετε και τα ρουμάνικα σε αυτήν την αίθουσα. Θέλω λοιπόν να στείλω το μήνυμά μου υπέρ της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που αναφέρθηκαν στον ευρωπαϊκό τουρισμό και το ρόλο που μπορεί να παίξει η πολιτισμική κληρονομιά. 140 μέλη έχουμε εδώ από διάφορες χώρες και κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέχρι τώρα για να προωθήσουμε την ανάπτυξη του πολιτισμικού πολιτισμού. Αυτό όμως πηγαίνει χέρι-χέρι και με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πολιτιστικός ε, τουρισμός δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν προστατεύσουμε τον πολιτισμό και τα μνημεία στις χώρες μας. Χάρη λοιπόν στα προγράμματα που εμείς προωθούμε, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των χωρών μελών στη σημασία που έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική. Πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα του τουρισμού και της πολιτισμικής κληρονομιάς και πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση για όλα αυτά. Αλλιώς η κληρονομιά αυτή που είναι τόσο διαφορετική, τόσο πλούσια και τόσο σημαντική για την ταυτότητά μας θα εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε ότι η κληρονομιά είναι πολύ σημαντική και για την οικονομία μας. Υπάρχουν ε, τουριστικές περιοχές κορεσμένες ε, σήμερα, πολύ φορτωμένες. Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περιοχές με τεράστιο τουριστικό δυναμικό και δυνατότητες. Και όχι μόνο στο Παρίσι, το Μιλάνο, τη Βαρκελόνη ή την Βενετία. Γι' αυτό πρέπει, οφείλουμε, οι πολιτικοί ηγέτες δηλαδή, να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους τουρίστες και όχι μόνο τους Ευρωπαίους να πηγαίνουν και σε αυτές τις περιοχές που είναι πάρα πολύ ελκυστικές γιατί διαθέτουν πολιτισμική κληρονομιά και αυτές. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω και να πω προσοχή, ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βοηθήσει την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, τότε Πώ θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι χρέο μα Οφείλουμε να οργανώνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως είναι η σημερινή και να πούμε ότι στον ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να περιλαμβάνεται και μια στρατηγική υπέρ τη ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά. Νομίζω θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε μαζί μα την πρόεδρο τη Επιτροπή Τουρισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τουρισμού. Συγγνώμη αν ξεπέρασα το χρόνο μου, όλοι τα πράγματα που νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να υποθούν για να προωθήσουμε την κληρονομιά μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ταπαρντέλ. Και θυμίζω ότι ο τουρισμός και η κληρονομιά βεβαίως θα πρέπει να μείνουν στα χέρια των κρατών, αλλά να υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Σόιντροβα. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που παραμείνατε εδώ για να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού που ε, ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και είμαι η συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ε, αυτό το σχέδιο εθελοντισμού μετά το 2020. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το σκέλος του πολιτισμού εδώ και έχει μεγάλο δυναμικό να προσελκύσει νέους με διάφορους τρόπους ε, στον πολιτισμό για να συμμετέχουν σε διεθνή έργα και προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει δύο σκέλη, και εθελοντικό σκέλος και ένα σκέλος με απασχόληση, αμοιβόμενη εργασία και καλύπτει την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες ε, εν αποθέσει. Ελπίζουμε να επιτύχει. Βεβαίως οι νέοι θα βρουν νέες ευκαιρίες, θα γνωρίσουν νέα περιβάλλοντα στην Ευρώπη, θα μάθουν τι σημαίνει να είσαι μέλος της ευρωπαϊκής ε, κοινωνίας. Γι' αυτό θέλω να ε, απλουστευτεί η διοίκηση του προγράμματος για να είναι πιο ε, εύλεπτο και πιο κατανοητό και πιο προσβάσιμο. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς πραγματικά εστιάζει στους νέους και θα δώσει αυτό μια νέα όθηση σε όλη την Ευρώπη μας. Θέλω να θυμίσω κάτι που είχε πει ο Άγιος Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος λίγο μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος. Η Ευρώπη αναγκάστηκε να ε, αναζητήσει ένα νέο προσδιορισμό στην ταυτότητά της πέρα από πολιτικά ε, συστήματα και στρατιωτικούς συνασπισμούς. Ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό της ως ήπειρο πολιτισμού. Μια γη ποτισμένη με ε, τη χριστιανική πίστη 2.000 ετών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα αυτές οι βαθιές σκέψεις φαίνεται να είναι ακόμα πιο επίκαιρες από την εποχή που είχαν εκφραστεί. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Η ε, Ευρώπη μπορεί να ανανεωθεί. Η ομορφιά θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο όπως ήλπισε κάποτε για την Ευρώπη ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Η Ευρώπη με την ομορφιά της μπορεί να μας ενώσει και πάλι με τον πλούτο και την ποικιλομορφία μας την πολιτιστική που έχουμε. Κατά τη διάρκεια αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτισμικής Κληρονομιάς είχαμε πολλές ωραίες ε, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Το Σεπτέμβριο 2018 έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στη χώρα μου, στο κέντρο της Ευρώπης, στη Τσεχική Δημοκρατία. Έχουμε μια έκθεση ε, για ε, τα χρόνια της ε, σύγχυσης και της απελπισίας. Είναι μια διεθνής διάσκεψη στο Κρόμερσιτς, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, και ελπίζω αυτά να βοηθήσουν όχι μόνο τους νέους ανθρώπους αλλά και την Ευρώπη ολόκληρη να ανακαλύψει και πάλι τον εαυτό της ως υπήρο πολιτισμού. Όπως ε, είχε εκφράσει την ευχή αυτή ο, ο Άγιος Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Τέλος αγαπητοί φίλοι στα γαλλικά επιτρέψτε μου να απαντήσω στην έκκληση του Ζαν Μισελ Ζαχ και επίσης του συναδέλφου Μιχαηλάνου διότι μας ζήτησαν να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε ε, τους ε, δημιουργούς και τα δικαιώματα των δημιουργών. Νομίζω ότι οφείλουμε να τους υποστηρίξουμε. Φυσικά, τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, των καλλιτεχνών γενικώ, των δημοσιογράφων των ίδιων ε, είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε και να προασπίσουμε. Βεβαίως πάντα εμείς οι θα πρέπει να βρούμε την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του διαδικτύου, στην ελευθερία της έκφρασης και ε, στα δικαιώματα των δημιουργών. Αλλά είναι δική μας δουλειά και καθήκον να βρούμε αυτή την ισορροπία και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Γκυλιόμ Κίντσα. Είστε έφορος ε, της ε, του Μουσείου του Λούβρου. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε με δύο ιδιότητες θα μιλήσω σε εσάς ως επαγγελματίας, ως έφορος ε, του Μουσείου του Λούβρου και ως ε, ιδιώτης, διότι με ε, την οικογένειά μου έχουμε πάρει ένα κάστρο, τον Νταμπιέρα, στη Γαλλία, το οποίο προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε σε εργαστήριο πολιτιστικό σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις που είναι πολύ αριθμές σήμερα και από την εμπειρία μου έτσι μπορώ να σας παρουσιάσω την τοπική και τη διεθνή διάσταση για μια ευρύτερη εικόνα των διακύβευμάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς σήμερα. Ήθελα να μιλήσω στο προηγούμενο πάνελ στη συντήρηση και την προώθηση, αλλά ήταν πολύ απλό. Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι αμάρτημα, είναι ένα πιστεύω το οποίο λειτουργεί μεν, αλλά όχι πλέον μόνο του. Είναι να πιστεύω, μια πεποίθηση που πρέπει να επανασχεδιαστεί όσον αφορά την προσέγγιση, την οικονομία, τα οικονομικά του και την κοινωνική του διάσταση. Στο πάνελ 3 λοιπόν για την καινοτομία ήθελα να προσθέσω εγώ την ε, κοινωνική ωφέλεια. Καινοτομία πρώτα απ' όλα, όχι απλά τεχνολογική. Στις προσεγγίσεις μας επίσης πρέπει να καινοτομούμε όχι μόνο στα μέσα, γιατί για να συνδέσουμε τους πολίτες να ενδιαφερθούν οι πολίτες, να καταλάβουν τι είναι η κληρονομιά, πώς σχετίζεται με το παρόν, ότι η κληρονομιά δεν είναι απλά κάτι παλιό, αλλά κάτι που συνεχίζεται, που έχει συνέχεια, ώστε να καταλαβαίνει πόσο επίκαιρο είναι. Πώς επίκαιρη είναι. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζω μια έκθεση για τον Ελ Γκρέκο στον Γκραν Palais του χρόνου στο Παρίσι. Ο Ελ Γκρέκο, ο οποίο σίγουρα είναι ένα ε, καλλιτέχνη από το παρελθόν, αλλά καθαρά Ευρωπαίο. Γεννήθηκε στην Κρήτη, ε, μετά δραστηριοποιήθηκε στη Βενετία, στη Ρώμη, μετά στην Ισπανία. Γιατί, διότι αναζητούσε εργασία. Και αυτό ήταν ένα μετανάστη. Τέλο, η οικονομία. Τα οικονομικά και αυτά πρέπει να επανεπινοήσουμε στο κάστρο αυτό στο οποίο σας μίλησα παλιότερα υπήρχε μια οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να την ξαναβρούμε. Ένα κάστρο είχε και μια κοινωνική δραστηριότητα. Πρέπει να του βρούμε μια νέα κοινωνική χρησιμότητα σε εποχές ε, δημοκρατικές σήμερα. Επιμένω στην κοινωνική διάσταση. Όταν υπολογίζω τι, ε, τι συμβαίνει εκεί στο Σαμπιέρα, όχι απλά δημιουργούμε πολλές θέσεις εργασίας, ε, άμεσες και έμεσες, Εκεί γίνονται και πολλές συναντήσεις, έχουμε πολλές αναμνήσεις, έχουμε το κάστρο αυτό που ανοίξαμε στον κόσμο ολόκληρο. Φιλοξενούμε ε, καλλιτέχνες αντί να φιλοξενούμε τουρίστες, διοργανώνουμε συναυλίες αντί για γάμους, δαπανούμε 100 ευρώ για ε, ένα φεστιβάλ γαλλοβρετανικό, όχι επειδή είναι το πιο απλό, είναι το πιο επικίνδυνο αλλά και το πιο καινοτόμο και αυτή την καινοτομία ε, θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Αυτή θα κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός μοντέλου ε, αποδοτικού οικονομικού, οικονομικά και ενό βιώσιμου. Για το, πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι η βιώσιμη επιλογή. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν κυκλικέ ε, συνεργατικέ αλληλέγγυε οικονομίε και τα διακυβεύματα να αφορούν κάτι παραπάνω από απλά την πολιτιστική κληρονομιά. Να αφορούν την ένταξη των ανθρώπων, το να κατανοούμε το περιβάλλον μας, να καταλαβαίνουμε την ταυτότητά μας, να αποκτούμε τα μέσα για να το προστατεύσουμε, να μην δημιουργούμε απλά δραστηριότητες αλλά και κοινωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο ε, ο πολιτισμός ε, παίζει κεντρικό ρόλο, αποτελεί έκφραση της κοινωνίας. Όποιος αποδυναμώνει τον πολιτισμό αποδυναμώνει και την κοινωνία. Θα αντιστρέψω την ε, συνήθι λογική Τελειώνουμε συνήθως λέγοντας θέλουμε περισσότερο πολιτισμό στη ζωή. Εγώ θα πω θέλουμε περισσότερη ζωή στον πολιτισμό, διότι σε τελική ανάλυση η κοινωνία δημιουργεί ε, πολιτισμό όταν ο πολιτισμός δημιουργεί ζωή. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και αυτό θα θεωρήσουμε εμείς τιμή μα. Ευχαριστώ για τα λόγια σα. Τώρα, είπατε περισσότερη ζωή στον πολιτισμό. Μπορώ να αποκτήσω δικαιώματα για αυτή τη φράση, για να μπορώ να τη χρησιμοποιώ και εγώ. Μου τα δίνετε, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που μας είπατε. Λέτε μια οικονομία με κοινωνική διάσταση να ξαναζήσει η δημοκρατία με νέα οικονομία που εσείς ονομάζετε κυκλική. Κυκλική, κοινωνική, βιώσιμη, λέμε, βάζουμε πολλές λέξεις πολλούς προσδιορισμού Τώρα το λόγο ο κύριο Παντερμαλής που είναι ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης. Παρακαλώ για δύο λεπτά. <clears throat> Thank you very much, Miss President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η καινοτομία στο Μουσείο της Ακρόπολης συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη του μουσείου αλλά και της περιοχής όπου βρίσκεται το μουσείο και ολόκληρης της πόλης των Αθηνών. Από την αρχή ο σχεδιασμός του μουσείου ήταν τέτοιος για να διασφαλίσουμε την άνεση του επισκέπτη όση ώρα περνάει στο μουσείο. Μέσα από μια σειρά καινοτόμων δραστηριοτήτων στο μουσείο, έχοντας προσέξει πάρα πολύ την διαχείριση των εσόδων και των εξόδων, αλλά επίσης φροντίσαμε ε, και το προσωπικό έδειξε τεράστιο ενθουσιασμό. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για τη μικροοικονομία ε, την τοπική με φοβερά ωφέλη, βελτίωση των τάσεων, ε, λιανικής κλπ. Παρά την οικονομική κρίση που είχαμε, η οποία συνέπεσε με το άνοιγμα του μουσείου. Παρόλα αυτά έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο, κάτι το οποίο βοήθησε ακόμα περισσότερο η Αθήνα να γίνει τουριστικός προορισμός εξοχήν. Τέλος το μουσείο χρηματοδοτείται από μόνο του από τότε που άνοιξε. Χωρίς να έχουμε επιχορηγήσεις από την κυβέρνηση για τη λειτουργία του. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια καινοτομία για ένα τέτοιο θεσμικό πολιτιστικό όργανο. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας κύριε Παντερμαλή. Τώρα, περνάμε στον κύριο Βερβάγεν από το Ίδρυμα Ευρωπαϊκά. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ που με φέρατε εδώ. Αναβάθμιση. Λοιπόν, θέλω να σας πω δύο λόγια για την οικονομική σημασία που έχει η ψηφιακή αλλαγή τη σημασία που έχει για το μέλλον τη Ευρώπη. Δέκα χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια σαφή και επεφοδισμένη απόφαση. Αποφάσισε ότι η πολιτισμική μα κληρονομιά ήταν πάρα πολύ σημαντική για να μείνει στα χέρια τη αγορά και μόνο και να αποφασίζει εκείνη πώ θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν οι πολίτε μα. Και έτσι δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή. Δέκα χρόνια αργότερα, σήμερα δηλαδή, έχουμε μία πλατφόρμα με περίπου 4.000 βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία με 50 εκατομμύρια θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνει η συλλογή μα και χρησιμοποιούνται και ξαναχρησιμοποιούνται από ερευνητέ, δημιουργού και πολίτε που ενδιαφέρονται. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν δεν ε, έφερε σε ζωή το επόμενο Google. Όχι, έγινε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Έγινε ένα καταπληκτικό δίκτυο διανομή, κόμβο για επαγγελματίε οι οποίοι θέλουν να μοιραστούν μεταξύ τους γνώση ε, ανοιχτά ε, ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες για λύσεις και να δημιουργήσουν νέες προδιαγραφές που προσφέρουν γνώση και ανάπτυξη δημιουργίας. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έψαξε να βρει μια φτηνή λύση απλώς να σκανάρει τα παλιά, αλλά απέκτησε μια παραπάνω φιλοδοξία, να αλλάξει νοτροπία και αυτή ακριβώς είναι πραγματική η δύναμη, το ότι η Ευρώπη βασίζεται σε αξίες και σε δράση. Πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, γιατί το ευρωπαϊκό μοντέλο έγινε ένα εξαγωγικό προϊόν όσον αφορά τον πολιτισμό. Το αντέγραψαν οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ινδία, από το Μεξικό μέχρι τη Βραζιλία. Και γιατί, γιατί δεν αποκλεί την ιδιωτική επιχείρηση, κάθε άλλο. Σέβεται απόλυτα επίσης το copyright, αλλά πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο οδηγεί σε, αλλαγή, σε αλλαγές από μέσα από τον κλάδο. Και αυτό είναι το σημαντικό γιατί επενδύει στην αλλαγή. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον. Μιλάμε εδώ για τα οικονομικά εφέλη. Αν δούμε τα νούμερα, και υπάρχουν πάρα πολλά που ακούστηκαν εδώ, εγώ θα καταλήξω σε ένα πολύ σύντομο συμπέρασμα ότι δαπανούμε πολύ λιγότερο από το 1% του ΕΠ μας στην Ευρώπη, στον κλάδο του πολιτισμού, ο οποίος συνεισφέρει όμως με 4,5% στο ευρωπαϊκό ΕΠ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή αυτή η μαθηματική πράξη, ότι δηλαδή η απόσβεση είναι τεράστια. Συνεπώς η έκκλησή μου είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στον κλάδο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που βασίζεται σε αξίες. Γιατί το χρυσορυχείο του πολιτισμού δεν είναι μόνο απόσβεση μέσα από τον τουρισμό κλπ αλλά βοηθάει την ταυτότητα, την ευημερία και την αλλαγή συμπεριφοράς και νοτροπίας. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανθίσει μόνο μέσα σε ένα περιβάλλον με συμμετοχή όλων και χωρίς δηλαδή αποκλεισμού. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη πλευρά. Αν δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, ξέρουμε ότι οι ριζοσπαστικές τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη αναδύονται όλο και περισσότερο. Οπότε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστική μας πρωτοκαθεδρία στην πολιτιστική κληρονομιά, πρέπει να αναλάβουμε υποχρέωση για επενδύσεις, για να μην γίνουμε η απικία της Silicon Valley. Ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια σας. Και δίνω το λόγο στον κύριο Σέμον Λίτλ. Είστε πρόεδρος της Interactive Software Federation of Europe. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Αντέλη. Τα βιντεοπαιχνίδια πρόσφατα προσθέθηκαν ε, στην πολιτιστική μας κληρονομιά και ήδη επηρεάζουν ε, τους πιο καθιερωμένους ε, καλλιτεχνικούς τομείς. Μπορεί να μην γνωρίζετε ότι έχει πολλά εκατομμύρια ανθρώπου που παίζουν βιντεοπαιχνίδια η Ευρώπη. Είναι κομμάτι του πολιτισμού μα. Δεν θα σα κάνει έκπληξη, αλλά σχεδόν το 50% τη Ευρώπη παίζει παιχνίδια τακτικά με τα παιδιά του για ψυχαγωγία, για εκπαιδευτικού λόγου, για να χαλαρώσει ή στο πλαίσιο κάποια θεραπεία. Ε, η σύνθεση ενό βίντεο παιχνιδιού βιντεοπαιχνιδιου πολύπλοκο. Έχει το λογισμικό που γράφεται από πολύ δημιουργικούς ανθρώπους ε, με υψηλές δεξιότητες. Αυτό ε, ε, καθορίζει την αλληλεπίδραση, αλλά ένα βιντεοπαιχνίδι περιλαμβάνει στοιχεία οπτικά, ηχητικά και μερικές φορές περίπλοκη αφήγηση. Και έχει πνευματικά δικαιώματα τα οποία καλύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία. Η τεχνολογία και το χαλιτεχνικό κομμάτι δημιουργούν αυτή την αλληλεπιδραστική εμπειρία. Τα βιντεοπαιχνίδια συνδυάζουν ε, σε άλλο επίπεδο τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Ε, ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά μέσα, χρησιμοποιούνται ως εκπαίδευση για την πολιτική μας κληρονομιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό στη, για τη σημερινή διάσκεψη. Το παράδειγμα είναι ένα παιχνίδι που ονομάζεται 1111 Memories Retold. Προγραμματίστηκε από μια γαλλική εταιρεία, την Digix Art το στούντιο Artman Animation στο Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιεύτηκε από την ε, Bandai Namco. Το 11 είναι ένα παιχνίδι τόσο καλλιτεχνικό που σχεδόν μοιάζει να είναι ένα αλληλεπιδραστικό ε, έργο ε, τέχνης. Λαμβάνει χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και περιγράφει τις εμπειρίες στα χαρακόμματα. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού συνεργάστηκαν με τις συλλογές του Ευρωπαϊκού. και η αγάπη ε, στο παιχνίδι και η έκφραση μέσω του παιχνιδιού ε, εκφράζει την ε, ανθρώπινη μας φύση. κάτι, το παιχνίδι δεν πρέπει να σταματά στην παιδική ηλικία. δεν υπάρχει ηλικία για να αναπτύξει κανείς το σύμπαν των βιντεοπαιχνιδιών. Et Και τώρα ο πρόεδρος του Project Click, ο κύριος ε, Λουίτζι Φούσκο Ζηρά. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι συντονιστή αυτού του έργου του Horizon, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτό το πρόβλημα της ε, σχέσης ε, της πολιτικής μας κληρονομιάς και της τοπικής ανάπτυξης. Ποιε αναπτυξιακέ διαδικασίε μα ενδιαφέρουν αυτέ που σχετίζονται με το τουρισμό όσο το δυνατόν πιο πολυβιώσιμο, όσο το δυνατόν πιο πολιτισμικό. Μα ενδιαφέρουν οι αναπτυξιακέ διαδικασίε που σχετίζονται με τι δημιουργικέ και καινοτόμε διαδικασίε και δραστηριότητε. Μα ενδιαφέρουν όλε οι ταπικέ δραστηριότητε που βοηθούν στην ανάπτυξη, στην ε, βελτίωση τη ευημερία, τη καλή ζωή του πληθυσμών. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Μα ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά επίσης το πραγματικό σημερινό διακύβευμα το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως ποιο η συμβολή στον εξανθρωπισμό των πολεών μας. Αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 26 του νέου θεματολογίου για τις πόλεις στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό διακυβεύεται αυτή τη στιγμή, διότι οι πόλεις μας δυστυχώς είναι όλο και πιο απάνθρωπες και στις χώρες μας συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Το ζούμε καθημερινά. Πώς ελπίζουμε εμείς να υλοποιήσουμε αυτή τη συμβολή ενισχύοντας, αναγεννώντας ε, την συνδεδεμένη υποδομή στις κοινωνίες μας μέσω της παγίωσης, του εορτασμού, ε, της προβολής της μνήμης, της ανάμνησης χωρίς απλά να προβάλλουμε τον οικονομικό μας πλούτο, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αξία συμβολική, πολιτισμική, πνευματική, για να το πω διαφορετικά. Στο project Click έχουμε εντοπίσει τρία σημαντικά σημεία αναφορά στην κυκλική οικονομία που είναι μια οικονομία συνεργατική ε, μαζί με το μοντέλο της κυκλικής ε, πόλης ε, και με την πολιτιστική κληρονομιά αυτή καθεαυτή. Με ποια μέθοδο σκοπεύουμε να εργαστούμε με νέα μοντέλα χρηματοδότησης και διακυβέρνησης που θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι αμοιβαία ε, κυκλικής οικονομίας ωφελών στην οποία θα συμμετέχουν οι ιδιώτες ε, οι κρατικοί φορείς και οι τοπικές κοινότητες. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αναφέρουμε πολύ συχνά εδώ τις τοπικές ε, κοινότητες. Στην πραγματικότητα αυτές οι τοπικές κοινότητες φαίνεται να είναι όλο και πιο κατακρεματισμένες. Όλο και πιο ατομιστικές ε, με ολοένα αυξανόμενους εγωισμούς. Το βλέπουμε αυτό στον κατακαιρματισμό και των κομμάτων και των εργασιακών ενώσεων και αυτή την αδυναμία εμείς προσπαθούμε να την σταματήσουμε αλλά πολύ συχνά τα προσωπικά συμφέροντα υπερισχύουν του κοινού καλού, της πόλης, της κοινωνίας, του γενικού καλού και αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο κίνδυνο εγγενούς ε, κρίσης ε, η οποία θα ε, γεννηθεί από το εσωτερικό και είναι συνεπώς πολύ επικίνδυνη οδηγεί σε απώλεια της αίσθησης κατεύθυνσης μιας κοινωνίας. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να συνδέσουμε την έρευνα ε, του τι είναι απαραίτητο για τις τοπικές ε, κυβερνήσεις, για τις περιφερειακές κυβερνήσεις, ώστε να συμβάλλουμε μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς να αναγεννηθεί η ανάπτυξη. Αλλά θεωρούμε ότι είναι και σημαντικό να βοηθήσουμε να αναγεννηθεί η κοινωνική γνώση, η κοινωνική ευθύνη. Η κοινωνική ευθύνη, το civil responsibility είναι άλλο ένα σλόγγαν που θέλουμε σε αυτό το θεματολόγιο. Ελπίζουμε μέσα σε δύο χρόνια να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα των οφείλειων αυτών μέσω της συνεργασίας μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ και μπορείτε και πάλι να τους χειροκροτήσετε για την ποιότητα των παρουσιάσεων τους και για την τιμή που μας κάνουν. Ε, ε, βλέπουμε από διαφορετικές σκοπιές ο καθένας. Ακούσαμε από το Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο του Λούβρου, τα προγράμματα επιτόπου ε, στις ε, διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και τους καλλιτέχνες που έχουμε εδώ. Ποιο είναι το ουσιαστικό και κεντρική ιδέα. Χωρίς τον πολιτισμό δεν κάνουμε τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε τα συναισθήματα να ζουν, δεν μπορούμε να κάνουμε τις ελευθερίες να ζουν, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, ιδιαίτερα ε, την αξία της ελευθερίας που πάντα θα πρέπει να την υπερασπισόμαστε. Σας ευχαριστώ και να καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Sit down, please. Chair, uh, Petra. Αγαπητή Πέτρα, ε, κύριε Αναπληρωτή Γενική Διευθυντή, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, είναι μεγάλη χαρά για το θεσμικό μας όργανο να σας καλωσορίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φέτος συμπληρώνονται 8 αιώνες από την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα. Είναι από τα πιο παλιά πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου. Στα πλαίσια αυτά, το πανεπιστήμιο που διευθύνεται ε, θέλησε να απονείμει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το χρυσό του μετάλλιο. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της κοινή μας πολιτιστικής κληρονομιάς απορρέει από την γνώση που έχουν διαδώσει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των αιώνων. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίω. χωρίς την κληρονομιά αυτή, την ε, πνευματική που αφήνεται και εξακολουθείτε να δίνετε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή και προνόμιο αυτή που έχουμε ε, στα πλαίσια της ε, διάσκεψης υψηλού επίπεδου που είναι αφιερωμένη στο, στην πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο στον αξιότιμο κύριο Πρίτανη, τον Ρικάρτο Ριβέρο Ορτέγα, για την απονομή του βραβείου. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι εκπρόσωποι ε, των ε, ευρωπαϊκών λαών ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκπρόσωποι του πολιτισμού, φίλες και φίλοι. Έχω την τιμή να πονέμω το μετάλλιο του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για τη συμβολή του Κοινοβουλίου στην πρόοδο και την ειρήνη των λαών της Ευρώπης. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας ε, στην ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας, που το 1218 έλαβε το όνομα του Πανεπιστημίου. Ο Αλφόνσο Ένατος το ίδρυσε και για πρώτη φορά συγκάλεσε ένα κοινοβούλιο που αναγνώριζε το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τις αφορούν. Η δημοκρατία, όπως και το πανεπιστήμιο, είναι ε, μέρος της καλύτερης ευρωπαϊκής ε, παράδοσης. Το πανεπιστήμιό μας από την αρχή έχει διατρανώσει ε, αυτή την πεποίθηση και το έχει αποδείξει η εκπαιδευτική μας ε, ταξίδευαν σε όλη την Ήπειρο για να μορφωθούν και να μορφώσουν. Ήταν προάγγελος του σημερινού προγράμματος Εράσμους και εμείς δεχόμαστε τους περισσότερους φοιτητές από όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κράτη. Είναι κοινέ οι αξίες μας και αρχές μας, η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ε, της ελευθερίας ε, και αυτά πρεσβεύουν και καθηγητές και καθηγήτριες στη Σαλαμάνκα. Η Ευρώπη θα πρέπει με λογική, με σύνεση να προστατεύει την ακαιρεότητά της ε, με αποφάσεις εφάμιλες των προκλήσεων. Μπορεί να βοηθήσει η πολιτιστική κληρονομιά προς την κατεύθυνση αυτή. Θυμίζουμε πάντα ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σύνολο ιδεών, αλλά ταυτόχρονα, όπως και το Πανεπιστήμιο, είναι και πηγή συναισθημάτων, αισθημάτων που μας ενώνουν και μας ανοίγουν προς τον κόσμο η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν. Όταν το δικό μας πνεύμα θα μπορέσει να συγκινηθεί αναβιώνοντας αυτό που είμαστε ότι είμαστε ενωμένοι σε αλληλεγγύη και ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί ε, κάλλιστα την Ευρώπη και τις αξίες της. Γι' αυτό το μετάλλιο αυτό αναγνωρίζει τους άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για μια Ευρώπη πιο ενωμένη εδώ σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που προστατεύουν τις αρχές και τις αξίες κλειδιά για την πρόοδό μας στους ηγέτες, όπως εσείς Πρόεδρε, που μπορείτε να ε, προσανατολίζετε τους λαούς προς την ομόνια, την ειρήνη και την επικοινωνία. Σε όλους αυτούς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, που ενώνετε την Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε. Φτάσαμε στην τελευταία φάση αυτή τη πολύ σημαντική ημέρα. Η μέρα μέσα στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με πολίτε οργανισμού, γυναίκε και ανθρώπου από το χώρο του πολιτισμού από όλου του διαφορετικού τομεί, προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα δυνατό για την ταυτότητά μας, για τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό παρότι διαφοροποιημένος παραμένει ευρωπαϊκός πολιτισμός. Δίνω το λόγο στην Πέτρα Κάμερεβερτ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού για τον τελευταίο γύρο χαιρετισμών και στη συνέχεια θα σας χαιρετήσω για να κλείσουμε αυτή την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Ήθελα και εγώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Πανεπιστήμιου της Αλαμάνκα. εργάστηκαν σκληρά για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τη διάδοσή τους στους νέους έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Μετά από ένα τόσο πολύ ωραίο και πλούσιο απόγευμα έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της διάσκεψης για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εγώ δεν θα αρχίσω να λέω μεγάλα λόγια προσπαθώντας να συνοψίσω όλες τις ιδέες που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα. Ακούσαμε πολλά. Είχαμε 44 ε, εξέχοντες ομιλητές. Ε, είναι ρεκόρ αυτό, μιλάει από μόνο του. Αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι ότι έχει ενισχυθεί η πεποίθησή μου ότι η Ευρώπη μπορεί να μην είναι απλά ένα ρητορικό εγχείρημα να γεμίσει όλες αυτές τις ιδέες με ζωή. Καθώς ε, κοιτάμε την πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις ανοιχτά για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Είμαι πεπισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν θα διαρκέσει μόνο τους επόμενους μήνες, θα επεκταθεί και πέραν του 2018 και θα αποτελέσει έναν φάρο που θα ευαισθητοποιεί τον κόσμο για, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πολυμορφία του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει. Εμείς ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ε, το Νοέμβριο θα κάνουμε μια ε, συνεδρίαση με τα μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων από όλα τα κράτη-μέλη όπου θα εστιαστούμε στη συμβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς ε, στο σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και στη δυνατότητα βιώσιμης διατήρησης των αποτελεσμάτων αυτού του έτους της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς μέσα στα επόμενα χρόνια. Πιο σημαντικό από όλες από αυτές τις πολιτιστικές ε, πρωτοβουλίες είναι η δέσμευση ενώσεων, οργανισμών και ανθρώπων αφοσιωμένων στην πολιτιστική κληρονομιά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας. Θεωρώ ότι η διάσκεψη μας σήμερα υπήρξε εξαιρετική. Ευχαριστώ. no tenemos la interpretación en todas las lenguas, por eso intentamos de hablar en inglés. Δεν έχουμε τη διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, λέει ο πρόεδρος. Κάποιες έχουμε ισπανικά, ελληνικά, γερμανικά, σουηδικά. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Σνιζάνα Ζάμαντιτ Μάρκοβιτ, εκ μέρου του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ταγιάννη, κυρίε και κύριοι. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια σύντομη ιστορία. Η πρόεδρος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Κάμερβερτ, είπε πόσο σημαντικό είναι να δείχνουν ενδιαφέρον και να εμπλέκονται οι τοπικές κοινότητες και ατομικά ο καθένας. Θα σας μιλήσω λοιπόν για μια γειτονιά της Μασαλίας, την Βόρεια Συνοικία, που είναι μια εργατική συνοικία. Όπως ε, κι αλλού ο κόσμος και εκεί εργαζόταν στη βιομηχανία. Τώρα όμως δεν υπάρχουν πια βιομηχανίες εκεί και έτσι η Βόρεια Συνοικία πλήττεται από ψηλά επίπεδα ανεργία, εγκληματικότητα, ναρκωτικά και πολλά άλλα προβλήματα. Στι αρχέ του 2000, λοιπόν, σύλλογοι κατοίκων που ανησύχησαν βέβαια για την ασφαλειά τους και την ευημερία τους, αλλά και εκείνη των παιδιών τους, αποφάσισαν να ασχοληθούν και να τροποποιήσουν την γειτονιά τους και να δημιουργήσουν το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα, να δώσουν και πάλι περηφάνεια στον κόσμο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της κοινή ε, κληρονομιάς, του κοινού πλούτου. Όμω, το πρόβλημα ήταν ότι εκεί στη Βόρεια Συνοικία δεν υπήρχε μια τέτοια κληρονομιά πλούτο, τουλάχιστον όχι με την παραδοσιακή έννοια. Εξού και δημιουργήθηκαν οι αρχές της σύμβασης του Φάρο που είναι μια νέα σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπη, η οποία δημιούργησε ακριβώ αυτή την έννοια της κοινή κληρονομιά στο δημόσιο χώρο. Επαναπροσδιορίστηκε το νόημα της κληρονομιάς δεν υπήρχε λοιπόν με την παραδοσιακή έννοια αυτή η κληρονομιά. Οι κάτοικοι όμω ενθαρρύνθηκαν για να δημιουργήσουν μία. Οπότε χρησιμοποιήθηκε ο κόλπος και οι καταράκτες του Ιαγιαλατκάς που αυτοί αποτέλεσαν και τον κοινό πλούτο, την κοινή κληρονομιά, ε, στοιχείο ταυτότητας για τους ανθρώπους αυτούς που σιγά σιγά έκτασαν μια κοινότητα. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετείχε και στήριξε την τοπική δράση και δημιούργησε αυτή την αλλαγή που ήταν πολύ θετική και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά εξαιτία ακριβώ αυτού του πλούτου. Και το σχέδιο απογιώθηκε. Ο δήμαρχος της Μασαλίας ενέκρινε και στήριξε τις δράσεις αυτές. Επιχειρηματίες από τα δικιά τους την πλευρά διέθεσαν ιδιοκτησία τους στο δημόσιο. Δημιουργήθηκε το Τέλ που αποτέλεσε κέντρο και κόμβο φιλοξενίας από τον οποίο πνεύτηκαν πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες ανά την Ευρώπη. Για μένα λοιπόν αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια τέτοια προσέγγιση απέναντι στην κληρονομιά. Για μένα αυτή η δύναμη της αλλαγής είναι κάτι πολύ σημαντικό και σημαίνει θετική κοινωνική, πολιτική και οικονομική δράση, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνίτων, το άνοιγμα, η επένδυση στη δημοκρατία και αποτελεί και ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να κάνει ένα διεθνές νομικό κείμενο, μια σύμβαση δηλαδή, εφόσον υπάρχει συνεργασία και δράση σε επίπεδα τόσο εθνικό όσο περιφερειακό και τοπικό. Έτσι η κοινωνία, οι επιχειρηματίες και άλλοι μπορούν να συμμετέχουν και επίσης βοήθησε φυσικά και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, διότι προσφέρει μέσα για την προώθηση ε, διαχείρισης προγραμμάτων όπως είναι το ΦΑΡΟ και να μπορούν έτσι να φτιάξουν τα δικά τους τέτοια προγράμματα, διάφορες κοινότητες και συνοικίες ανά την Ευρώπη. Σήμερα η γειτονιά αυτή η βόρεια εξακολουθεί να έχει κάποια προβλήματα, όμως χάρη στην κληρονομιά, στον πλούτο αυτό, με κέντρο τον ίδιο τον κόσμο και με διαχείριση από τον ίδιο τον κόσμο, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να λύσει αυτά τα προβλήματα στο μέλλον. Έτσι λοιπόν ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά βοήθησαν όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Και τελευταίο ομιλητή, ο Λούκα Γιαγιέρ, πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Αγαπητέ πρόεδρε Ταγιάννη, Κυρία Πρόεδρε Κάμερα Βέρτε και αγαπητά μέλη του πάνελ, είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε να μιλήσω εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο πλούσιες ήταν οι σημερινές ε, παρουσίες ε, και παρουσιάσεις. Ευχαριστώ για όλες τις ομιλίες. Εγώ ως πρόεδρος ε, όταν εξελέγει τον Απρίλιο ανακοίνωσα τον πολιτισμό ως μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας μου, δίπλα στην βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρήνη. Πολύ καιρό πριν γίνει πολιτικό έργο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, από τους ιδρυτές ε, και τη συνθήκη της Ρώμης υπήρχε η Ευρώπη ως πολιτιστικός χώρος μέσω της ανταλλαγής ε, εμπόρων, κληρικών, πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών. Είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο που βασιζόταν σε κοινά σημεία αναφορά σε έναν πολιτισμό που ε, έθεσε τα θεμέλια για τη σημερινή Ευρώπη και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σήμερα από το Πανεπιστήμιο του Σαλαμάκα ε, απονέμει το βραβείο αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επίτευγμά του στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η η ιστορία σας των 800 ετών είναι ένα παράδειγμα αυτό της ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ακαδημαϊκής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ρόλο κλειδί που διαδραματίσατε ώστε το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς να γίνει πραγματικότητα παρά όλα τα εμπόδια. Και έτσι μπορώ να πω ότι οι προτεραιότητες με βρίσκουν σύμφωνες Σύμφωνο. Συγκεντρώσαμε σήμερα Ευρωπαίους πολίτες για να συζητήσουμε πώς η δημοκρατία και ο πολιτισμός μπορούν να αναπτυχθούν σε μια ψηφιοποιημένη Ευρώπη. Πώς ε, η ετήσια εκδήλωσή μας, ε, Γιώργη Ροπιόρσεϊ, αφιερώθηκε στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενθαρρύνοντας νέους Ευρωπαίους να εκφραστούν για το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το ετήσιο βραβείο μας ε, για την κοινωνία πολιτισμού των πολιτών που θα απονεμηθεί στα τέλη του έτους θα αφορά την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τις ευρωπαϊκές αξίες. Η ΕΟ και είναι ο τόπος όπου η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, των πολιτών θα έχει να εκφέρει άποψη για το νέο θεματολόγιο τον πολιτισμό. Επίσης, εκπονούμε μία έκθεση για την πολιτιστική κληρονομιά και το αγροτικό περιβάλλον. Γιατί Σε ένα πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την καινοτομία και την έρευνα και την πολιτιστική κληρονομιά παραβλέφθηκε μία πρόταση η οποία λέει ότι η διοικητική αναγνώριση του πολιτισμού εξαρτάται από τη διάρκεια εντολής ε, υψηλοβάθμων Ευρωπαίων πολιτικών. Υπάρχει μια τάση, συνεχίζω, να τονίζεται η σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού στο τέλος τέτοιων θητιών. Αυτό συμβαίνει τώρα Έχουμε γίνει πιο σοφοί ή δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Όχι. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι έχουμε φτάσει σε ένα σταυροδρόμι σημαντικό, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν μια βαθιά ανάγκη επανίδρυσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αυτό δίνει νόημα και δύναμη σε αυτή την έκκληση για δράση που υπέγραψα και εγώ την περασμένη Παρασκευή με πολλά άλλα μέλη του πάνελ λόγω της εξαιρετικής ε, πρωτοβουλίας Europa Nostra στο Βερολίνο. Όλοι μας θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει ο πολιτισμός για ένα νέο βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Αυτό θα αποτελέσει τη δική μας αναγέννηση. Ευχαριστούμε. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Λούκα πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής. Τελευταίος ο μιλητής είναι ο κ. Ξενικού, Γενικός Διευθυντής της UNESCO. Έχετε τον λόγο. Κύριε Αντώνιο Ταγιάννη, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πέτρα Κάμερφερτ, Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Λούκα Γιάρ, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αξιότιμοι υπουργοί, επίτροποι, ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Εξ μέρους του Γενικού Διευθυντή της UNESCO, του κ. Λουρίσας, ε, ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε στην ε, σημαντική αυτή διάσκεψη για τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατέστησε δυνατή την εκδήλωση αυτή, για τη συνεργασία σας επίσης για την UNESCO. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή έρχεται μια σημαντική στιγμή, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον κόσμο, δεδομένου ότι η Ευρώπη όλο και περισσότερο διαφοροποιείται. Είναι πολύ σημαντικό την διαφοροποίηση αυτή να την υπογραμμίσουμε σαν τη δύναμη της Ευρώπης, σαν τα θεμέλια για ανάπτυξη, καινοτομία και ευημερία. Η πολιτιστική πολυμορφία εξάλλου αποτελεί και την ρίζα της ανάπτυξης, όχι μόνο της οικονομικής, αλλά την ανάπτυξη των ανθρώπων ως ανθρώπινο είδος. Και γι' αυτό και οι πρόσφατες ετάσεις ξενοφοβίας, εθνικισμών και αποκλεισμών είναι κατερνητικό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται συνειδητοποίηση για τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις ε, αξίες που αυτή υποστηρίζει. Πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά. Αποτελούμε πάρα πολλά σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία που έχει καταγράψει και η UNESCO για την ανθρωπότητα που δείχνουν τον πλούτο των ζωντανών παραδόσεων. Είμαστε στο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί μια ευκαιρία για να δείξουμε ακριβώς ότι αυτή η κληρονομιά αποτελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ακρογωνίο λίθο του ευρωπαϊκού οράματος, κάτι το οποίο πρέπει να εμπνεύσει τη μελλοντική δημιουργία. Η UNESCO λοιπόν χαίρεται πάρα πολύ που μπορεί να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το συνδυασμό και την ανάπτυξη πολλών ε, σημαντικών πρωτοβουλειών για φέτος, μεταξύ άλλων ε, προγράμματα για τους νέους. Κάτι το οποίο περιλαμβάνει την ε, πολιτιστική κληρονομιά στα σχολεία. Πρέπει να προστατεύσει η Ευρώπη τον πολύτιμο αυτό πλούτο, της παραδόσεις. Οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι προσθέτουν νέα στοιχεία στην, ε, στις παραδόσεις μας και στην κληρονομιά μας. Το Νοέμβριο, να ξέρετε ότι η UNESCO θα οργανώσει ένα φόρουμ για τους νέους στην Κροατία με την ευγενή στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατικών αρχών. Είμαι ευγνώμων προς τον Επίτροπο Λευράσκης και τους συνεργάτες του και το Γενικό Γραμματέα για την στήριξή τους και τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αντικατοπτρίζει την δέσμευση τόσο της UNESCO όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στους νέους για να συμμετέχουν και να προωθούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού αυτού έτους η UNESCO χαίρεται που μπορεί να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει το πρώτο σύνταξη ιδιώνο στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγγράφεται στο σχέδιο για τις πολιτιστικές ευρωπαϊκές διαδρομές, κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2016. Με στήριξη από το National Geographic, αυτή η νέα πλατφόρμα θα καταδείξει ότι οι διάφορες τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης μοιράζονται ένα κοινό πολιτισμό και θα οδηγήσει τους τουρίστες να πάνε σε λιγότερο γνωστά μέρη με μικρότερη επισκεψιμότητα και να ανταλλάξουν απόψεις για την κοινή τους κληρονομιά. Θα επιτρέψει επίσης και ανευπροηγουμένου συνεργασία μεταξύ αυτών που διαχειρίζονται το site ε, αυτό όπου συμμετέχουν 19 χώρε Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα η UNESCO θα είναι στο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και επιθυμεί η συνεργασία αυτή να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επαγγελματίες τη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιάς, ε, τα σχολεία, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και επαγγελματίε θα συνεργαστούν μαζί μας. Το πρόγραμμα αυτό εκφράζει επίσης και την πεποίθηση της UNESCO. Κάθε πρωτοβουλία διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα εργαλεία και τα ψηφιακά εργαλεία προφανώς τα οποία πρέπει να στηρίξουν τι στρατηγικέ μας γύρω από τον πολιτισμό. Τέτο αυτό το 2018 πρέπει να στεφθεί από καινοτομία. Πρέπει να προστατεύσουμε την κληρονομιά μας να παραμείνει ζωντανή και μόνο αν μείνει ζωντανή μπορούμε και να την προστατεύσουμε πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε σε θέση να υποδεχτούμε τη δημιουργία. Η ιδέα αυτή λοιπόν μια ζωντανή κληρονομιά, η οποία φέρει το όραμά μα προς το μέλλον είναι αυτή πολλών ευρωπαϊκών ε, χωρών όταν πριν από πάνω από 70 χρόνια είχαν σκεφτεί το 1% για την δημιουργία και αυτό θέλησα να περάσω στις επόμενες γενιές. Και θα τελειώσω με ένα τελευταίο νούμερο. Κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια άνθρωποι περνούν τα σύνορα της χώρας τους για να ταξιδέψουν, για ψυχαγωγία. Το νούμερο αυτό πρέπει να γίνει 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Με αυτήν ε, την ε, καταπληκτική πολιτιστική κληρονομιά, η Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδεύουν, αυτή την επιθυμία της ανακάλυψης νέων εμπειριών. Η κληρονομιά αποτελεί και τον πλούτο της Ευρώπης, αλλά και το μέλλον της. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κούκια για τη δεσμευσή σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της ημέρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση, όλους τους προσκεκλημένους, όλες τις προσωπικότητες, ε, ε, τις πολύ σημαντικές που ήρθαν εδώ από το χώρο του πολιτισμού. Ευχαριστώ τους βουλευτές και όλους όσοι αποφάσισαν να πρωταγωνιστήσουν, να συμμετέχουν ε, στα πάνελ αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας ημερίδας για όλους μας. Έχουμε, πιστεύω, στείλει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όλη την Ευρώπη, υπερασπιζόμενη την πολιτιστική ταυτότητα στην πολυμορφία της, ε, στην Ένωσή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρώτα απ' όλα την Μαγδαλένα Πιόρουν. Ε, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για αυτή την ημερίδα, για αυτό την πολύ σημαντική εκδήλωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της DigiLink, DigiCom, DigiEpol, την Ευρωπαϊκή Καλτ και Τράνα για αυτή την εκδήλωση και τους διερμηνείς για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Όλοι μαζί υπερασπιζόμενοι τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Αυτή είναι η στρατηγική μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να κάνουμε όλο και περισσότερε τέτοιε συναντήσει. Χρειαζόμαστε και τη δική σα συμμετοχή. Ευχαριστούμε.